Mesdames, Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το σχέδιο μερίσιας διάταξης μπορεί να εγκριθεί, εάν δεν έχετε αντιρρήσεις. Πες μας, Δομινίκ, ποιο είναι το πρόβλημα. Κυρία Πρόεδρε, δεν συμφωνώ με τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, διότι με ονομάζει κυρία Πρόεδρε, ενώ προείδρευα εγώ. Μάλιστα λαμβάνουμε υπόψη το σχόλιο σας, κυρία μου. Δεν ξέρω, αυτό σημαίνει ότι θα προαχθείτε. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε την διόρθωση. Δεν θέλετε να σας λέμε κυρία Πρόεδρε, εντάξει, δεν πρόκειται. Συνεχίζουμε τα πρακτικά τώρα της 1ης Φεβρουαρίου 2018 μπορούν να εγκριθούν αν δεν, έχουν, δεν υπάρχει αντίρρηση. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου δεν υπάρχουν, οπότε θα αρχίσουμε ευθύ αμέσω με την ανταλλαγή απόψε με τους Ευρωπαίους Δανειστές ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής των κανονισμών διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και με την προπαρασκευή της περίοδου πέραν του 2020, ε, η οποία είναι αυτή τη στιγμή εν εξελίξη, θα ήταν καλό να δούμε λίγο όλους τους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου, που είναι η ραχοκοκαλιά των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Οι Ευρωπαίοι συντονιστές έχουν οριστεί ακριβώς για να διευκολύνουν την συντονισμένη ανάπτυξη του κεντρικού δικτύου και βεβαίως αυτοί είναι που μπορούν να μας ενημερώσουν πιο υπεύθυνα για τις τελευταίες εξελίξεις και τις μελλοντικές, τα μελλοντικά στάδια πριν τελειώσει η θητεία τους. Ε, το στόχο σήμερα είναι να ακούσουμε, να συζητήσουμε, να δούμε τι, ποια πρόοδος έχει σημειωθεί, ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε στους εννέα ε, διαδρόμους ε, και βεβαίως η οριζόντια προτεραιότητα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών με τις θαλάσσιες αρτηρίες, με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Πολλά έχουμε να μάθουμε και για την υλοποίηση αυτών των διαδρόμων αλλά και τα οριζόντια ζητήματα όπως ε, η απανθρακοποίηση, τα ζητήματα ψηφιοποίηση τα ζητήματα χρηματοδότησης και βεβαίως οι δυτέ διτές μεταφορές τι πρέπει να γίνει επίσης για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα Τη ολοκληρωση του δικτύου εν ώψη μάλιστα και τη προπαρασκευής του μελλοντικού δημοσιονομικού πλαισίου. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω, να καλωσορίσουμε όλοι μαζί τους ε, συντονιστές, τους Ευρωπαίους συντονιστές ε, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Θα, δεν χρειάζεται να σας παρουσιάσω. Ο κύριος Γκρός είναι εδώ δίπλα μου. Είναι ο συντονιστής ε, ε, του διαδρόμου Ισμέτ, ε, του Ανατολικού, ο κύριος Έση ε, είναι ο συντονιστής του διαδρόμου του Ατλαντικού και η Καθρίνη Τροτμάν, την οποία γνωρίζουμε όλοι, συντονίστρια του διαδρόμου της Βαλτικής, ο κύριος Μποντεουίν, Βαλτική-Αδριατική, αυτός, ο διάδρομος δηλαδή, ο κύριος Μπάλας, συντονιστής ε, Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειο, ο κύριος Σίμψον. Πώς είστε κύριε Σίμψον. Πολύ καλά, πολύ ωραία. Είστε ο συντονιστής ε, για τις ε, θαλάσσιες αρτηρίες. Είστε και ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, έτσι. Καλό είναι να μιλάμε για τους προκατόχους μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Η κυρία Κάρλα Πέζ, ακριβώς δίπλα, η συντονίστρια ε, Ρίνος Δούναβης, ε, του, του, του διαδρόμου ρίνο Δούναβη, ο κύριος Πιέτνικ είναι ο συντονιστής της, ε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΜΕΣ και ο κύριος Βοητσόφσκι, Βοητσιτσόφσκι, συγγνώμη, για τις Άλπεις και το σχετικό διάδρομο. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ για αυτό τον, την ανταλλαγή απόψεων που είναι κεφαλαιόδης σημασία για μας. Ο, Πάλε, ο Πάβελ, τον Πάβελ Βοητσιτσόφσκι το βλέπω σχεδόν κάθε εβδομάδα. Για άλλα θέματα όμως. Ε, οι συντονιστές ε, τώρα του διαδρόμου ε, Σκανδιναβίας Μεσογείου, κύριος Κόξ ε, δεν είναι εδώ μαζί μας αλλά θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Μπάλλας αλλά και από τον κύριο Βοητσιτσόφσκι. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ σήμερα. Ε, η ανταλλαγή απόψεων θα λάβει χώρα σε δύο μέρη. Θα έχουμε ένα πάνελ Ευρωπαίων συντονιστών κάθε φορά με τους εκπροσώπους των διαφόρων ε, διαδρόμων αλλά και με κάποια θεματικά, θεματικές ενότητες. Κάθε παρέμβαση, μετά από ένα γύρο πανεμβάσεων των ομιλητών θα έχουμε και ανταλλαγή απόψεων με τους ε, παρευρισκόμενους. Καλό να μας κάνετε μια σύντομη παρουσίαση βεβαίως του φακέλου σας. Πέντε λεπτά θα έχει ο καθένας, είναι δύσκολο το ξέρω. Ε, σας παρακαλώ να σεβαστείτε τον χρόνο ομιλίας για να μπορέσουμε πραγματικά να προλάβουμε να έχουμε και διάλογο. Ξεκινάει λοιπόν η συζήτηση. Θα μιλήσουμε πρώτα για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών δικτύων των υποδομών μεταφορών. Ο κύριος Σέισι και ο κύριος Μπόντεβιν Έχετε πέντε λεπτά μαζί. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Σε αυτή την πρώτη παρέμβαση από τον κύριο Μπόντεβικ, λέει ο κύριος θα σας παρουσιάσουμε την έκθεση προόδου για τη λεγόμενη έκθεση CBS που προετοιμάσαμε πριν από δύο χρόνια κατόπιν ετήματος... το Σεπτέμβριο του 2015 του, της άτυπης Υπουργικής Συνόδου Μεταφορών ε, στο Μιλάνο. Είναι στην διάθεση όλων αυτή η έκθεση η οποία είναι δομημένη όπως και η προηγούμενη, ακριβώς όπως η προηγούμενη, 12 συστάσεις. Αυτό θα διευκολύνει την ανάγνωση και θα είναι και καλύτερο, θα είναι και πιο εύκολο μάλλον να δούμε ε, την πρόοδο που έχει σημειωθεί ε, τα τελευταία δύο χρόνια. Εμείς θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πώς μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη συμμετοχή ε, κεφαλαίων ιδιωτικών, μη δημοσίων, εν περιπτώσει, διότι οι δημόσιοι πόροι είναι όλο και πιο περιορισμένοι, οι ανάγκες ταυτόχρονα αυξάνονται, και αντιμετωπίζουμε μια σειρά από εμπόδια που δεν επιτρέπουν αυτή τη συμμετοχή. Το πλαίσιο δηλαδή αυτή τη στιγμή η συγκυρία δεν είναι πολύ καλή για την χρηματοδότηση, την υποστήριξη την οικονομική από ιδιώτε. Και σκεφτήκαμε λοιπόν ότι καλό θα ήταν να δούμε τι έχει συμβεί στον τομέα αυτό. Έχουν γίνει αρκετά και βεβαίω τι μένει να γίνει. Ποια ζητήματα δεν έχουν επιληθεί και ποια νέα προβλήματα έχουν εμφανιστεί. Εμείς έχουμε προετοιμάσει την έκθεση πρόοδου. Εδώ έχουμε μοιράσει τη δουλειά με τον κύριο Μπόντεβιγκ σε ό,τι αφορά το τι έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Πολλές από τις συστάσεις μας ελήφθησαν υπόψη και χαιρόμαστε γι' αυτό. Επίσης πολλά μέτρα ε, σίγουρα ακολουθούν το σωστό δρόμο. Παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μια ενιαία θηρίδα για σημαντικά ευρωπαϊκά project και ένα σύστημα τεχνικής συνδρομής μέσω του Jaspers αλλά και μέσω ε, του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Hub Ταυτόχρονα οι κανόνες περικρατικών ενισχύσεων αναθεωρούνται για να είναι πιο απλοί αλλά και πιο προβλέψιμοι από την αρχή της διαδικασίας. Η τροποποίηση της οδηγίας για τις εξαιρέσεις έχει οδηγήσει στο να μπορούμε να έχουμε περισσότερα project. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ένα, ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα έχει να κάνει με τις χρηματαγορές έχουμε επανεξετάσει τις εργαλείες, ε, τα εργαλεία συγγνώμη, ε, αφαιρεγγιότητας ε, για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, μακροπρόθεσμη οικονομική στηρίξη από τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς παράγοντες. Οι προσπάθειές μας ε, για ένα σαφέστερο πλαίσιο στον αφορά τις συμπράξει δημοσίου ιδιωτικού δικαίου έφεραν αποτέλεσμα μιας και έχουμε τι νέε κρατικέ γραμμές στον τομέα αυτών σε ό,τι αφορά την, οικονομική, καινοτομία έχουμε κάποια πρώτα στοιχεία ε, για να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες δανεισμού στον τομέα των μεταφορών και για να αναθεωρηθεί η οδηγία ΣΕΦ, να, μάλλον να προχωρήσει η αυτορύθμιση, συγγνώμη. Ε, βεβαίως ε, είναι μακρύς ο δρόμος. Πάμε προς αυτή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε χρηματοδότηση και επενδύσει στον τομέα των μεταφορών και στις σχετικές υποδομές και εκεί επικεντρώνεται η έκθεσή μας. Εμείς κυρίως θέλουμε να ενισχύσουμε την ποιότητα ε, των ε, project μας. Αυτό θα είναι το σημείο κλειδί για να στεφθεί από επιτυχία η προσπάθειά μας και να συμμετάσχουν οι ιδιώτε ε, σε αυτά τα project υποδομών. Έχουμε περίπου 3.000 project, ε, τεράστιες οικονομικές ανάγκες, περίπου 500 δισεκατομμύρια από το 2021 έως το 2030 ε, μόνο και μόνο για αυτό το δίκτυο πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες για να ληφθούν υπόψη και πιο μικρά project τα οποία ε, δεν μπορούν να προχωρήσουν λόγω του υψηλού διοικητικού άχθους. Θα πρέπει επίσης να διευρύνουμε τις πηγές χρηματοδότησης να βρεθούν περαιτέρω οικονομικοί πόροι μέσω παραδείγματο χάρη ε, της εφαρμογής της αρχής του ορυπαίνων πληρώνει και ο χρήστης πληρώνει ε, και μια αναθεώρηση της ε, οδηγίας ευρωβινιέτα. Θα πρέπει επίσης να έχουμε πιο ε, ε, προχωρημένες αναλύσεις σε ό,τι αφορά τα δια... τη των project. Μπορούν επίσης να αναζητηθούν και άλλες πηγές. Θα μπορούσαμε να ξαναδούμε το σύστημα ε, εμπορίας ε, ρήπων, Επίσης όταν θα εγκριθούν οι απλοποιημένες οικονομικές, οι οικονομικοί κανονισμοί μπορεί να ε, βελτιώσουν την πρόσβαση των κρατών μελών σε αυτά τα ευρωπαϊκά μέσα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπόντεβικ για να συμπληρώσει αυτή την παρουσίαση. Dear Chairwoman, Αγαπητή Πρόεδρε, κυρία Ντέλη, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα ο καθηγητής Σέκη ήδη σας ε, έδωσε μια εικόνα της έκθεσης πρόοδου μας και ε, ανέφερε και μια σειρά συστάσεις. Θα ήθελα τώρα να σταθώ σε δύο από τις ε, συστάσεις μας που θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικέ. Έχουν να κάνουν με την απλούστευση των διαδικασιών, δημοσίων προμηθειών και αδιοδότησης. Στο δικό μου διάδρομο Έχουμε συγκεκριμένα στρατηγικά σημεία, ε, κυρίως έχουν να κάνουν ε, με την διασύνδεση με την ε, Τσεχία. Είναι μια σημαντική στενοπόσο που παρεμποδίζει την ομαλή εμπορική δραστηριότητα Υπάρχει συγχρηματοδότηση εν μέρη από το ΣΕΦ, από την αυστριακή πλευρά. Από την ε, τσεχική πλευρά όμως, εδώ και χρόνια προσπαθούμε να οριστικοποιηθεί μια τελική εξολόγηση και να υπάρξει τελική αδειοδότηση του έργου. Ως ε, Ευρωπαίοι συντονιστέ έχουμε κάνει πολλέ προσπάθειε για να βρούμε λύσει, όμω παραμένουν καθυστερήσει και ένα από του βασικού ε, κανόνε είναι ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού σε ό,τι αφορά του αδιούχου για την τελική χρήση και στις δύο χώρες. Ε, αυτό είναι μια τυπική κατάσταση για πολλά τα διασυνοριακά μας έργα, και τα μικρά και τα μεγάλα διασυνοριακά, όπως το Μπρεν και το Ρέιν Βαλτική. Ε, για... Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στην εξομάλυνση αυτών των εμποδίων για να επιτύχουμε και να εφαρμόσουμε ε, με επιτυχία τις πολιτικές μας για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Είναι θετικό λοιπόν που η Επιτροπή και η σχετική αρμόδια Γενική Διεύθυνση έκανε μία μελέτη ε, που σε ό,τι έχει να κάνει με την αδειοδότηση και χαιρόμαστε που στο τρίτο πακέτο κινητικότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια πρόταση για ένα ευρωπαϊκό κανονισμό απλούστευση των μέτρων για την ταχύτατη εφαρμογή ε, των ε, πολιτικών για τα δίκτυα ΔΕΔΜΗ. Μία ιδέα που προέκυψε από την μελέτη και την οποία στηρίζουμε είναι η θέσπιση ενός ενιαίου αντιδοτικού μηχανισμού για τα προγράμματα TNT. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δραματίσει πιο άμεσο ρόλο στην διαδικασία αναθεώρηση προγραμμάτων ε, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα επιλεγμένα προγράμματα TNT, τουλάχιστον για τι ε, άδειε που προκύπτουν και απορρέουν άμεσα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να θεσπιστούν εθνικέ ε, αρμόδιε αρχέ, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενιαία θηρίδα για του ενδιαφερόμενους και θα είχαν την αρμοδιότητα έκδοση αδειών. Και στι δύο περιπτώσει πρέπει να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση προκειμένου να περιοριστεί ο χρόνος ε, αδειοδότησης. Εμείς προβλέπουμε διαδικασία που αφορούν την, τον περιορισμό ή μάλλον ότι σε καμία περίπτωση πρέπει να πέσει το επίπεδο των, ε, των απαιτήσεων και προποθέσεων. Είναι σημαντικό να το επισημάνουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά το, το τώρα του ζητήματο, εκεί θα πρέπει να καταβάλουμε τι μεγαλύτερε δυνατέ προσπάθειε για την απλούστευση των εθνικών ε, δραστηριοτήτων και διαδικασιών. Και αυτό μπορεί να μας ε, βοηθήσει να περιορίσουμε το ε, χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση. Όλα αυτά σας τα είπα για να σας δώσω μια πρώτη εικόνα των όσων προτείνουμε στην έκθεση πρόοδου μας. Τώρα θα ήθελα να κλείσω με την εξή δήλωση. Ως Ευρωπαίοι Συντονιστές έχουμε εργαστεί σκληρά τα τελευταία χρόνια για την ανάλυση και σύσταση ε, μιας σωστής και σταθερής διαδικασίας για την υλοποίηση των έργων TNT. Είναι πολύ υψηλέ επενδυτικέ ε, ανάγκε και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και ένα εύρωστο επενδυτικό σχέδιο. Θα πρέπει να συνίσταται σε τρία τμήματα οι επιδοτήσεις θα πρέπει να ε, αφιερώνονται μόνο σε αυτά έργα που έχουν την μεγαλύτερη δυνατή ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία, τα διασυνοριακά και αυτά που ε, έρουν σημαντικές στενοπούς. Τέτοια έργα ε, θα πρέπει να λαμβάνουν επιδότηση σημαντική από το ΣΕΦ. Δεύτερον, χρειαζόμαστε καλό σχεδιασμό των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών οργάνων και μηχανισμών Αυτά λοιπόν να πρέπει ε, να βοηθούν ε, τα σοβαρά σχέδια για έργα που μπορούν να περπατήσουν και έχουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Τρίτον, κάποια από τα έργα TNT θα μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με ένα μείγμα ε, χρηματοδότησης και πιστώσεων, το λεγόμενο blending ιδίως στα έργα τα οποία βρισκόνται σε μεταβατική φάση ε, ισχύει αυτό. Τα έργα δηλαδή που δεν εξαρτώνται πλήρως από τις επιδοτήσεις, ούτε είναι και αυτάρκη όμως. Και είχαμε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου υπήρχε πολύ σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον ε, και ήταν σημαντικό το γεγονός ότι υπήρξε επιδότηση εκεί και θα πρέπει αυτό να αποτελέσει ένα από τα μόνιμα εργαλεία για το μέλλον. Κλείνοντα, αυτό, αυτή η ισορροπημένη ανάμειξη των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων είναι ο μοναδικός ε, τρόπος να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Αυτό εμείς ε, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τις παρεμβάσει σας. Χωρίς να χάνουμε χρόνο, δίνουμε απευθεία το λόγο στον κύριο Κρό. Παρακαλώ. Για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λίγο για το πού βρισκόμαστε στους διάφορους διαδρόμους και βεβαίως ιδιαίτερα για το δικό μου. Είμαστε στη φάση του τρίτου ε, προγράμματος δράσης, τρίτη γενιά. Για όλους τους διαδρόμους θα βρείτε εδώ ένα κατάλογο των project που έχουν ξεκινήσει και αυτών που θα ε, ολοκληρωθούν στο μέλλον, ε, στο 2020-2021, έτσι, όχι ως το 2030. Σε αυτό το πρόγραμμα εργασιών ε, μπορείτε να δείτε πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τα διάφορα κριτήρια αποδοτικότητας ανά ε, διάδρομο ε, το, το οποίο εξετάζουμε συχνά, διότι η προσθέμενη αξία του διαδρόμου είναι αυτή η διασυνοριακή θεώρηση, αλλά και το γεγονό ότι έχουμε κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια τα οποία αποδεχόμαστε όλοι. Είναι μια σημαντική πτυχή αυτή. Και ένας τρίτος, μια τρίτη πτυχή που είναι σημαντική είναι ε, να μην μιλάμε μόνο για χρήματα, να μιλάμε και για οικονομικές επενδύσεις, επενδύσεις ε, για το περιβάλλον και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Πρόκειται για πτυχές ε, εξαιρετικά σημαντικές για την περίοδο 2020-2030. Ελπίζουμε να φτάσουμε στα, στα 13, 13, 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ναι, σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου. Οι πτυχέ που έχουν να κάνουν το περιβάλλον θα, θα αναφερθούν και από άλλους συναδέλφου σίγουρα. Εάν δούμε τώρα πιο συγκεκριμένα τον Orient East Med που ξεκινάει στο Αμβούργο και κατεβαίνει μέχρι την Αθήνα περιλαμβάνει και την Κύπρο εδώ έχουμε 415 projects σε 9 διαφορετικές χώρες ε, υπάρχουν πολλοί, ε, δίκ, πολύ διάδρομοι περνάνε από τις, από τις χώρες. Δεν είναι πάντα μεγάλα τα project αυτά βέβαια. Ξέρω ότι ενδιαφέρονται πολλοί συνάδελφοι. 82% των project ε, αφορούν ποσά από 1 έως 500 εκατομμύρια. Ε, δεν είναι δηλαδή τα πολύ μεγάλα project. Είναι και μια διαφοροποιημένη προσέγγιση αν θέλετε. Βεβαίως προσθέμενη αξία με τέσσερα από αυτά τα project είναι διασυνοριακά και 40% αφορούν το σιδηρόδρομο. Θα επανέλθω από αυτού. Αυτό σημαίνει ότι σε ό,τι αφορά το Orient East Med, σε ό,τι αφορά την άμεση χρηματοδότηση, ε, έχουμε ως τώρα 92% ε, ε, των διαθέσιμων μέσων που έχουν απορροφηθεί. Αυτό σημαίνει 2 δις για τον ε, συγκεκριμένο ε, διάδρομο ανατολικό και ανατολική Μεσογείου. Εδώ βλέπετε τι γίνεται με το σιδηρόδρομο, παραδείγματος χάρη, το σιδηροδρομικό δίκτυο. Το πράσινο σκέλος ε, είναι αυτό που συμμορφώνεται με τα κριτήρια αποδοτικότητας, Το υπόλοιπα δεν συμμορφώνονται ακόμα. Το ίδιο θα το βρείτε και για τις εσωτερικούς εσωτερικέ θαλάσσιε οδού. έχουν φτάσει μια συμφωνία σε αφορά τον Έλβα συζητήθηκε αυτό στην ε, Γερμανία και με την Τσεχία δηλαδή θέλουμε μπορούμε να πετύχουμε ένα στόχο να διατηρηθεί εδώ η εσωτερική αλλά λαμβάνοντας υπόψη να βεβαίω ότι τα 2,5 μέτρα που είναι το κριτήριο απόδοση ε, δεν είναι απαραίτητο να γίνουν σεβαστά όπως και στην προσέγγιση, στην προσέγγιση μας ως συντονιστές μπαίνουμε και σε διάλογο δηλαδή για να γίνουν πιο ελαστικά κάποια κριτήρια. Ό,τι αφορά τις επενδύσεις τώρα σε όλες τις εκθέσεις και στα σχέδια που θα σας υποβληθούν θα βρείτε ένα χάρτη όπου θα περιλαμβάνονται οι επενδύσεις που γίνουν οι επενδύσεις αυτές και ποιο είναι το ύψος τους. Οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο ε, σε ό,τι αφορά τους διαδρόμους, ε, διότι όπως είπα και στην εισαγωγή μου, δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση αυτό που μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει και ο αντίκτυπος ε, στο ΑΕΠ, παραδείγματο χάρη. Εμείς θέλουμε να υπάρξει μια αύξηση των της τάξης των 517 δισεκατομμυρίων έως το 2030. Θέλουμε να έχουμε και δημιουργία θέσεων Είναι σημαντικά επιπλέον στοιχεία. Ως συντονιστής, ε, ως συντονιστές ενδιαφερόμαστε και για πτυχές που δεν σχετίζονται με τη χρηματοδότηση. Εγώ ενδιαφέρθηκα ιδιαίτερα στη διασυνοριακή πτυχή. Έχουμε λοιπόν κάνει μια ανάλυση όλων των διασυνοριακών προβλημάτων που δεν συνδέονται με τη χρηματοδότηση αλλά που συνδέονται με την τεχνική. Η διαλειτουργικότητα, παραδείγματο χάρη αφενό, ε, πτυχέ ε, ε, επιχειρησιακέ ή αναπτυξιακέ, σε ό,τι αφορά την τεχνική ανάπτυξη τουλάχιστον. Για κάθε διασυνοριακό σημείο υπάρχει ένα σχήμα όπου αναφέρονται τα διάφορα προβλήματα. Ε, ε, έχουμε περίπου 10 ώρες ε, καθυστέρηση στο σύνολο του διαδρόμου για διοικητικού λόγους στα διάφορα σύνορα. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση είναι σημαντική γιατί τώρα να έχουμε ένα νέο ΣΕΦ αφενός ε, έχουμε σχέδια 40 δις αυτή τη στιγμή που είναι ανεξελίξη δεύτερον η διασυνοριακή προσέγγιση παραμένει σημαντική Τρίτον, θα πρέπει στο μέλλον λίγο περισσότερο ακόμα να δούμε τη σχέση μεταξύ του κεντρικού δικτύου και του συνολικού δικτύου και βεβαίω ε, εφόσον 80% των πολιτών ζουν σε αυτά τα hub πρέπει να λάβουν πόσο σε και αυτά τα ε, hub nodes και κάποια project χωρίς άμεση χρηματοδότηση δεν μπορούν να προχωρήσουν και χωρίς ε, χρηματοδότηση σε συνοριακό επίπεδο θα το κάνουν αυτό οι χώρες μόνες τους. Ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό για το μέλλον όχι μόνο των μεταφορών αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και ε, την αντιμετώπιση των κλιματολογικών προβλημάτων. Ευχαριστώ τον κύριο Γκράους. Ο κύριος ε, Βίνκ έχει το λόγο για πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, και εγώ θα ε, πω δύο λόγια ως προς το που βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό το φημισμένο ε, πρόγραμμα ERTMS. Ε, κάποιοι ίσως να το έχουν ακούσει, αλλά λίγοι γνωρίζουν περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Ουσιαστικά, εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ο αριθμός των τρένων που είναι εξοπλισμένα με RTMS είναι 4.000 ε, ή μάλλον 40.000 χιλιόμετρα είναι εκείνα που καλύπτονται με αυτό το σύστημα ενώ θέλουμε να έχουμε φτάσει ε, στα 70.000 χιλιόμετρα έως το 2030. Ουσιαστικά ε, τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Έχουμε αντικαταστήσει 23 συστήματα διαφορετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα νέο σύστημα, επί του οποίου έχουν συμφωνήσει όλα τα κράτη-μέλη και το οποίο έχει γίνει αποδεκτό ως το μοναδικό σύστημα σήμανση για του σιδηρόδρομους. Ε, ουσιαστικά έχουμε μία ε, τις ίδιες ε, προδιαγραφές ε, ουσιαστικά θα έχετε ακούσει για το baseline 3 αλλά ίσως ε, κάποιοι, θα έχετε ακούσει ότι έχουν γίνει και άλλα προγράμματα σε ό,τι αφορά στο baseline 2. Σιγά σιγά θα πάμε στο ε, baseline 3 ε, το οποίο θα είναι το κανονικό ε, το τελικό σύστημα. Επίσης αυτό που αποφασίσατε εσείς τα κράτη-μέλη είναι να υιοθετηθεί και το τεχνικό, ο τεχνικός επιλώνας του τέταρτου πακέτου για τους σιδηροδρόμους έτσι ώστε να υποστηριχθεί η εφαρμογή των προδιαγραφών του ERTMS και προκειμένου να ενισχυθούν και αρμοδιότητε τη σχετική αρχή έτσι ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει ε, τι υποχρεώσει διαλειτουργικότητα. Κάτι ακόμα που κάναμε προκειμένου να υπάρξουν περισσότερε δυνατότητε αξιοποίηση αυτού του RTMS είναι αυτή η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Εξάπλωση του European Deployment Plan, στο πλαίσιο του οποίου έχουμε θέσει κάποιου πολύ σφιδόδοξου στόχου εντό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλος βαθμός λεπτομέρειας όπου λέμε τι ακριβώς υλοποιείται, τι ακριβώς σχεδιάζεται και μέχρι πότε ε, το κάθε βήμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Κάτι ακόμα που έχουμε κάνει γιατί βέβαια πρόκειται για, κάτι, για ένα ζήτημα όχι μόνο τεχνικό αλλά και χρηματοδοτικό. Έχουμε business cases, ε, δηλαδή ορισμένε περιπτωσιολογικέ ε, μελέτε σε ό,τι αφορά την, ε, την, δυνατότητα επένδυση σε αυτό το τομέα. Δηλαδή ουσιαστικά εξετάζουμε ποια, θα είναι, ποιες, ποια θα είναι τα έσοδα δηλαδή, για του επενδυτέ, όχι μόνο για τα κρατημέλη αλλά και για εκείνου που θα κληθούν να επενδύσουν. Τώρα, ποια είναι τα ωφέλη τα οποία αναμένουμε να αποκομίσουμε από αυτή την εφαρμογή. Καταρχήν θα υπάρχει αυξημένη ικανότητα αυτομάτω με την εφαρμογή αυτού του συστήματο. Πριν από 10 χρόνια, όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, είχαμε αναφερθεί σε ε, εκτιμήσει για αύξηση κατά 40-50% των δυνατοτήτων. Ενώ με βάση την σημερινή μελέτη μπορούμε να έχουμε συμπληρωματικά 20-40% αν όχι περισσότερο. Ε, δεύτερο, μπορούμε να έχουμε περισσότερη αξιοπιστία, τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την, ε, τον άξονα εκεί του, του, του Βερολίνου, η αξιοπιστία έχει βελτιωθεί ε, πολύ συγκριτικά με το προηγούμενο σύστημα. Ταυτόχρονα έχει μειωθεί σημαντικά το κόστος συντήρησης, γιατί αν εξετάσουμε ε, επιμέρους ε, προδιαγραφές οι οποίες ε, θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο του baseline 3, ουσιαστικά θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από μία σειρά από όλες ε, προδιαγραφές που αφορούσαν το παλαιότερο σύστημα σήμερα. Και επίσης υπάρχουν βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Γιατί δεν μιλάμε εδώ για βελτίωση κατά 2 έως 3%, μιλάμε για πολύ ψηλότερα ποσοστά βελτίωσης. Κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με τεράστιε τις επενδύσεις και βέβαια ε, δεν αφορά μόνο ε, έναν ε, άξονα, αλλά πολλαπλούς. Τι θα πρέπει να κάνουμε σε ό,τι αφορά τη διατηρητικότητα Φυσικά θα έχουμε το ERTMS, το οποίο θα αυξήσει τη διαλειτουργικότητα, αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν και μία σειρά από περαιτέρω μέτρα, τα οποία δεν χρήζουν τόσο υψηλών δαπανών, και τόσο υψηλών επενδύσεων, αλλά τα οποία μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω και σημαντικά την ε, διαλειτουργικότητα. Και εδώ αναφέρομαι ειδικότερα σε διασυνοριακέ ε, προσπάθειε, για παράδειγμα διαδικασίε αδειοδότηση και ούτω καθεξής. Γιατί δηλαδή θα πρέπει ε, κανεί να για ένα ταξίδι από τη Γαλλία στη Γερμανία ή από το Βέλγιο προς τις κάτω χώρες να υπάρξει, να χρειάζεται να περάσει κανείς από ένα πολύ επαχθές σύστημα διοδότησης. Έχουμε κάποια τρένα μήκου μήκους 450 μέτρων. Ε, μπορούμε να πάμε στα 700 μέτρα ε, και αυτό σημαίνει ε, ακόμα υψηλότερη παραγωγικότητα. Άρα λοιπόν υπάρχουν μία σειρά από περαιτέρω υπερβάσει εντό εισαγωγικών που μπορούμε να κάνουμε και οι οποίες θα ενσωματωθούν μέσα σε αυτό το σχέδιο. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ τώρα σε ένα σημείο καμπής, σε ένα κρίσιμο σημείο και επιτρέψτε μου εδώ να επιμείνω ε, και να ζητήσω από εσά ως μέλη του Κοινοβουλίου να μας δώσετε τα ε, όσα πρέπει να επιτύχουμε ως το 2023. Γιατί ως τότε, γιατί θέλουμε να καταδείξουμε τόσο από τεχνική όσο και από επιχειρησιακή άποψη το σύστημα πράγματι θα λειτουργεί έτσι ώστε το, το υπόλοιπο εκείνο το διάστημα, δηλαδή το 2023 στο 2030, θα, ε, θα είμαστε πλέον σε θα έχουμε πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε ε, τη, τα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα με τον τρόπο που ε, έχουμε προβλέψει. Άρα λοιπόν ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτή την περίοδο 2018-2023. Πρόκειται ένα ε, πρόγραμμα το οποίο θα ενώσει ακόμα περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βελτιώσει την κινητικότητα αλλά και την οικονομία λόγω και την μείωση των σχετικών δαπανών σε ό,τι αφορά τις μεταφορές και οπότε ε, υποστηρίξτε μα, γιατί εδώ έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Ξέρουμε ακριβώ τι προτιθέμεθα να κάνουμε και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τρότμαντ, έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. εκτό μικροφώνου η μελητρία. Um, Πρώτα απ' όλα, η Rail Baltica, που είναι το βασικό έργο αυτού του ε, διαδρόμου, Ξέραμε ότι υπήρχε η κύρωση ε, μιας ε, διακυβερνητικής συμφωνίας των κρατών της Βαλτικής και υπήρξε και μια άλλη φάση για τις νέες κατασκευές ε, στις χώρες της Βαλτικής. Υπήρχε οικονομική στήριξη τάξης 1,6 δις το οποίο κατανεμήθηκε στην Πολωνία και στις χώρες Βαλτικής για αυτές τις υποδομές. 3,1 δις είναι η συνολική χρηματοδότηση ΣΕΦ. Το Amsterdam Σίγλουξ, Προχωρά, προχωράνε τα έργα για την ολοκλήρωση ε, μέχρι το 2019. Μπορείτε να πάτε να το επισκεφτείτε αν θέλετε. Αυξάνεται ο αριθμό των καινοτόμων έργων σε όλο το διάδρομο. 23 έργα από τα 78. Αυτό δείχνει ότι ε, ο διάδρομος αυτός ε, έχει άμεση σχέση με την καινοτομία. Και βλέπετε ότι αυτός ο διάδρομος έχει αντίκτυπο και στην ενίσχυση της οικονομικής διάστασης, ε, στην απασχόληση, 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας κάθε χρόνο μέχρι το 2030. Και βλέπουμε ότι οι διάδρομοι μπορούν να ε, τονώσουν την καινοτομία λαμβάνοντας υπόψη και αντιμετωπίζοντας ε, τις τεχνολογικές προκλήσεις. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσουμε καινοτόμε λύσεις σε, με συντονισμένο τρόπο μεταξύ κρατών και υπάρχουν και ορισμένες εμβληματικές πρωτοβουλίες, εμβληματικά έργα ε, της πληροφορικής, οδικής ασφάλειας και το καθεξής σε διάφορους διαδρόμους για να ενισχύσουμε αυτές τις ε, διακυβερνητικές, ε, μάλλον διασυνοριακές οργανωτικές λύσεις. Έχουμε εργαστήρια για εναλλακτικά καύσιμα, ψηφιακή κινητικότητα και ε, υποδομές ε, μεταφοράς εμπορευμάτων, αυτόνομη οδήγηση και το Βέβαια, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με φύ τρόπο τον ελάχιστο ε, διαθέσιμο αστικό χώρο και απαιτείται συνεργασία και των πόλεων και περιφερειών. Τώρα σε ό,τι αφορά τις υποδομές για τα εναλλακτικά καύσιμα. Εδώ οι διάδρομοι μπορούν να διευκολύνουν την εφαρμογή των πολιτικών αξιοποιώντας ε, στο έπακρο την διαθέσιμη χρηματοδότηση, κάνοντας αναλυτική χρήση των υποδομών, ε, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις ε, στην αγορά των κρατών μελών. και για τα clean vehicles και σε άλλες ε, ε, αντίστοιχες εμπειρίες μάθαμε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την ε, καθαρή μετακίνηση στην Ευρώπη. Είχαμε σε 13 κρατημέλη 340 σταθμούς ε, φόρτισης σε πολλούς ε, διαδρόμους και πιο, με βάση και τον Orient Med μετά το Mega E, 200 σταθμοί Ultra Charging σε 13 κράτη μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο κεντρικό δίκτυο με μόχλευση μεγαλύτερη πρωτοβουλία σε 20 χώρε. Και ο Ρέμεμπου 2 στο Ρότερνταμ συμβάλλει στην ανάπτυξη ενό ε, πλήρου ε, συστήματο με υποδομέ φόρτιση ε, και καθαρή ενέργεια. Αυτά τα τρία έργα βρίσκονται υπό την διαδικασία υπογραφή. Τι περιμένουμε από το ΣΕΦ. Το ΣΕΦ μεταφορέ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τα βιώσιμα διασυνοριακά έργα, 14 στο δικό μου διάδρομο. Θα πρέπει να διατηρηθεί αυτό ο στόχο για να πετύχουμε του στόχου μα για αποτελεσματική και αποδοτική ε, διασυνοριακή μεταφορά και σύστημα μεταφορών. Θα πρέπει να ε, ωφελούνται στόχοι όπω ε, τα εμβληματικά έργα η ανάμειξη του ΣΕΦ με άλλα ευρωπαϊκά συστήματα όπως το ΕΦΣΥ θα είναι χρήσιμα για προγράμματα που φέρουν ε, ε, ωφέλη και κέρδη βράχη ή μέσο πρόθεσμα και με την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Μετά έχουμε ε, μηχανισμούς προώθησης μη παραδοσιακών έργων όπως ε, στην τομέα της υλικοτεχνικής υποστήριξης και σε άλλους, ε, που εδώ πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό του φορέα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Τρότμαν. Τελευταίος ομιλητής. Ο κύριος Μπάλλας για πέντε λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι υπεύθυνο για τον διάδρομο Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος που ξεκινάει από το Μπέλφαστ, Γλασκόβι, Εδιμβούργο και φτάνει έως ε, την Ηλιόλου στη Μασαλία. Ε, Παρίσι, Λίλη, Λουξεμβούργο, Βέλγιο και κάτω χώρες ε, συμμετέχουν επίση. Πρόκειται για μια, μια πολύ πυκνή περιοχή, διότι τα έξι αυτά κράτη-μέλη εκπροσωπούν 20% του πληθυσμού τη Ένωση της Ένωση των 28 και 26% του ΑΕΠ. Και αυτό φαίνεται βεβαίως και από το πόσες διασυνδέσεις υπάρχουν. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή όπου ε, περιλαμβάνονται περίπου 7.000 χιλιόμετρα σειροδρομικού δικτύου, 4.000 χιλιόμετρα ε, θαλασσίων οδών, το ίδιο σε ό,τι αφορά τις χερσαίες οδούς, 25 ε, ε, εσωτερικά λιμάνια, πάρα πολλά εξωτερικά λιμάνια. Έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εργασιών. Μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το τρίτο σχέδιο δράσης. Ε, έχουμε πάνω από 350 project και επενδύσεις της τάξεως των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ε, τα βασικά θέματα, κάποια παραδείγματα πρώτα μάλλον, σύνδεση μεταξύ ε, του ΣΕΝ και του ΣΧΑΡ, ε, βελτίωση της πρόσβασης ε, στο Παρίσι, Δουνκέρκη, Βέλγιο, κατοχώρες, ε, αποτελεσματικό ποταμίσιο δίκτυο, η σύνδεση με την ενδοχώρα των λιμανιών και πολλά ακόμα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βασίζεται κυρίως σε θαλάσσιες οδούς, διότι δαπανούμε 70% των χρημάτων που έχουμε στη διάθεσή μας για τα εσωτερικ, τις εσωτερικές θαλάσσιες και τα λιμάνια. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα ε, της ε, διτής μεταφοράς. Αυτό ε, φέρνει νέα αποτελέσματα, θέτει και νέους στόχους, δίνει μια νέα διάσταση. Για πρώτη φορά στην ιστορία των ευρωπαϊκών μεταφορών έχουμε μια στενή διασύνδεση μεταξύ σιδηροδρόμων, χερσαίων μεταφορών, ιστορικών θαλασσίων οδών, λιμανιών, αερολιμένων και συνδυάζουμε ε, διασυνδέσεις οδικές και σιδηροδρομικές, γέφυρες, δυνατότητε σύνδεση μεταξύ της αντοχώρας και των λιμανιών. Όλα, συνδέονται μεταξύ τους. Οι στόχοι είναι πολλαπλοί πολλοί, οι πολλοί τρόποι μεταφοράς ε, περιλαμβάνουν ε, πολλά νέα στοιχεία, έξυπνες, ε, έξυπνα εισιτήρια, προσβασιμότητα, αποδοτικότητα, μείωση των σημείων συμφόρησης, πέρασμα από τις οδικές στις δρομικές μεταφορές και βεβαίως έχουμε και τα modal nodes ε, αστικά κυρίως, ε, ε, ζητήματα κυκλοφοριακού, όπου και πάλι πρέπει να μειώσουμε τα σημεία συμφόρησης και προστασία του περιβάλλον. Το 2018 είναι το έτος των πολλαπλών τρόπων μεταφοράς για την DG Move. Δίνουμε μεγάλη έμφαση σε αυτή τη σημαντική πτυχή και να τελειώσω αναφερόμενο σε μια από τις βασικές ανησυχίες μας ε, αφορά, το, αφορά κάτι μοναδικό στην ιστορία της Ένωσης, το Brexit. Εγώ εκπροσωπώ εδώ το μόνο διάδρομο που περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο και επειδή πολλά στοιχεία των διαπραγματεύσεων στο Brexit παραμένουν ασαφή, εμείς επικεντρωνόμαστε σε ζητήματα όπως το πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε νέα εμπόδια στις μεταφορές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα Ιρλανδικά σύνορα, πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε ε, την ε, ε, διασύνδεση μεταξύ Ιρλανδίας και της υπηρετικής Ευρώπης ε, πώς με τον συνάδελφο Brian Simpson θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις θαλάσσιες αρτηρίες με όλα αυτά τα ζητήματα και παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν εμείς θεωρούμε ότι η συνέχεια και η ακαιρεότητα αυτού του διαδρόμου πρέπει να παραμείνει στο μέτρο του δυνατού. Αυτό θα εξαρτηθεί βεβαίω από του μελλοντικού οικονομικού διαγωνισμού μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση. Οικοδομούμε εδώ το μέλλον και προσπαθούμε ε, να ξεπεράσουμε όχι μόνο αυτές τις δυσκολίες αλλά και τις ε, ε, αλλαγέ τι κυβερνητικέ. Διότι εμεί εκπροσωπούμε το μακροπρόθεσμο συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι βέβαιο ότι ο διάδρομο Βόρεια Θάλασσα Μεσογείου είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Τέλο, πρόκειται για ένα διάδρομο ο οποίο συνδέεται με τέσσερι ακόμα μεγάλου ε, διαδρόμου ε, ε, στο πιο πολυπληθέ ε, και βιομηχανοποιημένο κομμάτι τη Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. ευχαριστώ και τον κύριο Μπάλλα. Θα δώσω τώρα το λόγο στα μέλη μα και θα ξεκινήσω με τον Βιμ Βαντενκάμπ. Ε, Δυστυχώ ε, πρέπει να πάω στην Επιτροπή Απασχόληση, διότι εκεί έχω πρέπει να υπερασπιστώ και το πακέτο κινητικό του. Οπότε ο, ο αντιπρόεδρο, ο κύριο Ρικέ, θα προεδρεύσει. Θα επανέλθω όμω. Θα επανέλθω. Μην στενοχωριέστε. Ο κύριος Βιμ Βάντεν Κάπ έχει το λόγο τώρα για, τώρα για τέσσερα λεπτά το πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα μεγάλη η τιμή να έχουμε εδώ τους ε, συντονιστές των έργων TNT. Ε, Προσωπική μου άποψη είναι ότι το TNT είναι ένα από τα καλύτερα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως το σώμα των συντονιστών είναι, να είναι και πιο σημαντικό από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδίω όταν συνομιλώ με τον κύριο Μπαλάς που λέει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις ε, είναι λίγο παροχημένες, ενώ οι συντονιστές, ή μάλλον είναι ε, προσωρινής φύσεως, ενώ οι συντονιστές μένουν ε, για πάντα. Γι' αυτό είναι σημαντική δήλωση. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσφέρει έργο. Γιατί γίνεται πολλής λόγος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγα όμως προσφέρουμε πρακτικά. Και νομίζω ότι τα έργα εδώ είναι έμπρακτα. Στην αρχή όταν μιλούσαμε για τα TNT, μιλούσαμε κυρίως για τον σίδηρο και το τσιμέντο. Δηλαδή, οδικό δίκτυο και σιδηροδρομικό δίκτυο. Βλέπουμε τελευταία ότι ασχολούμαστε περισσότερο με την βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση. Όμως, δεν άκουσα καμία αναφορά στις μεταφορές ως υπηρεσία, Transport as a Service. Ε, ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα την, ε, πρωτοβουλία, την έκθεση πρωτοβουλίας, της CIS, ε, που κάνει λόγο για τις μεταφορές ως υπηρεσία που θα μπορούσε να ε, προποθέτει μικρότερες υποδομές, κυρίως στις πόλεις και νομίζω ότι είναι καλό ένας από τους συντονιστές να οικειοποιηθεί και αυτή την αρμοδιότητα για τις μεταφορές ως υπηρεσία και να μας πει κάτι ως προς αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπόντεβικ ε, για την παρουσίαση της έκθεσης προόδου. Συμφωνώ απολύτως ότι η απλούστευση των διαδικασιών είναι πολύ σημαντική. Εγώ προσωπικά θα έλεγα θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό το σκέλος στις προϋποθέσεις επιδοτήσεων των έργων TNT, γιατί και η Εθνική Υπηρεσία δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση ότι θα λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, βλέπω ότι πολλά έργα αυτή τη στιγμή ε, μένουν στάσιμα λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Τίποτα δεν άκουσα επίσης για την επιτυχία του ΕΦΣΙ. Είναι όντω επιτυχέ το ΕΦΣΙ για τα έργα τέντι; Κάπω το παρακάμπτεται, να περιμένουμε κάποια επιτυχία στο μέλλον. Πώ έχουν τα πράγματα. Και σημαντικό θέμα είναι και αυτό του ΣΕΦ. Από το άποψη θεωρώ ότι το καλύτερο λόμπινγκ ξεκινάει από το κράτο μέλο. Οπότε προς εσάς κύριε Μπόντεβιχ, έχετε μιλήσει με την κυρία Μέρκελ για το ΣΕΦ και κύριε Σέκη, έχετε μιλήσει με τον ε, Πρωθυπουργό τη Ιταλία για το ΣΕΦ. Κυρία Τρότμαν, εσεί μιλήσατε με τον κύριο Μακχόν για το ΣΕΦ. Και ε, κύριε Γκρό, εσείς έχετε μιλήσει με τον Πρωθυπουργό Μισελ για το ΣΕΦ. Και εσείς, ούγκρο είστε νομίζω. Μιλήστε με τον κύριο Ορμπάν για το ΣΕΦ. Ο Βίνξ πάει με τον Γκρός, Βέλγος. Διπλά λοιπόν χρήματα από το ΣΕΦ. Γιατί εάν δεν έχουμε τη στήριξη των ε, Υπουργών Οικονομικών, δεν πάμε πουθενά. Πρέπει πραγματικά να ξεκινήσει η άσκηση πιέσεων στο εθνικό επίπεδο γιατί το ΣΕΦ είναι και καλύπτει τα καλύτερα ε, έργα και μπορούμε έτσι να εξασφαλίσουμε πόρους. Ο κύριος Γκρός συμφωνεί. Κύριε Βίνξ, το ERTMS είναι ένα εξαιρετικό έργο. Και νομίζω ότι πρέπει ε, να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά πολύ κριτική υπάρχει στην πράξη σχετικά με τις διαφορές ρυθμού στην ε, υλοποίηση. για παράδειγμα, κάποιοι θα ήθελαν να... Οι Ολλανδοί θα ήθελαν να πάνε με τους Γερμανούς, το γερμανικό σύστημα, όμως ε, αυτό καθυστερούσε στο παρελθόν, η σημερινή ε, κατάσταση έχει αλλάξει, όμως ε, τι γίνεται με την διαφορά στον ρυθμό υλοποίησης. Δεύτερον, κυρία Τράουτμαν. υπήρξε έργο που αυξήθηκε ο προπολογισμό κατά 700.000 ευρώ. Τι έγινε, ποιανού ήταν το λάθος. Και μετά Brexit. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας κύριε Βάλλας. Αν μπορούμε να τους κρατήσουμε ε, με το μέρος μας για τα έργα TNT, να το κάνουμε. Ίσως να μην μας επιτρέψει ο Μπαρνιέ, αλλά μπορεί αυτό να αλλάξει το μέλλον. Κάτι τελευταίο, Πρόεδρε, για τα όσα ανέφερε ο κύριος Μπάλλα για το έτος της ε, πολυτροπικότητας. Την περασμένη εβδομάδα κάναμε μια συζήτηση στην Επιτροπή Τραν για την μεταφορά εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμου ε, στα ε, ελβετικά τούνελ. Οι Ελβετοί θέλουν για κάθε φορτηγό να ζητήσουν 323 ευρώ. Υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι μεταφορείς που πουλα, ε, πληρώνουν αυτό το ποσό και δεν πηγαίνουν ε, στο τρένο. Πώς ε, θα το επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστούμε κύριε Βαντερκάμπ. Η κυρία Σάντερ για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, τα μισά τουλάχιστον αυτό που είπε ο κ. Βαντερκάμπ θέλω ως χρόνο. Να ευχαριστήσω όλους τους δονηστές για τις παρουσιάσεις τους έως τώρα. Πρώτα απ' όλα κύριος Σέκη και ο κύριος Μπόντεβικ ε, να πω ότι βεβαίως ε, είναι στην πρώτη γραμμή ε, για το πώς θα βρούμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν αν πέρα από αυτά που γνωρίζουμε αν υπάρχει κάτι άλλο, κάποιο άλλο στοιχείο που θα μας επιτρέψει να βρούμε τα χρήματα αυτά τώρα. Διότι σε κάθε μία από τις προτάσεις, ευρωβινιέτα, ε, παραδείγματος χάρη, ε, αλλά είναι τόσο τα προβλήματα με την Ευρωβινιέτα που δεν θα έρθουν από εκεί τα λεφτά από ό,τι φαίνεται. Ε, το ρηπαίνον πληρώνει, εντάξει, καλές ιδέες, αλλά πιο συγκεκριμένα ε, δεν βρίσκουμε κάτι. Κάτι άλλο τώρα. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχει προσθεμένη αξία το ΣΕΒ, όμως ε, εδώ, όταν μιλήσαμε για τα δύο μελλοντικά project για την Ευρώπη μετά το 2020, ήταν το Erasmus Plus και το Horizon 2020. Εγώ ήθελα να βάλω το ΣΕΦ ε, με μια τροπολογία, αλλά ε, μόνο και μόνο επειδή ήξερα αυτόν που υποβάλλει τι τροπολογίες, αλλά ε, δεν φαίνεται να υπάρχει ε, υπεποίθηση για την προσθέμενη αξία αυτής της νέας ε, διαδικασίας, της συντονισμένης, της μα ε, του ΣΕΒ. Ε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να γίνει πιο γνωστό αυτό. Και κάτι άλλο τώρα. Με το Brexit δεν πρόκειται να πετύχουν να φτάσουμε στο 100% του προπολογισμού. Αυτό λένε όλοι. Ε, Βεβαίω αλλάζει από ό,τι φαίνεται το κλίμα στο Βερολίνο, λιγότερη λιτότητα, περισσότερε επενδύσει, αλλά 100% του προπολογισμού δύσκολα θα το φτάσουμε. Ε, πιστεύετε ότι πρέπει λοιπόν ήδη να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε ότι πέρα από τα χρήματα τα οποία θα μπορέσουμε να βρούμε θα, χρειαστούμε, θα χρειαστεί να υποχρεώσουμε το Συμβούλιο να μας δώσει κάποια πράγματα αυτής της αρχής ε, διασυνοριακή νομοθεσία παραδείγματος χάρη που να υποχρεώνει τα ευρωπαϊκά project ε, να έχουν κάποιες να, να από κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία θα υπερισχύει των εθνικών νομοθεσιών. Να είναι υποχρεωτικό όμως αυτό. Για το θέμα των χρημάτων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Αντί να επανέρχονται στα ταμεία των κρατών μελών, τα χρήματα αυτά να επιστρέφουν στο ΣΕΒ και να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εκ νέου, εκεί. Τρίτον, στο ΕΦΣΙ όλα αυτά που προτείνονται στο ΣΕΒ, ένα σημαντικό μέρος ε, να αφορά τις μεταφορές και τις υποδομές μεταφορών. Ε, κρατικές ενισχύσεις τώρα. Θα πρέπει ίσως να δούμε εάν μπορούμε να εξορροπήσουμε κάπως τα πράγματα. Υπάρχουν ε, κάποιες κρατικές ενισχύσεις που αφορούν ευρωπαϊκά project, ε, ευρωπαϊκούς στόχους. Ε, εκεί να είμαστε πιο ευέλικτοι. Βεβαίως για τις χώρες εκείνες που υπάρχει πρόβλημα με το έλλειμμα, ε, Ισπανία και η Γαλλία, με το Eurotouring ε, ε, να πούμε ότι ξέρετε εκεί πρέπει ο χρυσό κανόνα κάπως να τον ε, παρακάμψουμε, να τον μετριάσουμε, έτσι ώστε κάποιες απαραίτητε επενδύσεις για αυτά τα project που έχουν ήδη ξεκινήσει να μην προσθεθούν στο έλλειμμα των χωρών αυτών. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν πρέπει ήδη να σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα πέρα από τα χρήματα δηλαδή που θέλουμε να ζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο κανόνων, ε, να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά τα project, διότι όπω γνωρίζετε, ακόμα και αν είχαμε πολλά λεφτά, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούν να περάσουν επειδή προκύπτουν προβλήματα ε, διάθεσης των χρημάτων αυτών. Και κάτι ακόμα για το μέλλον. Υπάρχει κάτι εδώ το οποίο δεν το λάβουμε υπόψη μας επαρκώς. Έχω ένα παράδειγμα που αφορά την Γρανάδα, υπήρχε ένα άλλο παράδειγμα με ένα τούνελ στη Γερμανία. Ε, τα έργα στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένες φορές αφήνουν χωρίς τρένο ή χωρίς κινητικότητα, χωρίς τρόπο ε, να μετακινηθούν κάποια εδάφη ε, για κάποιο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να προσμετρήσουμε τι θα χρειαστεί να γίνει για να μην έχουμε να υπάρξει σημαντική, σημαντικός επηρεασμός της κινητικότητας σε κάποιες περιοχές, ε, είτε μιλάμε για σιδηρόδρομου, είτε μιλάμε για θαλάσσιε οδού και βεβαίω από εκεί πέρα υπάρχει το θέμα τη συντήρηση. Κάποιο να θέσει επιτάπητο για το θέμα τη συντήρηση των ευρωπαϊκών αυτών υποδομών, διότι και αυτό έχει τη σημασία του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Κυρία Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για το γεγονό ότι δεν παρευρέθηκα σε όλες τις ομιλίες εδώ, ε, γιατί ήμουν προσκεκλημένη σε μια σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές ε, ε, πλωτές οδούς, οπότε δυστυχώς μόλις τώρα καταφέρα να έρθω, οπότε δεν ξέρω... Ντομενέκ, αν θα ήθελε εσύ να αξιοποιήσει ένα μέρο τη δική μου παρέμβαση, των ερωτήσεων δηλαδή από την πλευρά τη Άλντε. δεν είμαι σίγουρο λοιπόν αν οι ερωτήσει που έθεσα έχουν ήδη απαντηθεί από του ομιλητέ. Πάντω, σε ό,τι αφορά την κυρία Τράουτμαν, ε, ε, η ερώτηση που θα ήθελα να τη θέσω είναι σχέση με αυτόν τον ε, άξονα. Είναι ευχαριστημένη με το state of play ή όχι. Για παράδειγμα, είδαμε και λίγο το ρομπότικα και στο πλαίσιο μια αποστολή τη Άλτε και θέλουμε σε κάθε περίπτωση έστω και στο απότερο μέλλον να υπάρχει σύνδεση σύνοδρομική ψηλής ταχύτητας. Μετά σε ό,τι αφορά το ε, ERTMS, ε, δυστυχώς και αυτή την ομιλία από τον κύριο Βίγκ δεν ε, μπόρεσα να την παρακολουθήσω, πάντως με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ERTMS σε ό,τι αφορά δύο συγκεκριμένες πτυχές. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τη Γερμανία, η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι ικανοποιητική, γιατί γνωρίζω πω ε, δεν λειτουργούν πάρα πολύ καλά τα πράγματα στη Γερμανία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ERTMS. Για παράδειγμα, η Αυστρία πάντοτε κινούνταν πολύ ταχύτερα από τη Βαβαρία, για παράδειγμα. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση στο ενδιάμεσο διάστημα στη Γερμανία. Ε, δεύτερο τώρα ζήτημα, πάλι σε ό,τι αφορά το ERTMS. Το Brexit ε, ε, θα έχει επιπτώσει σε ό,τι αφορά την πλήρη εφαρμογή του ERTMS ε, σε όλα τα εδάφη. Γιατί εγώ είμαι ε, αισιόδοξη ε, και ακόμα ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή δεν θα εφαρμοστεί το Brexit. Αλλά εάν πραγματικά φτάσουμε στο σημείο του να εφαρμοστεί πλήρω το Brexit, θα υπάρξει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του RTMS, επειδή δεν θα προχωρήσει εκεί πλέον η υλοποίησή του. Αυτά σε ό,τι αφορά το RTMS, αλλά και τώρα. Σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του κ. Μπαράς και την, το Ηνωμένο Βασίλειο, σε ό,τι αφορά το δικό σα άξονα, εδώ περιλαμβάνεται το Ηνωμένο Βασίλειο και εκεί θα έχουμε τεράστιε αλλαγέ, γιατί ουσιαστικά θα σπάσει εντό εισαγωγικών αυτό ο άξονα, εάν φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ΕΒ. Ε, και ε, ουσιαστικά ε, αυτή η διακοπή, αν θέλετε, του δικτύου, αυτή το που θα γίνει. Ε, κατά τη δική σα άποψη, θα έχει επιπτώσει και για την Ιρλανδία και ό,τι αφορά δηλαδή ε, την επιθυμία τη Ιρλανδίας του να μπορεί να ε, χρησιμοποιεί το δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου για να συνδέεται με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ε, δεν βλέπω βέβαια ποια είναι η λύση, αλλά θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας άποψη σε σχέση με αυτό. Ε, εντάξει, δεν πήρα το λόγο για πέντε λεπτά, αλλά δυστυχώ δεν άκουσα όλε τι παρεμβάσει, οπότε θα περιοριστώ σε αυτά τα ερωτήματα για να μην επαναλάβω ενδεχομένω κάποια από τα όσα ήδη υπόθηκαν. Ευχαριστούμε. Πίτερ, για πέντε λεπτά. Α, όχι. Ο Μάικλ. Ο κύριος Κράμερ. θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για αυτές τις ε, ε, παρεμβάσεις και να στήσω και εγώ μια κριτική απέναντι σε εμάς τους ευρωβουλευτές ότι δεν έχουμε τόσο ε, ε, πολλούς συναδέλφους ε, που παρευρίσκονται εδώ γιατί ε, βέβαια από αυτά τα προγράμματα εποφελούνται πάρα πολλά κράτη-μέρη, λαμβάνουμε κονδύλια για όλα αυτά και δυστυχώς έχουμε πολύ λίγους συναδέλφους που παρευρίσκονται σήμερα εδώ και αυτό είναι, ε, μας τροπιάζει λίγο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους συντονιστές και τη συνεργασία μας. Ε, καλό είναι εδώ να υπάρχει συνεργασία γιατί βέβαια υπάρχει αλληλεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων σας ε, και αυτών των αξών ε, κάτι στο οποίο είχαμε δηλαδή ασκήσει κριτική στο παρελθόν ότι δεν υπήρχε ο κατάλληλος συντονισμός. Από εκεί και μετά ε, σε ό,τι αφορά αυτά τα ε, προγράμματα ε, τη δημιουργία υποδομών, πάντοτε υπάρχουν κονδύλια, πάντοτε υπάρχει χρηματοδότηση, αλλά σε ό,τι αφορά τη συντήρηση δεν βλέπουμε πολλά. Και αυτό παραμένει ένα πρόβλημα. Υπήρχε στο παρελθόν και συνεχίζεται. Δηλαδή υπάρχουν επενδύσει στι υποδομέ, αλλά από εκεί και μετά τα κράτη-μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα για αυτά τα ακριβά έργα να συνεχίσουν τη συντήρησή του. Οπότε αυτό είναι μια δική μου παρατήρηση. Τώρα, κύριε Σέφη, σε ό,τι αφορά την Ευρωβινιέτα υπάρχουν κάποια ε, και οδικά και άλλα έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν όπου ε, ουσιαστικά δεν έχει εφαρμοστεί, ε, δεν έχουν εφαρμοστεί τέλη διοδίων, δεν έχει εφαρμοστεί η βινιέτα. Οπότε ε, τι σκοπεύετε να κάνετε, θα υπάρχει μια τέτοιου είδου προπόθεση ότι δηλαδή ναι θα λάβετε χρηματοδότηση αλλά μόνο εφόσον εφαρμόσετε και τέτοιου είδου βινιέτα. Η Ελβετία για παράδειγμα αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα ω προ το πώ μπορεί να χρηματοδοτήσει κανεί έργα στι συνδρομικέ μεταφορέ χρεώνοντα ένα υψηλότερο τέλο διοδίων. Τώρα κύριε ό,τι αφορά τη σύνδεση Αυστρία και Εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά. Από ό,τι γνωρίζω, ένα οδικό έργο σχολιάστηκε από τον πρώτο Γιούγκερ ε, ω προ τι υπερβολικέ επιπτώσει δεν μα αφορούν τόσο πολύ. Θα συνεχίσουμε αυτό το έργο. Πέτρο ε, Βέλα δεν ε, είχε καν το χρόνο να αναφερθεί σε αυτό και για μένα αποτελεί ιδιαίτερα προβληματικό αυτό το, ε, αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραβαίνει τις, ε, τους κανόνες τους οποίους έχει ε, θέσει η ίδια στον εαυτό Τώρα, κύριε Γκρόσε, 30% ε, συνδρομικές μεταφορές δεν είναι χαμηλό αυτό το ποσοστό. Πώς θα επιτύχουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Θα συνεχίσει δηλαδή το ποσοστό συνδρομικών μειούμενο αντί να αυξάνεται. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας τότε σε σχέση με το περιβάλλον. Και σε ό,τι αφορά τα διασυνοριακού χαρακτήρα προβλήματα, για μένα εδώ το ζήτημα δεν είναι μόνο τεχνικό, αλλά είναι και ζήτημα πολιτικής βούλησης, αλλά και ε, ε, ε, τιμολόγησης. Για παράδειγμα, αν ε, πάμε ε, ε, διαβώ τα σύνορα και πάω μέχρι τον Γκέρλιτ για παράδειγμα για μια σχεδόν ίδια απόσταση πληρώνω τη διπλάσια τιμή σε σύγκριση με μια απόσταση εντό τη ίδια χώρα. Οπότε αυτό συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα. τώρα κύριε Βίνκ, πράγματι είναι θετικό το ότι ακούσαμε ότι εφαρμόστηκε το σύστημα σε 70.000 χιλιόμετρα και ότι χάνουμε πραγματική εναρμόνιση αφού μέσω ERTMS δεν υπάρχουν τόσο ε, πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Το ε, ερώτημα που θα ήθελα να θέσω ε, έχει επιληθεί αυτό το ζήτημα μεταξύ Eurostat και ERA δεν υπάρχει αυτός ο εγωισμός μεταξύ αυτών των αρχών των εισαγωγικών που δεν θέλαν να μοιράζονται μεταξύ τους τα σχετικά δεδομένα. Ε, πράγματι ισχύει πλέον αυτή η συνεργασία μεταξύ τους, μεταξύ γύρω στα Ε, από εκεί και μετά υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα στην αρχή ε, του, της εφαρμογής του συστήματος ε, ε, μεταξύ ε, Βερολίνου και Μονάχου. ήταν και πολύ λυπηρό αυτό που είχε συμβεί. Θα ήθελα να μου πείτε αν πράγματι έχει επιληθεί αυτό το πρόβλημα. τώρα, σε ό,τι αφορά τη Ρέλ Μπάλτικα, κυρία Τράουτμαν, απευθύνομαι σε εσά ουσιαστικά από ό,τι ακούσαμε έχει συναυθεί η σχετική σύμβαση και ούτω καθεξής. Αλλά έχει καθοριστεί συγκεκριμένη γραμμή. Υπήρχε και μια ε, διαφορά απόψεων με την Εστονία. Τελικά, ποια θα είναι η γραμμή, θα περνάει από το Πέρνου ή όχι. Έχει επιληθεί αυτό το ζήτημα. Ε, θα με χαροποιούσε το να ακούσω ότι πράγματι επιλύθηκε. Ε, κύριε Μπάλλα τώρα, 70% ε, ε, μα είπατε πλωτέ οδοί και θαλάσσιοι λιμένε. Εντάξει, εδώ το σχετικό ερώτημα το έθεσε συνάδελφο Μάσινερ, οπότε δεν θέλω να το επαναλάβω. Για μία ακόμα φορά ευχαριστώ του ομιλητέ για αυτέ τι παρεμβάσει και θα παραμείνουμε βέβαια σε επαφή. Ευχαριστώ κύριε Στέλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσουμε όλους ε, τους συντονιστές. Πραγματικά σημαντική η σημερινή συνεδρίαση. Θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή γειτονία. Γιατί έγινε πολύ λόγος για στενοπούς και επίλυση αυτών των προβλημάτων μεταξύ κρατών μελών, αλλά τώρα πρέπει να εξετάσουμε ευρύτερα τι συμβαίνει και με τους γείτονες, ιδίως στις χώρες της ε, Ανατολικής Τερικής Σχέσης ε, και τα Δυτικά Βαλκάνια. Εκεί θα ήθελα να επικεντρωθώ και να, να απευθύνω τα ερωτήματά μου προς τον κύριο Γκρός και την κυρία Τρότμαν, γιατί νομίζω ότι αυτοί οι δύο διάδρομοι αφορούν αυτές ε, τις περιοχές σε ό,τι αφορά τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα θυμάστε, αν δεν με πατάει και με μνήμη μου, ότι είδαμε επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που έγινε στη Σύνοδο Κορυφής της Δυτικά Βαλκάνια στη Βιέννη ε, υπό την ευρύτερη διαδικασία του Βερολίνου. Ήταν ε, μια πολύ θετική κίνηση και εξέλιξη σε ό,τι αφορά ε, την ευρύτερη περιφέρεια, αλλά εσείς ως συντονιστέ. θα ήθελα να με ενημερώσετε. Βλέπετε να έχουν υπάρξει βελτιώσεις σε ό,τι αφορά Βαλκάνια. και στις χώρες τη ανατολική Τερικής σχέση, γιατί υπήρχαν πολύ ωραίε ιδέες για την Ουκρανία, τη Μολδαβία, αλλά στην πράξη τι βλέπετε. Όταν συνομιλείτε με τα ενδιαφερόμενα μέρη ή τι κυβερνήσεις. Σχεδόν το ξέχασα, αλλά υπήρχαν φήμες για την ανάγκη ε, διεύρυνση τη εντολή σα για αυτέ τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Και θυμάμαι, κύριε Γκρόζο, ότι μια φορά μου είχατε πει ότι είχε πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ήταν τεχνικό ζήτημα που θα πρέπει κάπω να επικαιροποιήσουν ε, την εντολή σα. Για να συμπεριλάβει και αυτή την ε, αρμοδιότητα, την ευρύτερη δικαιοδοσία. Συνέβη αυτό τελικά. Δεν το παρακολούθησα. Και προς τον κύριο Βίνκ, ένα ερώτημα για το ERTMS. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ νέων και παλαιότερων κρατών μελών στα ζητήματα μεταφορών. Για την ε, περαιτέρω ανάπτυξη του ERTMS εντοπίστηκε και εδώ διαφορές μεταξύ νέων και παλιών κρατών μελών ή ανατολικών και δυτικών σε ό,τι αφορά ε, την διάδοση και εφαρμογή των προτύπων ERTMS. Ευχαριστούμε κύριε Δεδί. Για τρία λεπτά ο κύριος Κύρκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριος Βαντενκάμπ, τα προσυπογράφω και τα εύσημα για το πάνελ. Μέχρι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα υποβάθμιζε τους σιδηροδρόμους προς όφελος των οδικών αξώνων και των κατασκευαστών όπως επίσης είχε αρνητική στάση για τις ιδιωτικοποιήσεις στα πλαίσια του πελατειακού κρατισμού 40 χρόνων. Τον τελευταίο καιρό έχει, αλλάξει το κλίμα. Ιδιωτικοποιήσεις στο λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι Θεσσαλονίκη, Κινέζοι, Γάλλοι, Γερμανοί, οι Ιταλοί έχουν αναλάβει τα τρένα. Ολοκλήρωση ηλεκτροκίνηση μέχρι το 19 σε όλο τον βόρειο-νότιο άξονα. Καινούριο project με σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βουλγαρία, Λαϊμάνια, ε, Μπούργκας και Ρούσε Βλέπουμε δηλαδή πως το τοπίο αλλάζει εντελώς. Επίσης σύνδεση του Δούναβη μέσω του Αξιού με τη Θεσσαλονίκη, παράκαμψη του Βόσπορου με τη συνδρομική γραμμή που σας ανέφερα από ένα, πάρα πολύ, έργο με πάρα πολύ ιδιωτικό ενδιαφέρον. Βλέπουμε λοιπόν πως και projects τρέχουν και η θέση της Ελλάδας αλλάζει. Ε, αυτό που μέχρι τώρα ήμασταν αυτοί που βλέπαμε τα τρένα να περνούν, και δεν ακολουθήσαμε αυτό που πολύ σωστά ο κύριος Κράμερ λέει άμα κινείται βάλτε σε τρένο για να είμαστε και περιβαλλοντικά πιο σωστοί αλλά και πιο οικονομικοί. Τώρα έχει αλλάξει τελείως αυτή η κατάσταση και γι' αυτό ακριβώς η υλοποίηση των διαδρόμων όπως ε, τους περιέγραψε ο κύριος Γκρός και οι καθυστερήσεις πρέπει να δώσουμε και το παραπάνω για να μπορέσουμε να να μειώσουμε και τα εμπόδια που φέρνει η πανταχού παρούσα γραφειοκρατία και θα ήθελα λίγο παραπάνω ε, λόγια από εσά γι' αυτό. Επιπλέον, στο θέμα που είπε και ο συνάδελφο για τα Δυτικά Βαλκάνια, τώρα βλέπουμε πώ και με την βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράμε σε μια ε, πιθανή λύση του προβλήματος που είχαμε όπως όλοι γνωρίζετε με την πρώην Ιουσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στη βάση ενός σύνθετου ονόματος και απάλληψης του αλυτρωτισμού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως και προχωράμε σε μια επίλυση των διαφορών με την Αλβανία πάλι με την συμπαράσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα της ε, οικονομικής ζώνης. Αυτό κάνει και την Ελλάδα όπως είναι ήδη η Βουλγαρία όπως είδαμε τη Βουλγαρική Προεδρία αρρωγό στην προσπάθεια που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα έξι σημεία, ένα από τα οποία ήταν οι μεταφορέ, ώστε να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων για μια ενδεχόμενη κάποια στιγμή στο μέλλον ένταξη που είναι πάρα πολύ σημαντική και για τη χώρα μου. Γι' αυτό παρακολουθούμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι γίνεται. Ελπίζουμε καθυστερήσει που είχαν σημειωθεί, ειδικά στι περιοχέ Ρουμανία, Βουλγαρία και τη σύνδεση με την ήδη καθυστερημένη Ελλάδα που τώρα όμω αλλάζει σελίδα, να μπορέσουμε να τι εξαλείψουμε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Euh, Ευχαριστούμε κύριε Κύρκο. Κλείνουμε αυτό τον ε, κύκλο παρεμβάσεων με τη δική μου παρέμβαση. Κάποιες ερωτήσεις και απολευράζουμε, λοιπόν στους κυρίους ε, Μπόντεβικ και Σέκη για τα οικονομικά. Επιμείνατε ιδιαίτερα στη σημασία των ε, εσωτερικών και εξωτερικών ρυθμίσεων και κανονισμών σε ό,τι αφορά και τα χρηματοδοτικά μέσα, αλλά και έξω τι συμβαίνει δηλαδή στις αγορές. Αυτό είναι σημαντικό. Όλοι οι συνάδελφοι εξέφρασαν προβληματισμό σε ό,τι αφορά τον όγκο ε, των επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων που θα, μπορούσαμε να, πρέπει να διατηρήσουμε ε, και συμμερίζομαι και εγώ αυτόν τον προβληματισμό και την ανησυχία. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής η χρηματοδότηση των υποδομών μεταφορών από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλούς ε, κύκλους και πολλά επίπεδα γιατί ε, έχουμε ακόμα και περιφερειακά ταμεία, ταμεία συνοχή, και για τη συνοχή και για το EDF. Έχουμε λοιπόν πολλούς τρόπους ε, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν διακυβέρνησης που είναι πολύ σημαντικό. Και η θέση που έχετε εσείς ως συντονιστές είναι να βλέπετε ποιος θα συντονίζει όλα αυτά. Έχουμε την εντύπωση ότι δεν υπάρχει αυτός ο συντονισμός, γιατί η διακυβέρνηση αυτή δεν είναι του ίδιου χαρακτήρα. Δηλαδή, η διακυβέρνηση του ΣΕΦ είναι κεντρική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η αποκεντρωμένη διακυβέρνηση των Ευρωπαϊκών ε, Ταμείων είναι διακυβέρνηση σε επίπεδο κρατών μελών. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι πώς μπορούμε να τα συντονίσουμε όλα αυτά. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Και κατά πόσο υπάρχει διαφορά, φαντάζομαι πως ναι, μεταξύ της κεντρικής και αποκεντρωμένης διακυβέρνησης. Γιατί Έχουμε πολλά επίπεδα διακυβέρνηση χρηματοδότηση και αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Η δική σα θέση ποια είναι. Θεωρώ απολύτως ε, ζωτική σημασία σε αυτό το θέμα. Είδαμε και στο τελευταίο στο δημοσιονομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική, ουσιαστικά είχε καταργηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης υποδομών μεταφορών από ε, τα ταμεία του ERDF. Μα είναι τρελό. Και κανείς δεν έχει πει τίποτα. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της πολυεπίπεδης χρηματοδότησης. Περνάει ο χρόνος για το ERTMS. Πρώτον, τα δίκτυα χρηματοδότησης του ERTMS, όπως σωστά είπε και ο κύριος Βίνκ, είπατε ότι είναι ένας από τους ε, λίγους κλάδους όπου υπάρχει η απόσβεση της επένδυσης. Ε, αυτό έγινε επειδή έχετε διαμορφώσει ε, συνέργειες με τον ιδιωτικό κλάδο ή επειδή αυξήσατε την ικανότητά σας, αυξήσατε τις επιδόσεις στις υπηρεσίες. Αναφέρατε διάφορα στοιχεία, αλλά αυτό το 30% είναι πολλά χρήματα. Οπότε, μήπως στο συνδρομικό δίκτυο θα έπρεπε το ERTMS να έχει ένα διαφορετικό γνώμονα. Δεύτερον, όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να συμμετέχουν στο σύστημα. Αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε ότι ή έχετε προτάσεις να κάνετε προς αυτό. Τρίτον για το ERTMS, Baseline A, 1, 2 3 γιατί όλοι οι πάροχοι μιλούν για την 2, ε, εντάξει, έχουμε βρει τη σταθερότητα, θα περάσουμε στην 3. Κάποια στιγμή θα σταματήσουμε αυτά τα τέλη, γιατί ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα των ε, παρόχων. Ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε και στην baseline 6 πριν ε, δούμε αν θα δεσμευτούμε. Μετά για την κυρία Τρότμαντ. ποια είναι η γνώμη σας για την για τις προτάσεις ε, των χωρών της Βαλτικής ε, σε ό,τι αφορά τις, τους ρωσικούς άξονες που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Και κάτι τελευταίο για τον κύριο Μπάλας. Υπάρχουν εργασιακές σχέσεις και συνεργασία με την ομάδα Μπαρνιέ. Και αν μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα προς αυτό. Ο κύριος Κράμερ θέλει το λόγο για ένα λεπτό. Εκτός μικροφώνου, κύριος Κράμερ. Une minute en micro, non, oh. ναι, ο επικεφαλής ε, των σιδηροδρόμων έλεγε 10.000 ε, ε, χιλιόμετρα ERTMS στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ούτε μία ένα σιδηρόδρομο ο οποίο ουσιαστικά να μπορεί να μεταβεί από το ένα σημείο στο άλλο. Τελικά αυτό εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. Παραμένουν αυτέ οι διαφορέ ή όχι. Ευχαριστούμε. Τώρα στρέφουμε προ του συντονιστέ μα. Θα του δώσουμε και πάλι το λόγο για τέσσερα λεπτά έκαστο αυθαίρετα το λέω, αλλά γιατί όχι, για να απαντήσουν ε, στα ερωτήματα που τους έχουμε απευθύνει και για να μας δώσουν τα τελευταία σχόλιά τους. Παρακαλώ κύριε Μπόντεβικ και Σέκη. Αφού είστε δύο, ένα πεντάλεπτο συνολικά θα έλεγα. Τότε θα ξεκινήσω με τα ερωτήματά εκείνα για τα οποία θα μπορούσα να απαντήσω απευθείας στον κύριο Βαντεκάμ να πω ότι σε ό,τι αφορά το ΕΦΣΙ, το Μέσο Στρατηγικών Επενδύσεων, ε, τα προγράμματα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές είναι πολύ περιορισμένα, κυρίως εστιάζει σε ζητήματα ενέργειας και επιχειρηματικότητας. Οπότε πρόκειται μόνο για ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και γι' αυτό είπαμε ότι θέλουμε να βασιστούμε περισσότερα σε αυτήν την ιδέα του blending, για παράδειγμα της μεκτής χρηματοδότησης. Ε, ε, είχε αναφερθεί γι' αυτό και σε ό,τι αφορά τον, ε, τον αξονά μας και εκεί είχαμε αναφερθεί σχετικά ζητήματα στην έκθεση CBS. Είχαμε πει από, το, από τα 50 δισεκατομμύρια 20 συμπληρωματικά 20 δις από το ΣΕΦ και ε, περίπου ίδιο ύψος χρηματοδότηση από την πλευρά των κρατών μελών. Εάν ε, καταφέρναμε να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο συγχρηματοδότησης και πάλι η αναλογία θα ήταν ένα προς πέντε. Οπότε χρειαζόμαστε μία πολύ σταθερή χρηματοδότηση από το μηχανισμό, από το ΣΕΦ. Αλλά βέβαια γνωρίζουμε από την άλλη πλευρά ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα ακριβώ εν ώψη και των διαπραγματεύσεων για τον Brexit και ούτω καθεξή. Επίση, ε, στην κυρία Αγιάλα Σέντερ να πω το εξή ναι, ήδη έχουμε ε, επιτύχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. 97% ε, ε, επίπεδα απορρόφησης των κοντιλίων. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για κάθε κράτος μέλος που προέβη σε μια τέτοια επένδυση ουσιαστικά σε επίπεδο μακροοικονομικής σημασίας λαμβάνει τα διπλάσια σε επιστροφή. Και εδώ βέβαια έρχομαι στο επόμενο ζήτημα, τη διασυνοριακή συνεργασία. Πράγματι θα πρέπει να βελτιώσουμε εδώ τα πράγματα γιατί ο χρονικός συντονισμός ε, και, η, και η συνεργασία μεταξύ των δικτύων είναι απολύτω απαραίτητα. Ε, και ε, κύριε Κράμερ, αυτό που είπατε, όχι, εγώ δεν το άκουσα, αλλά εκείνο που αναφέρεται ε, και στο permitting study, δηλαδή στην άδεια ε, και εξακολουθεί να αποτελεί δική μα ε, αξίωση, είναι το, τα έργα τα οποία έχουν γίνει και σε επίπεδο προκήρυξης των διαγωνισμών και σε επίπεδο αδειοδότησης να υπάρξουν πιο απλά ε, συστήματα. Γιατί σε ό,τι αφορά και το πρόβλημα μεταξύ Τσεχία και Αυστρία, ακριβώ εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Στο ότι δηλαδή η διαδικασία αξιολόγηση είναι πολύ περίπλοκη, το ίδιο πράγμα το ε, πρέπει να αξιολογηθεί τρει διαφορετικέ φορέ και για κάθε ε, μία από αυτέ τι τρει αξιολογήσει μπορεί να υπάρξει και προσφυγή. Αυτό είναι που περιπλέκει τα πράγματα. Άρα λοιπόν θέλουμε ναι υψηλά πρότυπα, αλλά ταυτόχρονα απλουστευμένε διαδικασίε σε ό,τι αφορά και την προτίμηση των δημοσίων και σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συντονισμό μεταξύ των συντονιστών, το, τη συνεργασία του. Ναι, υπάρχουν πράγματι εδώ αλληλεπικαλύψει ε, ορισμένων αξώνων με άλλους. Και η κανονική διαδικασία την ακολουθούμε είναι ότι όταν προβαίνουμε σε συνομιλίες ε, πάντοτε τις κάνουμε από κοινού και με τους υπόλοιπους θυγόμενους εντός εισαγωγικών συντονιστές. Και αν δεν είναι σε θέση να παρευρεθούν σε αυτές τις συζητήσεις, σίγουρα υπάρχει ένα συντονισμός μεταξύ μας ε, γιατί όλοι οι ε, συναρμόδιοι συντονιστές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα όσα συμφωνούνται είναι 100% σωστά. Έρχομαι τώρα στο ερώτημα του κ. Ρικέ. Σε ό,τι αφορά το μηχανισμό ΣΕΦ, έχουμε πολύ σαφή εράρχηση προτεραιοτήτων. Θέλουμε δηλαδή να επιτύχουμε συγκεκριμένους στόχους και θέλουμε σε κάθε περίπτωση το κεντρικό σύστημα να, είναι, ε, να, να τεθεί σε λειτουργία. Ενώ σε ό,τι αφορά τι περιφερειακέ διασυνδέσει, ε, τα πράγματα αλλάζουν. Γιατί υπάρχουν πολύ ισχυρά εθνικά συμφέροντα και αυτό σημαίνει ότι σε, ε, στο πλαίσιο κάθε αξίωση που κάνουν δεν είναι πάντοτε δεδομένη η ευρωπαϊκή υπεραξία. Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να εστιάσουμε στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Όχι αποκλειστικά μένα, αλλά σε ό,τι αφορά για παράδειγμα περιφερειακού χαρακτήρα αξιώσει, πάντοτε να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ακριβώ στη σύνδεση με τον άξονα. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτυγχάναμε περισσότερα με τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μα ε, και σε ό,τι αφορά ε, τι υπηρεσίε ε, μεταφορών. Αυτό που είπατε, πράγματι οι μεταφορέ είναι υπηρεσίε που αποτελούνται από software, από λογισμικό και hardware, εξοπλισμό από την άλλη. Ε, και οι συντονιστέ ενδιαφέρονται μεν για το hardware, για τον εξοπλισμό, το υλισμικό, αλλά από την άλλη πλευρά μα ενδιαφέρει και το software, το λογισμικό, γιατί ε, το κατάλληλο λογισμικό μπορεί να καταστήσει αυτό το hardware, το λογισμικό πιο ε, λειτουργικό. Ε, και νομίζω πως ε, αυτό μπορεί να αποτελέσει μια, ένα καλό σκεπτικό ως προς το πώς μπορούμε να επενδύσουμε αυτά τα κονδύλια στο μέλλον. <laughs> Ο κύριος εκεί. Ναι, να προσθέσω κι εγώ ένα-δυο πράγματα σε αυτά που είπε ο κύριος Μπόντεβιγκ. πρέπει να προσπαθήσουμε προφανώς να εμπλέξουμε εδώ και τους υπουργού οικονομικών. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μόνοι μας αδόν Κιχώτης. Έτσι χρειαζόμαστε βοήθεια και τη δική σας βοήθεια. Ε, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε και κάποια στοιχεία ότι τα, χρήματα αυτά ε, ορθά δηλαδή φέρνουν αποτελέσματα σε σχέση και με άλλες ευρωπαϊκές δαπάνες. Επίσης, ε, είναι καλύτερο να δαπανώνουν τα χρήματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο από σε εθνικό επίπεδο για τέτοιου είδους project. Και αυτό με φέρνει στο σχόλιο του κυρίου Ρικέ για την διαχείριση του ΣΕΦ ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο με το Περιφερειακό Ταμείο. Θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε προς μια άμεση διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις επενδύσεις εκείνες που συνδέονται με σημαντικές, ε, σημαντικά σχέδια υποδομής. έχουμε παραδείγματος χάρη το Ταμείο Συνοχής. 10 εκατομμύρια ε, που έχουν διατεθεί με βάση τις διαδικασίες του ΣΕΒ και είναι καλή η εμπειρία. Θα πρέπει να το μελετήσουμε περισσότερο βέβαια Κανείς δεν διαμαρτύρεται πάντως ε, και θα μπορούσε αυτό να διαβριθεί περαιτέρω και ε, σε άλλα ε, ταμεία. Κυρία Σέντερ, Αγιάλα Σέντερ, πώς θα εξασφαλίσουμε όταν γίνονται αλλαγές κυβερνητικές ότι τα μακροπρόθεσμα σχέδια δεν θα ξεχαστούν. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να εκδώσει κάποιες εφαρμοστικές αποφάσεις με την συμφωνία των εθνικών κυβερνήσεων που εμπλέκονται που θα εξασφαλίζουν ότι αν, ανεξάρτητα με τις όποιες αλλαγές γίνουν ε, η δέσμευση παραμένει ε, και σε εθνικό επίπεδο, σε λόγω χώρες, ε, αλλά ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης αναφερθήκατε στον χρυσό κανόνα. Εντάξει βεβαίως είναι πολύ λεπτό το ζήτημα, πολύ ευαίσθητο, αλλά ε, τουλάχιστον με την Eurostat μπορέσαμε να διευκρινίσουμε πολύ καλύτερα κατά τη γνώμη μου το πώς ε, τέτοιου είδου επενδύσεις επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό του ελλείμματος. Υπάρχει ένα εγχειρίδιο εδώ και ένα χρόνο Όλοι είναι ικανοποιημένοι με αυτό, το καλωσόρισαν. Βεβαίως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Οποιαδήποτε πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή είναι καλοδεχούμενη. Θα προσπαθήσουμε να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι αυτό ολοκληρώνει ε, αυτά που είπε ο συνάδελφος, ε, τα συμπληρώνει αυτά που είπε ο συνάδελφος μάλλον. Εκτός μικροφώνου ο πρόεδρος όμως, και δεν ξέρουμε σε ποιον έχει δώσει το λόγο. Καταρχήν, ε, να πω ότι σε ό,τι αφορά τους ε, ε, βρισκόμαστε στο 38% σε ό,τι αφορά την πρόοδο των έργων, αλλά στο 70% σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα πράγματα σε συγκεκριμένη περιοχή είναι αρκετά δύσκολα. Και αυτό το διαπιστώνουμε ότι δηλαδή είναι δύσκολο η αξιοποίηση των σιδηροδρόμων να φτάσει σε επίπεδα αντίστοιχα με, άλλα, ε, με άλλον αξόνο. Για παράδειγμα, τα πιο ισχυρά έργα σε ό,τι αφορά του σιδηροδρόμου ε, λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Αλλά στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια ε, προβλήματα σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του, της έννοιας του άξονα σε ό,τι αφορά του σιδηροδρόμου. Άρα λοιπόν ε, η κατάσταση, αν θέλετε, και η πρόοδος εξαρτάται από το κάθε κράτος μέλος. Τώρα, επανέρχομαι ε, λίγο στην, ε, στην περιοχή των Βαλκανίων. Έχουμε μια σαφή εντολή αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχουμε. Γιατί μετά από τις συναντήσεις που κάναμε στο παρελθόν, σε ό,τι αφορά την περιοχή των Βαλκανίων, ορισμένα κράτη-μέλη θίγονται άμεσα, αλλά ε, κάποια κράτη-μέλη δεν συμφωνούσαν πλήρως με αυτήν την χαρτογράφηση. Ε, τις συνδέσεις δηλαδή που προτείνονταν στο πλαίσιο αυτών των αξώνων εντός εισαγωγικών μεταξύ δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βαλκανικών χωρών και γι' αυτό θεωρήσαμε πως ήταν σημαντικό να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία σε ό,τι αφορά τη ευθυγράμμιση των απόψεων και νομίζω πως αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Για το μέλλον προτείνω πως θα έπρεπε να υπάρξει και ένας ειδικό συντονιστή σε ό,τι αφορά την περιοχή των Βαλκανίων έτσι ώστε να εφαρμόζει τα ίδια κριτήρια με αυτά που εφαρμόζουμε σε ό,τι αφορά τα KPS και ε, οπουδήποτε αλλού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδοτική άποψη, ο, ο κύριος ο Επίτροπος Χάνη είναι ο αρμόδιος και νομίζω πως εδώ δεν υπάρχει διαφορά απόψεων ε, μαζί του. Απλώς υπάρχουν διμερού, διμερούς χαρακτήρα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν σε πολιτικό επίπεδο προτού ε, πραγματικά επιτύχουμε ε, φτάσουμε σε κάποιες επιτυχίες σε αυτόν τον ε, τομέα. Πάντως ε, αποτελεί σημαντικό αυτό το ζήτημα για μας τώρα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν. Βίμ αναφέρθηκε στις μεταφορές ως υπηρεσίες. Δεν με ακούς βέβαια αυτή τη στιγμή Βίμ, αλλά δεν πειράζει. Επαναλαμβάνω, ε, αναφέρθηκε στι ε, μεταφορέ ω υπηρεσίε. Ε, εγώ και η Κατρίν Τράουτμαν κάναμε μια ενδιαφέρουσα προετοιμασία σε ό,τι αφορά τα αστικά κομβικά σημεία, τα urban nodes και ίσω η Κατρίν να αναφερθεί σε αυτά σε λίγο γιατί πραγματικά αυτή η αυτό το concept των urban nodes είναι πολύ σημαντικό γιατί το ζητούμενο δεν είναι να αναπτύξουμε αυτούς καθεαυτούς του άξονε. θα πρέπει αυτοί οι άξονε να καταλήγουν ακριβώ σε αυτά τα αστικά κομβικά σημεία έτσι ώστε οι σχετικέ υπηρεσίε μεταφορών να συνεχίζουν να, να παρέχονται εκεί. Και νομίζω πως ε, αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε τώρα σε ό,τι αφορά το ΣΕΦ. Euh, Συμφωνούμε ότι το ΣΕΦ παραμένει ένα σημαντικό και ωφέλιμο ε, μέσο και ένας μηχανισμός ε, γιατί και ο Επίτροπος Έτιγκερ συνομίλησε μαζί μας για να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε στο μέλλον αλλά είναι γεγονός αυτό που είπε και ο Βήμ, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα τα κράτη-μέλη να πείσουμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να πούμε ότι δεν μιλούμε μόνο για χρήματα, μιλούμε για απτά συγκεκριμένα έργα. Σε κάθε χώρα να πούμε ορίστε ένα κατάλογο έργων που αναλαμβάνουμε. Κανεί δεν το κάνει αυτό. Έχουμε μια ξεκάθαρη ε, λίστα ανά χώρα. Και ότι δεν ε, μιλούμε μόνο για χρήματα, Πρόκειται για συγχρηματοδότηση για συγκεκριμένα από τα έργα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σωστό. Σε ό,τι αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία και τον ε, συντονισμό, θα σας δώσω την προσωπική μου γνώμη. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Όταν βλέπουμε χρήματα που επενδύονται σε επίπεδο κρατών μελών, ε, στα διαρθρωτικά ταμεία σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, νομίζω ότι ο ενισχυσμένος ενισχυμένο συντονισμό ε, είναι κάτι το ενδιαφέρον. Γιατί δεν θέλουμε προς να αντλήσουμε πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία. Θα ήταν πιο σκόπιμο ε, να προσανατολίσουμε καλύτερα την αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. Και αν αύριο συνολικά έχουμε να κάνουμε με το κεντρικό δίκτυο και το συνολικό δίκτυο και τα κομβικά σημεία, τα urban nodes, ε, τότε μπορούμε να ξαναδούμε την προσέγγιση για να έχουμε μία κοινή ε, προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων. Αυτή θα ήταν μια καλή ιδέα για το μέλλον, σε ό,τι αφορά τον συντονισμό και την αξιοποίηση. Κλείνοντας, να πω ότι Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες σε ορισμένες χώρες δημιουργούν προβλήματα, ιδίως σε χώρες με υψηλό έλλειμμα. Το γνωρίζουμε αυτό και προτείνουμε ότι ίσως θα πρέπει να ληφθεί, αυτό υπόψη, να ληφθεί υπόψη η ευρωπαϊκή υπεραξία για να δώσουμε κάποια ευελιξία. Δεύτερον, στα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται από τα κράτη-μέλη οι ευρωπαϊκοί πόροι πολύ συχνά αξιοποιούνται για χρηματοδοτήσεις που δεν κάνουν όμως τελικά τα κρατημέλη, είτε στο φορά το διάδρομο είτε φορά τη συντήρηση. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις χώρες ε, που δεν έχουν μέσα λόγω ελλείμματος, ισχύει και για άλλες χώρες. Έχουμε ξεκάθαρες αναφορές και εκθέσεις που δείχνουν ε, ακριβώς αυτό το φαινόμενο και για την δημιουργία και για τη συντήρηση υποδομών. Και εδώ δεν είναι μόνο ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να μπει και στην αιρεσιμότητα. Ότι εμεί επενδύουμε και θα πρέπει εσεί παράλληλα να επενδύσετε για τη συντήρηση των υποδομών. Αλλά αυτό είναι η δική μου γνώμη. Ευχαριστούμε πολύ. Να διατηρήσουμε όμω το χρονοδιάγραμμα όσο μπορούμε, γιατί μετά θα πάρουμε χρόνο από του άλλου ε, συντονιστέ. Ο κύριο ε, Κάρελ Βίνκα έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. για να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς υλοποίησης που ρώτησε ο κύριος Βαντερκάμπ, είναι όντω πρόβλημα, αλλά έχει λυθεί από το σχέδιο δράσης. Και τώρα με τα διάφορα κράτη-μέλη εξετάζουμε πώς μπορούμε να συντονίσουμε και να τα ενσωματώσουμε όλα αυτά από κοινού. Για παράδειγμα, στη Γερμανία Μιλούμε για ένα νέο έργο γιατί από γεωγραφική άποψη είναι πολύ σημαντική αυτή η χώρα και συμφωνήσαμε μαζί τους, όχι μόνο με τον Υπουργό Μεταφορών αλλά και οικονομικών, να επενδύσουμε σε 7 διασυνοριακά σημεία ε, διέλευσης που θα ε, υλοποιηθούν μέχρι το 2023. Από αυτή την άποψη καταργούμε τον κατακαιρματισμό μέσω του σχεδίου δράσης. ναι, μπορώ να σας πω ότι ε, είναι ικανοποιητική η συζήτηση αυτή τη στιγμή με τη Γερμανία. Έχει υψηλό βαθμό ψηφιοποίησης η Γερμανία που στηρίζεται από την Deutsche Bahn. Όμως έχουμε πλέον συνεργασία και με την DB, το Υπουργείο και την Επιτροπή που κατά τη γνώμη μου ε, είναι αρκετά καλή συνεργασία. Έχουμε πολλέ συνεδριάσει. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία και τη σχέση μα με το Ηνωμένο Βασίλειο, πρώτα απ' όλα βλέπουμε ακόμα μεγάλο ενδιαφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου ε, στην ανάπτυξη του συστηματό μα, Φαντάζομαι πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό που ανέφερε ο κύριος Βάλλας ε, από πλευρά πολιτική. Όμω δεν υπάρχει λόγο να θεωρήσουμε ότι δεν του ενδιαφέρουν αυτά που κάνουμε. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι δεν πρόκειται εμεί να αλλάξουμε το σύστημά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να υποβάλει συγκεκριμένε απαιτήσει σε καμία περίπτωση. Για το ερώτημα του κυρίου Κράμερ, για το κόστος συντήρησης, όλα αυτά μπαίνουν ε, στο business case, τα λαμβάνουμε υπόψη. Για τα χιλιόμετρα, 4.000 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή και θέλουμε να αναπτύξουμε 7.000 χιλιόμετρα στην περίοδο 18-23. Θα έχουμε λοιπόν 17.000 τότε. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει πλήρης ε, διαφάνεια με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Είναι ιδιαίτερα δραστήριοι και στο σχέδιο δράσης, που είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, γιατί έχουμε πολλά ενδιαφέροντα μέρη, τους κατασκευαστές, τις NSAs, τον κλάδο. Είναι δύσκολο λοιπόν να τα συγκεράσουμε όλα αυτά, αλλά η αέρα διδερματίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί έχει και σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του τέταρτου συνδρομικού πακέτου για το χρονοδιάγραμμα. Αν υπάρχει κάτι που τρέχει για τα 4.000 χιλιόμετρα, όχι προς το παρόν, αλλά έχουμε προβλέψει ότι από το 2019 και μετά παράδοση θα γίνεται με βάση τη χώρα που θα μπορεί να τα τρέξει όλα. Αυτή είναι η συμφωνία με τους παρόχους. Ε, για το άλλο ερώτημα, πράγματι υπάρχει διαφορά μεταξύ παλαιότερων και νεότερων κρατομελών. Τα νεότερα κρατημέλη, κατά μέσο όρο, έχουν πολύ παροχημένες υποδομές. Πρέπει λοιπόν να ανανεώσουμε για τη σήμανση, αλλά πέραν τούτου πρέπει να ανανεώσουμε και όλα, όλες τις υπόλοιπες υποδομές και τον εξοπλισμό. Υπάρχει λοιπόν διαφορά. Και βέβαια το λαμβάνουμε αυτό υπόψη στα προγράμματα. Ο κύριος Ρικέ μας ρώτησε για τις ε, εταιρικές σχέσεις με τον ιδιωτικό κλάδο. Ναι, ξεκινάει τώρα αυτή η διαδικασία. Για παράδειγμα, στι 100 ε, χώρε είχαμε μια τέτοια περίπτωση, όπου οι ιδιωτικοί εταίροι συμμετέχουν στα επενδυτικά προγράμματα. Ιδίω στον τομέα τη διαλειτουργικότητα. Και βεβαίω ε, θα του πιέσουμε γιατί υπάρχουν ε, και business cases που βγάζουν νόημα. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα συνεργαζόμαστε με την γαλλική κυβέρνηση και την SNCF για την σύνδεση Παρίσι-Λιόν. Γιατί χρειάζεται και μια τέταρτη διαδρομή τέτοια σιδηροδρομικών γραμμών. Υπήρχε δυνατότητα να φτιάξουμε νέα συνδρομική γραμμή που θα κόστιζε δύο δις. Όμως, επειδή αυξάνουμε την ικανότητα με το ERTMS δεν χρειάζεται να φτιάξουμε νέα συνδρομική γραμμή. Οπότε τώρα με 500-600 εκατομμύρια καθαρίσαμε. Είναι λοιπόν ε, ένα τέτοιο παράδειγμα που συμφωνώ ότι είναι ακραίο, αλλά αυτό σας δείχνει το πλεονέκτημα που έχουμε. Σε ό,τι αφορά το OBU, πολιτική μας είναι η baseline 3 ε, θα πρέπει να μπορεί να τρέξει οπουδήποτε. Πρώτα θέλουμε οι υποδομές να ε, συμμορφούνται με τις προϋποθέσεις και δεύτερον ο OBU είναι baseline 3 που θα πρέπει να είναι σε θέση να τρέξει παντού με αυτόν τον εξοπλισμό. Συμφωνώ ότι υπήρξε σύγχυση για την baseline 2 και 3. Τώρα η πολιτική είναι ξεκάθαρη. Σε ό,τι αφορά το OBU και τις υποδομές, πιέζουμε για εφαρμογή της baseline 2. Για το OBU απαιτούμε να υπάρχει το baseline 3 για να πηγαίνει οπουδήποτε. Με το baseline 2 δεν γίνεται αυτό. Για το baseline 3 διορθώνει ορισμένα σφάλματα και προσθέτει κάποιες λειτουργίες που δεν υπήρχαν στο 2. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται πλέον baseline 2, αλλά έχουμε λύσει κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ τον κύριο Μην Βλέπω ότι είστε όλοι συνεπαρμένοι με το θέμα που σα απασχολεί. Η κυρία Τροτμάν για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Προσπαθήσω να το σεβαστώ. Πρώτα απ' όλα το θέμα του κύριου Κάμπ για την κινητικότητα ω υπηρεσία. Το ερώτημα που έθεσε είναι το ε, soft κομμάτι σε σχέση με την υποδομή που είναι το πιο σκληρό. Ε, εμείς συμφωνούμε, το ενσωματώνουμε αυτό, είτε μιλάμε για, για τα εναλλακτικά καύσιμα, μιας και έχουμε την υποδομή διανομής, έχουμε την πληροφόρηση και έχουμε και την προσβασιμότητα στην υπηρεσία μετά, που ε, το αλλάζει κάποιες υποδομές όπως τα parking που θα παρέχουν υπηρεσίες πλέον, υπηρεσίες κινητικότητας, όχι μόνο δηλαδή για να μπορέσει κάποιος να παρκάρει το αυτοκίνητό του αλλά και να βρει πληροφορίες, να το ε, φορτώσει, να αγοράσει άλλα μέσα μεταφοράς ή να έχει όλες τις πληροφορίες που, που χρειάζεται στη διάθεσή του. Είναι λοιπόν πολλές οι πτυχές ε, της κινητικότητας ως υπηρεσία. Η διάρθρωση στον βορρά της Ευρώπης ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον βεβαίω συνεχίσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο, θα δούμε. Έω τη Φιλανδία έχουμε τρία project που έχουν αναπτυχθεί για τα LTS και ασχολούμαστε κυρίως με τις υποδομές και τις εφαρμογές και τα σχετικά δεδομένα. Ε, θέσατε το ερώτημα των διαδικασιών που μπλοκάρουν κάποια στιγμή τη διαδικασία και τα, την όλη υπόθεση. Έχουμε πει ότι πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό και πρέπει να εντοπίσουμε όλους τους κανονισμούς εκείνους που παρεμποδίζουν στην πραγματικότητα ε, το να έχουμε μια ε, ροή ε, κανονική των μεταφορών ε, διότι προκύπτει κάποιο κόστος ή κάποιο εμπόδιο. Για, για, το, για τους να πω στον κύριο Κράμερ ότι στον διάδρομο Βαλτική Βόρεια Θάλασσα 70% ε, των πρόσφυγων αφορούν στο σιδηρόδρομο. 2,4 ε, δισεκατομμύρια για 21 project που αφορούν τους σιδηρόδρομους έναντι 450 εκατομμυρίων ε, για τις οδικές μεταφορές. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει προτεραιότητα σε κάποιους διαδρόμους ε, στον τομέα των διαδρόμων για να απαντήσω στον κύριο Ρικέ τώρα. Οι γραμμές ε, οι ρωσικές δεν προβλέπονται η χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά ε, τα project αυτά, τα ευρωπαϊκά. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν ε, κάποια, ε, κάποιος αδύναμος κρίκος ε, ή στην περίπτωση της Φιλανδίας παραδείγματος χάρη όπου η διάσταση είναι η ρωσική διάσταση, η ρωσική απόσταση ό,τι αφορά το, το άνοιγμα των γραμμών. Ε, ε, σε ό,τι αφορά τώρα το Ray Baltica. Ε, κατά πόσο είμαι ικανοποιημένη η κυρία Μάισνερ με την κατάσταση. Και ναι και όχι. Ναι, διότι προχωράει το project. Ε, για να απαντήσω και στον κύριο αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος ε, να μην σεβαστούμε τι προθεσμίες εφόσον ε, ε, υπάρξει διαιώνιση της συζήτηση για την, της συζήτησης για την οργάνωση εφαρμογής. Η τελική απόφαση θα πάρθει τον Ιούλιο φέτος. Έχουμε διαπιστώσει επίσης ότι σε ό,τι αφορά τους διάφορους διαγωνισμούς και τις προσφορές έχουμε καταφέρει να σεβαστούμε τους διαγωνισμούς του ΣΕΦ ε, και αυτό ήταν καλό, ήταν επωφελές για όλους. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να συνεχίσουμε, θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, στην αγορά των ε, οικοπαίδων, των μεταφών, να ολοκληρωθεί επίσης η διαδρομή από τη Λιθουανία έως το πιο νότια ο σχεδιασμός της γραμμής δηλαδή. Ε, πάντως υπάρχει σημαντική πρόοδος σε επίπεδο Πολωνίας κυρίως ε, που ήδη ανέφερε ε, ότι θα προχωρήσει τη διέλευση προς τη Λιθουανία και υπάρχει και η απόφαση μπορεί να πάρθει ακόμα για την τελική, ε, το τελικό σχεδιασμό της γραμμής. Ε, και από λιθωνικής πλευράς και από πολωνικής πλευράς μένουν ακόμα κάποιες μελέτες. Είναι φυσιολογικό αυτό. Τώρα, τι γίνεται με το υδροζέλ, το υδρογόνο ίσως, μεταξύ Βελγίου ή μάλλον στο Μπενελούξ υπάρχει ένα σε πειραματικό στάδιο ε, για μηχανές, το για μηχανές τρένων υδρογόνου, που θα χρησιμοποιούν υδρογόνο, ε, γίνεται μια πειραματική προσπάθεια και σε ό,τι αφορά την μηχανή, αλλά και σε ό,τι αφορά τι δημόσιε μεταφορέ, όπω ε, το τρένο. Ε, δοκιμάζουμε αυτή τη μορφή ενέργεια και τελειώνοντας να πω ότι για του σιδηρόδρομου, και αυτή είναι, ε, είναι κάτι που μας απασχολεί ω συντονιστέ, πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί αλλά θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αλλαγή στην νοοτροπία διότι δεν είμαστε και τόσο αποτελεσματικοί στην πράξη τελικά. Αλλά ε, προχωράμε. Σημειώνεται πρόοδο σιγά σιγά κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα για να τελειώσουμε αυτό το πρώτο κομμάτι, ο κύριο Μπάλα και στι τέσσερα λεπτά έχει, όπω και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ. Ξεκινώ από το ερώτημα του κύριου Ρικέ. Κατά πόσο είμαστε σε επαφή με την ομάδα Μπαρνιέ. Όχι, όχι ακόμα τουλάχιστον. Είμαστε διατεθειμένοι βέβαια. Έχουμε καταγράψει τα προγράμματα και τα έργα στην Αγγλική Επικράτεια. Επιπλέον, τα τελευταία τέσσερα χρόνια ε, έχουμε δει και έχουμε επισκεφθεί ουσιαστικά όλα τα έργα σε όλη την Αγγλική Επικράτεια. Έχω λοιπόν μία γνώση της κατάστασης και γνωρίζω πολύ καλά ότι η DG Move είναι πλήρως προετοιμασμένη. Δεν μπορούμε βέβαια να αρχίσουμε από τώρα να επισερχόμαστε σε τέτοιες ε, λεπτομέρειες. Ε, θέσατε ένα ερώτημα κυρία το οποίο ουσιαστικά αποτελεί ε, την άλλη πλευρά του νομίσματος το πρόβλημα, δηλαδή αυτό της απόστασης από την Ιρλανδία. Ουσιαστικά δηλαδή τώρα ε, με το Brexit θα έχουμε ένα, μια χώρα διέλευσης αν θέλετε των μεταφορών ε, ανάμεσα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εδώ το ερώτημα που θα μας απασχολήσει είναι ε, τα ζητήματα του εκτελονισμού στην, στα σύνορα εκεί, τα νότια σύνορα, αλλά από εκεί και μετά υπάρχει και το ζήτημα της φυσικής διασύνδεσης. Δηλαδή και οι γέφυρες εκεί, οι σύνδεσεις και γενικότερες συνδέσεις με ε, ταξί Δηλαδή και Μεγάλη Βρετανία είναι κάπω καινούργια αυτή η κατάσταση, καινούργιο το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, αλλά υπάρχουν και κάποιες αντίστοιχες ε, ε, περιπτώσεις που είχαμε εντοπίσει στο παρελθόν. Για παράδειγμα, στα Δυτικά Βαλκάνια υπήρχε για παράδειγμα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την Αυστρία και την Ελλάδα. Δηλαδή, για μια τέτοια σύνδεση ο, και σήμερα η, ο άξονα, η σύνδεση διέρχεται από άλλε χώρε. Οπότε η συγκεκριμένη συνδέση θα είναι πολύ σημαντική. Και βέβαια οι επιπτώσεις από τον Brexit θα είναι σημαντικές γιατί αυτή η χώρα συμμετείχε στην, ε, στον ενιαίο χώρο για 40 χρόνια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει ακόμα στη φάση που θα μπορούσαμε να δούμε ακριβώς τι θα συμβεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βαλάς. Έτσι φτάνουμε στο τέλος ε, της πρώτης ενότητας και ευχαριστώ τους ε, συντονιστές γιατί ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και διαδραστική αυτή η συζήτηση και όπως πάντα μας δώσατε πολλές διευκρινήσεις, νέες πληροφορίες ε, και μια ξεκάθαρη εικόνα των όσων ε, συμβαίνουν σε αυτά τα δίκτυα που μας είναι τόσο πολύτιμα. Θα κλείσουμε εδώ λοιπόν το πρώτο πάνελ, να δώσουμε τώρα το λόγο μάλλον να καλέσουμε τους ε, κυρίους Σίμψον και την κυρία Πέις. Θα συνεχίσουμε μετά την συζήτηση και με τον κύριο Βασιβόσκη και τον κύριο Μπαλάς. Πολύ ωραία. Plus à ma place Δίνω πρώτα το λόγο για πέντε λεπτά στον Brian. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ντομινίκ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και πάλι εδώ μαζί σας. Όπως ξέρετε, εκπροσωπώ ε, την οζέοντια προτεραιότητα του ΤΕΝΤΗ θαλάσσιες αρτηρίες, μια πολιτική που είναι πολύ σημαντική για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TNT. Εμείς επικεντρώμαστε κυρίως ε, στην ναυτιλία μικρών αποστάσεων, μια βιομηχανία με ιδιαίτερα διασυνοριακή φύση που συμβάλλει στην βιωσιμότητα στα μεταφορικά δίκτυα, ε, προστατεύει το περιβάλλον και υποστηρίζει και τους συνεργικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, απαιτείται περαιτέρω ψηφιοποίηση. Οι επενδύσει στη συνδεσιμότητα, τι μεταφορέ, την ενέργεια και τι τηλεπικοινωνίε είναι πολύ σημαντικέ. Η ναυτιλία πολύ συχνά αμελείται παρότι, παρόλο το πολύ σημαντικό της ρόλο. Και αυτό με οδηγεί στην πρώτη μου παρατήρηση. Συνέργειες. Στον Στο επόμενο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε ως στόχο την επίτευξη μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα μεταξύ επιμέρου τομέων πολιτική, ε, παράλληλα διασφαλίζοντα ότι οι μεταφορέ παραμένουν στο επίκεντρο επενδύοντας στις καθαρές τεχνολογίες μπορούμε να υποστηρίξουμε πιο αποτελεσματικά και τα δίκτυα TNT και την αυτιλία. Ο τομέας αυτός συμβάλλει ιδιαίτερως ε, στους ε, επιμέρους ευρωπαϊκούς, ευρωπαϊκούς στόχους και για το περιβάλλον και για τα ορυκτά καύσιμα και γενικότερα για την ευρωπαϊκή πολιτική για την κλιματική αλλαγή. Ε, καινοτομία επίσης είναι ένας τομέας με υψηλό κόστος, μεγάλο ρίσκο και δύσκολες συνθήκες και τέλος ψηφιοποίηση, ηλεκτρονικά έγγραφα, ε, διευκόλυνση ε, των ε, διαδικασιών και η ενιαία θηρίδα, όλα αυτά αποτελούν πρότυπα τυποποίηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο πρόγραμμα και έκθεση προόδου θα εκδοθεί από κοινού με τους υπόλοιπους συντονιστές τον, πέρσι τον Απρίλιο σας παρουσίασα τις ε, βασικές προτεραιότητες. Αυτές θα βασιστούμε. Είναι ένα μελλοντοστραφές έγγραφο που θέλει να καλύψει τις μελλοντικές τάσεις και τι είδους ε, θαλάσσιες υπηρεσίες μπορούμε να προσφέρουμε και να υποστηρίξουμε. Τα τέντη εν γέννη και ιδίω ε, στην αυτιλία έχουν να κάνουν με μια σειρά στοιχεία μεταφορών, καινοτομία, έρευνα και ψηφιοποίησης πρέπει να βασιστούμε ε, στην επιτυχία των υφιστάμενων ε, μηχανισμών TNT και να φέρουμε βελτιώσεις για να μεγιστοποιήσουμε την ε, ευρωπαϊκή υπεραξία. Περαιτέρω συνέργειες μεταξύ των TNT και των τομέων διασύνδεσης θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω εξέταση με βάση τη λογική του TNT. Τα περισσότερα έχουν να κάνουν με την ε, παροχή ηλεκτρονικού ρεύματος στις ακτές, ε, μείωση του διοξιδίου ε, του άνθρακα και εξάλληψη των διαφόρων μικροσωματιδίων, νόξ κτλ. Χρειάζεται όμως καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ μεταφορών και ενέργειας γιατί σε επίπεδο λιμένα αυτό συνήθως σημαίνει και εθνικές επενδύσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα εναλλακτικά καύσιμα και την περαιτέρω ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε επενδύσεις σε μεγάλους λιμένες με βάση το φυσικό αέριο, FSRUs, παράλληλα όμως χρηματοδότηση και σε εθνικό επίπεδο. Εδώ μιλούμε για τον απαραίτητο συνδυασμό ε, επενδύσεων μεγάλης κλίμακας ε, στην ενέργεια και ε, εφαρμογών μικρής κλίμακας στις μεταφορές. Όταν μιλούμε για την ψηφιοποίηση, γίνεται πολλής λόγος για την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή ενιαία θηρίδα, μια λύση που έχει δοθεί από τις μεταφορές. Χρειαζόμαστε όμως και ένα σύνολο επενδύσεων για τα ηλεκτρονικά έγγραφα, κάτι το οποίο μπορεί να υποστηρίξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το θεματολόγιο της για την ψηφιοποίηση. Το τελευταίο παράδειγμα της ε, απεξάρτησης από τον άνθρακα με καλύτερη λεπίδρυση μεταξύ μεταφορών και έρευνας ε, είναι εξίσου σημαντικό. Αν περιμένουμε από τον κλάδο να έχει σημαντικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, θα πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και στην ε, ανάπτυξη για τις μη ορυκτές πηγές. Και έτσι αναδεικνύεται η σημασία της συνέργειας μεταξύ ε, έρευνας και μεταφορών. Κυρίε και κύριοι, έχουμε 331 θαλάσσια λιμάνια στο δίκτυο TNT. 408 ε, με μεταφορά εμπορευμάτων και 455 με συστήματα ρορό καθημερινά μεταφέρουν και επιβάτες και εμπορεύματα. Δεν πρέπει να μελήσουμε λοιπόν αυτό το τόσο σημαντικό τομέα και σας παρακαλώ να τον ε, στηρίξετε στα μελλοντικά σας σχέδια. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Monsieur Simpson. Ευχαριστώ τον κύριο Σίμψον. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Πέλς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, είμαι εδώ για να μιλήσω μαζί σας ε, για τον διάδρομο Ρήνο-Δούναβη. Είναι πραγματικά συναρπαστικός ο διάδρομος. Τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι έξι από τα εννέα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στον διάδρομο αυτό, Ρήνο-Δούναβη, λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα θεατρικά ταμεία. Κροατία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Τσεχία, ε, αντιλαμβάνεστε ότι και η Βουλγαρία αντιλαμβάνεστε ότι σε μεγάλο βαθμό ε, βλέπουμε όλες τις προκλήσεις, όλες τις δυνατότητες και όλα τα εμπόδια που μας απασχολούν. Βλέπουμε επίσης και που είναι ε, τα σημεία ε, τα αδύναμα. Και βεβαίως η προσπάθεια που πρέπει να γίνει σε επίπεδο Δούναβη κυρίως, ιστορικά, οι εσωτερικές ναυτικές οδοί συνδέουν τους ανθρώπους, τους πολιτισμούς, τις οικονομίες, ε, θα πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε στον Δούναβη να παίξει με επιτυχία το ρόλο, το κεντρικό ρόλο που του αξίζει. Γνωρίζουμε ότι όταν μιλάμε για το εμπόριο καλύτερα είναι να έχουμε καλούς γείτονες παρά μακρινούς φίλους. Είναι πολύ σημαντικό και ο ρόλος εδώ του, του Δούναβη είναι πολύ σημαντικός. Είναι λοιπόν σημαντικό για μας να αντιμετωπίζουμε συνεχώς τα εμπόδια που υπάρχουν στην αυσιπλοεία. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε οπωσδήποτε τις διοικητικές αλλά και τις επιγραμμικές διαδικασίες. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από την αρχή του προγράμματος ΣΕΦ το 2014. Το ΣΕΦ στο χαρτοφυλάκιο αυτό ε, καλύπτει 24 δράσεις, 382 εκατομμύρια χρηματοδότηση σε τρεις κυρίως τομείς παρέμβασης. Πρώτον, η βελτίωση των υποδομών, δεύτερον οι μελέτες που αφορούν περιβαλλοντικές ανησυχίες και είναι πολλές αυτές και η εφαρμογή σε όλο το Δούναβι του ΡΙΣ. Και βεβαίως έχουμε την εμβληματική ε, πρωτοβουλία έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε ε, τις πτυχές εκείνης του Δούναβι, τις, τις κομμάτια εκείνα του Δούναβι που είναι πιο, πιο ε, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την, την, ε, την αυσιπλοεία σε όλο το μήκος του Δούναβη. Όλοι γνωρίζετε ότι σε περίοδους ξηρασίας δεν μπορεί κανείς ε, να ταξιδέψει στο, σε όλο το Δούναβη Γι' αυτό λοιπόν ο κλάδος, οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν τελικά όσο θα χρειαζόμασταν για να υπάρξει πραγματική χρήση του Δούναβη. Και το καταλαβαίνω, βέβαια και εγώ το ίδιο θα έκανα. Οι πολιτικές, οι πολιτικές από τις εμπλεκόμενες ε, χώρες ε, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την έγκαιρη εφαρμογή των δράσεων του ε, διαδρόμου αυτού. Επίση, δεν πρέπει απλώ να αποδεχόμαστε το project, αλλά θα πρέπει να το οικειοποιούμεθα σε τοπικό επίπεδο. Μετά από μια αργή εκκίνηση βλέπω ότι αυτό γίνεται όλο και πιο συχνά στο δικό μου διάδρομο τουλάχιστον. Από την εκκίνηση της θητείας μου πριν από τέσσερα χρόνια, μιλάω τώρα για τους σιδηρόδρομους, είχαμε απτά αποτελέσματα και μπορέσαμε να καλύψουμε ορισμένα κενά τα οποία ήταν κρίσιμα. Παραδείγματο χάρη, χάρη στο ΣΕΦ και τις 31 δράσεις στους σιδηροδρομούς όπου υπήρξε συνολική στήριξη 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ αυτή τη στιγμή, ευρώ, αυτή τη στιγμή ε, φτάνουμε στα αποτελέσματα που περιμέναμε 246 χιλιόμετρα σιδηροδρόμων δημιουργήθηκαν με ελάχιστες απαιτήσει ε, του TEN-T ε, ηλεκτροδότηση που επιτρέπει περι, περαιτέρω διεύρυνση μεγαλύτερη ταχύτητα 487 εκατομμύρια επίσης οδικών ε, ε, ε, μάλλον δισοδομικών γραμμών θα έχουν πλέον ε, θα είναι εξοπλισμένα με ARS. Ε, στο παρελθόν έγιναν δύο ερωτήματα για την συντήρηση. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα η συντήρηση. Χάρηκα που τέθηκαν τα ερωτήματα αυτά, διότι εγώ πάντα τα θέτω. Ε, στη Ρουμανία βλέπουμε ότι πολλοί, πολλές οδοί έχουν κλείσει. Ε, και αυτό για λόγους συντήρησης. Ε, ένας ιερόδρομος ε, σε μια αστυνομική γραμμή, η οποία δεν συντηρείται, είναι πραγματική καρμανιόλα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου αυτό. Θα πρέπει να το προσέχουμε. Ο κεντρικός μας στόχος είναι να αναπτύξουμε μια βιώσιμη και αποτελεσματική ένα βιώσιμο αποτελεσματικό δίκτυο που να εξασφαλίζει την συνέχεια του δικτύου υποδομών πέρα και από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Οκτώβριο του 2016 ήμουν στη Σερβία και από κοινού την κυρία Μιχαηλόβα ε, την, την ε, ε, Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Μπέκερς, τον Εκκληστικό Διευθυντή της ΕΝΕΑ, ε, ΕΝΕΑ υπογράψαμε λοιπόν μια μια συμφωνία για ένα project με τη Σερβία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πιο σημαντικά προβλήματα συμφόρησης, ε, του Δούναβη ε, στην ε, Σερβία. Είναι ένα και ένα από τα πιο, πιο σημαντικά σημεία διέλευσης συνόρων. Το να διευκολύνουμε λοιπόν την, ε, τις μεταφορές προς τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Αυστρία, την Τσεχία είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η δουλειά. Είναι προφανές ότι ένα σημαντικό σημαντικό προκλήσεις είναι μπροστά μας ε, που ε, παρεμποδίζουν τη μελλοντική εφαρμογή των δράσεων του διαδρόμου. Εγώ είμαι είμαι αισιόδοξη εκφύσεως. Ε, η κάθε πρόκληση είναι μια ευκαιρία για μας και θα ήθελα εδώ στο Νίκο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας μας βοηθήσετε να πετύχουμε τους στόχους μας στις μεταφορές, στις εσωτερικές, στην εσωτερική τα project αυτά διέπονται από περίπλοκη διαδικασία και αυτό διακυβεύει την επιτυχία των project. Τα πρώτα χρόνια του, προγράμματος ΣΕΦ και η εφαρμογή του στο επιτόπου σε ό,τι φορά τις εσωτερικές ε, ε, οδούς αυσυμπλοείας ε, δημιουργήσαμε μια συνεργασία μεταξύ εξόλου των εμπλεκομένων φορέων και των περιβαλλοντικών ομάδων και μηχανισμών όπως το MITID. Εμείς πιστεύουμε ότι η συνέργεια μεταξύ φύσης και ναυσιπλοείας είναι εφικτή το να, το εργάζεται κανείς μαζί με τον ποταμό ε, είναι πολύ πιο σοφό και πολύ πιο αποτελεσματικό και πολλά από τα project του ΣΕΒ προσπαθούν να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ό,τι φορά τη διαχείριση των, του, του, των υδάτων, ε, να μπορούμε να έχουμε σωστή ναυσιπλοεία αλλά σε οικολογικέ συνθήκε. Τα τελευταία δύο σημεία που θέλω να αναφέρω τώρα θεωρώ ότι αποτελούν μέρο του ίδιου τη ίδια πρόκληση. Οι αλλαγέ ε, στην νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών ε, και οι περίπλοκες ε, διαδικασίες χρηματοδότησης ε, καθυστερούν. Καθυστερούν την, την εφαρμογή. Η μελέτη στην Ρουμανία για τους παραδείγματος χάρη θα πρέπει αυτό να ξεπεραστεί και από τα κράτη-μέλη καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου των project. Συμπερασματικά, πολλά project δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για να δημιουργηθεί ένα συνολικό ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών η προσέγγιση είναι όχι μόνο αποτελεσματική από τεχνική πλευρά, αλλά δημιουργεί και μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των χωρών και προωθεί τι ανταλλαγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχει να κάνει αυτό και με ένα αίτημα που αφορά το μέλλον. Εάν στι επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ ε, δεν συνεχίσουμε με του διάδρομου αυτού, όλα αυτά τα χρήματα, και εδώ συμφωνώ με την Κάθριν, ε, θα, έχουν, θα οδηγήσουν σε ένα μοσαϊκό με μπαλώματα και όλα αυτά τα χρήματα που θα έχουμε δαπανίσει ε, θα έχει γίνει αυτό εις μάτιν. Να πω τώρα ότι θα πρέπει ε, όλοι να βασιστούμε στα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει ήδη. Δεν θέλουμε απλώς να κλείσουμε κάποια κενά στο δίκτυο. Θέλουμε πραγματικά να μεγιστοποιήσουμε μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο για τον Ευρωπαίο πολίτη. Κεντρική διαχείριση των κοινωνικών κονδυλίων, ε, μεταρρύθμιση και νέες δυνατότητες ανάπτυξης. Και νομίζω ότι έχω ήδη περάσει το χρόνο που μου αναλογεί. Να πω ακόμα κάτι. Πρέπει να συμπληρώσουμε την προσέγγιση ε, σε ό,τι αφορά τον, τον διάδρομο και σε επίπεδο δημοσιονομικό. Ιδάλλως και πάλι είναι σαν να χάνουμε τα χρήματά μας. Δεν μπορούμε ε, να το πράξουμε αυτό απέναντι στους φορολογούμενους μας. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Πέζ. Βλέπω ότι σα συνεπέρνει αυτό που έχετε να πείτε και όλοι ξεπερνάτε το χρόνο ομιλία. Από εδώ και πέρα όμω θα είμαι αυστηρή. Λυπάμαι για του υπόλοιπου. Ο κύριο Βακοσάφσκι. Σχεδόν το είπα, σχεδόν το πέτυχα. Ευχαριστώ, πολύ κύριε Πρόεδρε. Βόιτσεγόφσκι. Θα σας ε, αποκαλώ με το μικρό από εδώ και πέρα να σας πειράζει. Ξέρω ότι παίρνω το θάρρος, αλλά για να μην, έχουμε, να μην κάνουμε πάλι λάθη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ να μιλήσω γρήγορα και αγγλικά. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με τον ε, πιο σύντομο, αλλά και πιο πολυτροπικό και ανεπτυγμένο άξονα Ρήνου Δούναβη. Πρώτα έχουμε να κάνουμε ζητήματα συμμόρφωσης και θέλουμε να λειτουργούμε με γνώμονα της δράσης. Είπε ο κύριος Βαντερκάμπ ότι πολλές φορές ε, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες. Μπορώ λοιπόν να εξ αρχή να συγχαρώ τους Γερμανούς ε, και τον κύριο Γκρόσε. Ήμουν εκεί όταν αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε με τον Έμερ Χόπερχάουζεν. Υπήρξαν αντιδράσεις από την τοπική κοινότητα για τα υψηλά επίπεδα θορύβου και για λόγους ασφαλείας. Όμως βλέπω ότι το πιο σημαντικό είναι όχι αυτά που είχαμε σχεδιάσει, αλλά αυτά που έχουμε πετύχει. Είχαμε λοιπόν μία σειρά έργα όπως ε, το αεροδρόμιο Μαλπένζα και η συνδρομική διασύνδεση στο τερματικό σταθμό 1 και 2 χρηματοδοτήθηκε από το ΣΕΦ. Ένα πολύ ενδιαφέρον έργο ήταν ε, σύνδεση με το λιμένο στο Ζαλμπρούκεν που αποτέλεσε και έμπνευση για άλλο έργο. Λειτουργούμε λοιπόν με γνώμονα τις ενέργειες. Ε, περίπου 50% ε, σκοπεύουμε να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι το 2020. Είπε ο κύριος Βίνκ 25% για τη RTMS, το κλείδι της επιτυχίας είναι η διακυβέρνηση. Θα ήθελα να το επισημάνω αυτό. Και συνδέουμε και τις δύο προσεγγίσεις από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Έχουμε κατακαιρματισμένη διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτό το συντονισμό των πολιτικών τέντη και διασύνδεσή τους με ξεκάθαρους στόχους γιατί συνεχώς μιλούμε για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Σίγουρα υπάρχει ε, και η δράση των πρωτοπόρων, όπως το τούνελ Γκούταρτ στην Ελβετία και αλλού, που ξεκίνησαν πρώτοι δηλαδή και περιμένουν τους υπόλοιπους ε, να ολοκληρώσουν ε, τους άξονες. Πρέπει λοιπόν να συμβάλλουμε με τις πολιτικές ΣΕΦ και ΤΕΝΤΗ. Γιατί σε αυτό το επίπεδο είναι σωστή η διακυβέρνηση. Βέβαια, σε συνεργασία και με τους βασικούς μας εταίρους, που είναι εξαιρετικά σημαντικοί. Ευχαριστούμε τη CCNR για τη στήριξή τους για την απεξάρτηση από τον άνθρακα και την ψηφιοποίηση των περιφερειακών συστημάτων ε, στα ποτάμια και όλους όσοι ασχολούνται με τα επίπεδα θορύβου, με τα τρένα των 700 μέτρων. Μικρές επενδύσεις μπορούν να μας φέρουν όμως απτά και σχετικά αποδοτικά μέτρα για να έχουμε έτσι μεγαλύτερα τρένα. Μίλησα για την πολυτροπικότητα προηγουμένως. Εύκολα όμως μπορούμε να έχουμε προβλήματα λόγω αυτού του συστήματος. Έχουμε δηλαδή ε, τρόπους μεταφοράς που δεν είναι πάντα πλήρως αξιόπιστοι. Ένα υπόρρευμα λοιπόν το οποίο μεταφέρθηκε όχι στο συνδρομικό δίκτυο αλλά σε φορτηγά. Αυτό ήταν λοιπόν μια ανεπιθύμητη επίπτωση ε, λόγω της ε, έλλειψη αξιοπιστία, Κάτι λοιπόν που δεν πήγε στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Θέλουμε λοιπόν ε, πολυτροπικότητα και σίγουρα ο άξονας Ρήνου Άλπαιων είναι ο πλέον πολυτροπικός. Τέλος, τα όσα είπε και ο κύριος Κράμερ και αν είναι πολύ δύσκολο χωρίς την απαραίτητη στήριξη να περάσουμε από το δικό δίκτυο στο συνδρομικό. Μιλήσατε για τους Ελβετούς και τα υψηλά τέλη που είναι τριπλάσια για τα βαρέα οχήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που τηρήσατε και το χρονικό όριο. Κύριε Σέκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω να σας ε, ενημερώσω και εγώ από την πλευρά μου σε σχέση κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τον δικό ε, και θα βρείτε περισσότερα ε, στοιχεία στο τέταρτο έγγραφο σχέδιο εργασιών το οποίο θα έχει εγκριθεί και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον επόμενο μήνα. Κάποια σημαντικά επιτεύγματα σε ό,τι αφορά λοιπόν τον Ατλαντικό άξονα είναι το άνοιγμα του κομματιού του που είναι του ε, που ε, είναι και το πιο ανεπτυγμένο στον κόσμο και προχωράει με γοργούς ρυθμούς, αλλά και εδώ βέβαια αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα, ειδικότερα στην Ισπανία. Ε, όπου τα πράγματα προχωρούν καλά και στην Πορτογαλία αναμένεται να ξεκινήσουμε στις επόμενες μέρες αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια κενά τα οποία για παράδειγμα ηλεκτροδότησης Καθώ και λιμένες εσωτερική ναυσιπλοεία, τα οποία θα επιληθούν μόνο μέσα στα επόμενα χρόνια. Όμως, οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο επίπεδο πάντοτε του Ατλαντικού άξονα είναι η διαλειτουργικότητα, ειδικότερα στην υπηρετική Χερσόνησο, ε, ένα πρόβλημα το οποίο θα το ξεπεράσουμε σταδιακά, αλλά βέβαια χρήζει και χρόνο και χρηματός ε, το να το επιτύχουμε. Και νομίζω πως εδώ η καλύτερη ιδέα θα ήταν μέσα στο εγγύς μέλλον να προετοιμάσουμε ένα σχέδιο δράσης ως προς το ε, τι ακριβώς θα χρειαστεί από άποψη χρόνου, από άποψη κονδυλίων και ενδεχομένως ε, θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα ξεχωριστό έργο γι' αυτό. Πάντω, σε κάθε περίπτωση η Ισπανία και η Πορτογαλία συνεργάζονται πολύ καλά μέσω και τη διακυβερνητική ομάδα εργασία που έχει ε, συσταθεί, η IG, με την ονομασία ΑΒΕ που έχει συσταθεί για αυτό το σκοπό. Και βέβαια συμμετέχουμε και εμεί σε ένα και προσπαθούμε να δώσουμε όθηση ε, σε αυτήν την συνεργασία που μέχρι τώρα λειτουργεί καλά. Μια άλλη βασική πρόκληση είναι οι διασυνοριακές συνδέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας ε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη στάση της γαλλικής ε, κυβέρνησης μετά από την έκθεση του σε ό,τι αφορά την υποβάθμιση, αν θέλετε, της, ε, των, ε, της προτεραιότητας ορισμένων διασυνοριακών ε, συνδέσεων με την Ισπανία σε ό,τι αφορά τον Ατλαντικό άξονα. Βέβαια θα τηρήσουμε στάση αναμονής για να δούμε ποιες αποφάσεις θα ληφθούν και είμαστε πεπισμένοι και αισιόδοξοι ότι αυτές οι πολύ σημαντικές πτυχές της υλοποίησης του Ατλαντικού άξονα θα ξεπεραστούν, θα επιληθούν καθώς αφορά βέβαια την πολύ καλή εφαρμογή του, του ευρωπαϊκού δικτύου. Τώρα επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάποιες συμπληρωματικές ε, πτυχές. Ε, κατά την πρώτη μου παρέμβαση, ε, την οποία έκανα από κοινού με τον κύριο Μπόντεβεκ, ε, σας περιγράψαμε κάποια από τα βασικά στοιχεία της έκθεσης πρόοδου μας και τώρα θα ήθελα να συμπληρώσω αυτή την έκθεση πρόοδου με κάποια ακόμα στοιχεία. Καταρχήν σε ό,τι αφορά την βελτίωση των σχετικών διαδικασιών, το streamlining. Ε, σίγουρα θα πρέπει να απλουστεύσουμε εδώ τα πράγματα, πράγμα το οποίο βέβαια αποκρισταλώθηκε και από τη συζήτηση που έγινε σήμερα εδώ και μια σχετική μελέτη σε ό,τι αφορά το streamlining, ε, έγινε το 2015 και θα υποβληθεί και μια νομοθετική πρόταση μέσα στο Μάιο, ελπίζουμε πως θα στεφτεί με επιτυχία. Δεν θα επανέλθω στο ζήτημα των καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς το λόγο ζήτημα έχει συζητηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά τα όσα θα συμβούν μέσα στα επόμενα χρόνια και ειδικότερα στο πλαίσιο του επόμενου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου σε ό,τι αφορά το μηχανισμό ε, συνδέοντα την Ευρώπη. Και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τα κονδύλια, αλλά αφορά και την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών, όπω αναφέρθηκε από όλους μας εδώ στην αίθουσα σήμερα. Και άλλα στοιχεία, όπω για παράδειγμα η ενίσχυση του ρόλου των συντονιστών, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην καλύτερη επιλογή των σχετικών έργων και αυτό με τη σειρά του ε, σε καλύτερα σχέδια εργασιών σε ό,τι αφορά του επιμέλου αξιών. Ε, Επίση, θα πρέπει να επιμείνουμε στην ποιότητα ε, των έργων και όσο περισσότερα ιδιωτικά κονδύλια, ιδιωτική χρηματοδότηση ε, ε, ε, υπάρχει σε ένα έργο, θα πρέπει να έχουμε και περισσότερε αναλύσει, όχι μόνο δεσμότητα, αλλά σε ό,τι αφορά αυτά τα έργα. Τώρα, σε ό,τι αφορά του υφιστάμενου κανόνε, Ε, εδώ ε, θα πρέπει να έχουμε μια ε, συνολική προσέγγιση καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί σημαντική διάσταση της πλήρους εφαρμογής των, των, των αξώνων και εδώ βέβαια εδώ αναφέρομαι και στο ζήτημα της ε, ενδιαφέροντος και τα blending calls αλλά από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αναφέρθηκαν όπως αυτά της διαλειτουργικότητας, του ERTMS και όσα τέθηκαν σήμερα εδώ. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε πολύ στοχευμένοι σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητές μας, ειδικότερα σε ένα περιβάλλον όπου ε, υπάρχει περικοπή των, της χρηματοδότησης. Το λόγο ο κύριος Βόντικ τώρα για πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Will es ε, etwas weil. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι που αναφέρθηκα μία σειρά από ναι. θέματα και βέβαια με τη σειρά μου χαίρομαι που μπορώ να, να αναφερθώ στο ζήτημα της ε, σύνδεσης ε, του όλων των χωρών της Βαλτικής και της ε, Πολωνίας με, την, μέχρι τα λιμάνια της Ιταλίας. Εδώ το ζητούμενο είναι ή μάλλον αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι όχι μόνο αναλύσαμε σωστά την ε, κατάσταση, αλλά πραγματικά βλέπουμε καλή πρόοδο σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις ε, σιδηροδρόμους και την ηλεκτροδότηση εδώ. ουσιαστικά ε, ήδη ο ε, άξονας πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του TNTS, TNT. σε ό,τι αφορά το ERTMS τώρα χρειαζόμαστε εδώ περισσότερες επενδύσεις Ειδικότερα στην Πολωνία και στη Σλοβενία εδώ χρειάζονται περισσότερε επενδύσει γιατί υπάρχουν ελλείψει, αλλά αυτέ οι χώρε ήδη κάνουν κάποιε προσπάθειε. Τώρα, οι δικέ μου ε, προποθέσει ε, πρέπει να πούμε ότι έχουν συμπεριληφθεί μέσα και στα εθνικά σχέδια δράση. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα ίδια κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί σε ό,τι αφορά την επένδυση 35 δισεκατομμυρίων ευρώ με βάση ακριβώ αυτό το συντονισμό που έχει γίνει. Δηλαδή από τα 70 δισεκατομμύρια συνολικά τα 50 ήδη είναι ε, δεσμευμένα, οπότε κάτι τέτοιο αποτελεί ε, επιτυχία. Και ε, εδώ πράγματι η διακυβέρνηση σε ό,τι αφορά τον άξονα πέτυχε, γιατί έχουμε για παράδειγμα διοργάνωση τακτικών φόρα, τα οποία λαμβάνουν χώρα με όλους τους συναρμόδιους φορείς και η συζήτηση εκεί που γίνεται σε κλίμα εμπιστοσύνης. Υπάρχουν και ειδικέ ομάδες εργασίας σε ό,τι αφορά τις, τους λιμένες, του τερματικού σταθμούς εμπορευμάτων και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσεγγίζουμε τα επιμέρους θέματα πολύ εξειδικευμένα και σε ό,τι αφορά τα 8 σημαντικά διασυνοριακά ε, σημεία στα οποία αντιμετωπίζαμε μεγάλε δυσκολίε, έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε πολύ σαφεί ε, συμφωνίε μεταξύ των κρατών μελών, διμερεί και τρίμερει συμφωνίε, πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία πράγματι μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ ε, από το ΣΕΦ έχουν ειστρέψει σε αυτόν τον ευρωπαϊκό άξονα, πράγμα το οποίο καθιστά και αυτό με τη σειρά του σαφές ότι ε, υπάρχουν επιτυχίες οι οποίες σημειώνονται με αυτές τις ε, επενδύσεις. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε στις στα σημεία τα συνοριακά στα οποία υπάρχουν ελλείψει. Για παράδειγμα, η Αυστρία επενδύει ιδιαίτερα εδώ στο Ζέμερν και εδώ θα συμφωνήσω με του άνθρωπου ότι δηλαδή συχνά τα όσα επενδύουμε στην υποδομή χάνονται γιατί ακριβώς δεν υπάρχει καλή διασύνδεση διασυνοριακά και ακριβώς ε, ε, η καλή σύνδεση με τον ε, εμπορματικό άξονα 5 είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά και για τα υπόλοιπα σημεία εδώ υπάρχουν δηλαδή ε, σημαντικά έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ακόμα οριμάσει αρκετά. Για παράδειγμα δεν έχουν ε, ληφθεί ακόμα οι κατάλληλε κατασκευαστικέ άδειε, δεν έχουν γίνει οι κατάλληλε μελέτε για τι περιβαλλοντικέ επιπτώσει και ούτω καθεξής. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ λίγο στην αποτελεσματικότητα του μηχανισμού ΣΕΦΕ. Αν εξετάσουμε αυτόν τον ε, άξονα, στο blending call καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 300 εκατομμύρια ευρώ, τι σημαίνει αυτό, ότι οι χώρες ε, ε, της, ε, του προγράμματος συνοχής εποφελούνται και αξιοποιούν αυτέ τι δυνατότητες, οπότε αυτό αφορά και τη συζήτηση που κάναμε στο παρελθόν. Και το είπα αυτό και στο ε, ε, παρελθόν. Εάν έχουμε ε, απορρόφηση της άξης του 97% και εάν τα 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ του τμήματος για την πολιτική συνοχή έχουν απορροφηθεί στο σύνολό τους, αυτό αποτελεί πραγματικά επιτυχία, πραγματική επιτυχία. Και σε αυτό το πλαίσιο βέβαια η επίτευξη των στόχων των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από το πώς θα δημορφωθεί το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διακοπεί αυτή η πρόοδος που έχει επιτευχθεί ε, με το επόμενο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω πως το ε, ΣΕΦ κατέδειξε ακριβώς ότι μπορούμε να επιτύχουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μέσω της συντονισμού των επιμέρους δικτύων και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτή την έννοια στο κόνσεπτ του, του του άξονα και νομίζω πως από εκεί και μετά θα πρέπει να θέσουμε και κάποιες ορισμένες αρχές ε, όπως για παράδειγμα το use it or lose it, δηλαδή αξιοποίησέ το ή ε, δεν θα το, μπορείς να το αξιοποιήσεις περαιτέρω. Ε, γιατί αυτοί, αυτές οι προσπάθειες είναι προσπάθειες από κοινού. και βέβαια στο πλαίσιο της αξιοποίησης του άξονα, μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ήδη ότι ναι, ήδη άξιζε τον κόπο, αλλά και σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις συνεχίζουμε και τις εργασίες μας προκειμένου να τις διορθώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπάλας και στον κύριο Βοσισόφσκι. Εξ ονόματος των δύο συναδέλφων που δεν μπορούσαν να είναι εδώ σήμερα, έχετε λοιπόν το λόγο για πέντε λεπτά έκαστο. Ο Πάκος δεν είναι εδώ. Θα τον εκπροσωπήσω λοιπόν. Στα αγγλικά βεβαίως. Τώρα, για τον μεγαλύτερο άξονα. Γιατί ο προηγούμενος είναι, ήταν ο μικρότερος που ανέφερα. Ο άξονας Σκανδιναβίας ε, Μεσογείου λοιπόν καλύπτει 9, πάνω από 9.000 ε, χιλιόμετρα συνδεδομικού δικτύου. Είναι τριπλάσιος λοιπόν από τον άλλον. Δεν είναι ο ο άξονας με το μεγαλύτερο φόρτο, αλλά είναι ο μεγαλύτερος. Έχουμε ακολουθήσει ε, τους ε, στόχους με βάση τους κανονισμούς TNT. Ε, Θέλουμε να περάσουμε σε μεγαλύτερα τρένα των 740 μέτρων, με καθαρά καύσιμα και με άλλες παραμέτρους. Διαφορετικός άξονας λοιπόν, αλλά με τις ίδιες προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση κύριος Φόλξ ε, μιλάει για τον ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση και εισάγει καινοτόμα στοιχεία των ε, εργαστηρίων. Τέσσερα τέτοια εργαστήρια ακολούθησαν μια ιδιαίτερη προσέγγιση διαχείρισης μεταξύ ομοτήμων και επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα στοιχεία του άξονα. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι τα έργα. Έχουμε δύο μεγάλα διασυνοριακά έργα. Planner Πέισταλ προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027. Αν ολοκληρωθεί θα είναι 5 χιλιόμετρα μεγαλύτερο από το τούνελ Γκόταρτ, που αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο σειροδρομικό τούνελ στον κόσμο. Μπορεί λοιπόν τότε αυτό να γίνει το μεγαλύτερο τούνελ στον κόσμο. Σέρμαν Μπέλτ είναι η δεύτερη σύνδεση και ήδη έχει προχωρήσει αυτό το έργο από τη Δανία. Τίθεται βέβαια και ζήτημα πρόσβασης στη Γερμανία. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2028. Στο μέλλον πολύ σημαντικά στοιχεία είναι η διαλειτουργικότητα, ψηφιοποίηση, απεξάρτηση από τον άνθρακα και εναλλακτικά κάψιμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριε Μπαλάς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Τώρα, εκπροσωπώ τον συνάδελφο Λορενσιάν Μπριγχόρστ, συντονιστής για τον άξονα της Μεσογείου. Μου ζήτησε να πω μερικά λόγια για κάποια βασικά επιτεύγματα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την Κόπερ, αυτή την, αυτόν τον άξονα στη Σλοβενία, που ολοκληρώθηκε το 2016 και έτσι διασφαλίζεται η σύνδεση με τον ασιατικό λιμένα μετά πρόσβαση από το Μιλάνο Μαπένσα και επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου από τον τερματικό σταθμό 1 προς τον τερματικό σταθμό 2. Όλοι γνωρίζουν το πιο σημαντικό εγχείρημα είναι η σύνδεση, η συνδρομική σύνδεση Λιών-Τωρίνου που θα είναι η πρώτη συνδρομική ε, σύνδεση μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, νότια των Άλπαιων με μήκος 58 χιλιόμετρων. Υπάρχει ευρεία στήριξη και από τις δύο πλευρές και από την γαλλική και την ιταλική κυβέρνηση και η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται σε 10 χρόνια από τώρα, 2028. Υπάρχουν ε, και άλλες ευκαιρίες και δυνατότητες, σύνδεση λιών με άλλε πόλεις ε, που θα μπορέσουν να αποφορτήσουν τα δικά δίκτυα, αύξηση της ικανότητας ε, του συνδρομικού δικτύου Τη Λιών που θα μείωνε την κίνηση μεταξύ Μασαλίας και Ισπανίας, μετά αύξηση της ικανότητα στο Βλέσσα Βερόνα Βενετία, σε αυτή τη συνδρομική γραμμή. Προκλήσεις υπάρχουν στην μετάβαση από το Iberia στο UIC και στα σχετικά πρότυπα, η RTM, στη συνδέση και με την ε, Γαλλία και με τη Σλοβενία. Τέλος, ε, η διασυνοριακή σύνδεση μεταξύ Φιγκέρες και Περπινιό θα πρέπει να συνεχιστεί σαν προσπάθεια. Βλέπετε στη διαφάνεια τις προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. χωρί να χάσουμε περαιτέρω χρόνο, να δώσουμε το λόγο στα μέλη μα Σε ένα δεύτερο κύριο τραπέζι για τρία λεπτά. Ο κύριο Βιμ Βαντερκάμπ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην πρόκληση, πρόσκληση είδα ότι ο Μπράιαν Σίμψον τώρα είναι συντονιστής σε ό,τι αφορά τις ε, θαλάσσιες αρτηρίες και τη βιωσιμότητα. Είναι νέος τίτλος ή είναι ένας τίτλος τιμής. Τι συμβαίνει. Και συνεχίζω στα Ολλανδικά τώρα. Πρόεδρε, υπάρχει δρεμία κριτική ως προς το Single Maritime Window, την ενιαία θαλάσσια θηρίδα, το οποίο έχει είναι στάσιμο, έχει κολλήσει, είναι κρίμα, ίσως και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να μας πει τώρα ο Μπράιαν πώς βλέπει τα πράγματα από εδώ και πέρα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το κινήσει εκ νέου. Θα πρέπει σε αυτό να εμπλακεί και ο σχετικός συντονιστή για τις θαλάσσιες αρτηρίες. Πώς ρυθμίζεται. Και τέλος, ένα τρίτο ερώτημα προς τον Μπράιαν ε, αν έχει επαφές με τον ε, Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ΑΕΜΟ, που είναι στο Λονδίνο, που διαρματίζει πολύ σημαντικό ρόλο ε, στην ναυτιλία. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει κατά πόσο βρίσκεται σε επαφή με τον IMO και αν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Τώρα, στην κυρία Πέις, ε, δηλώνω κάθετα αντίθετος στο ότι η συντήρηση θα αποτελέσει τμήμα των αξώνων TNT. Τα κράτη-μέλη έχουν αρμοδιότητα, ευθύνη. Και αν δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη της συντήρησης, δεν τους αξίζει άξονας, για να το πω ξεκάθαρα. Με μία και μοναδική εξαίρεση. Για το Δούναβι. Ε, που θεωρούμε ότι είναι μία επένδυση. Και, θεωρού, και θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Πείς κατά πόσο όλοι συμφωνούν με αυτό το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, εταιρικέ σε γειτονικέ χώρε. Ο συνάδελφος Τέλη έφυγε, αλλά μιλήσαμε για ένα βράδυ κάποια στιγμή και οι γεωπολιτικές ε, σχέσεις με τις γειτονικές χώρες είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο και δεν ξέρω πώς ε, λαμβάνουμε υπόψη αυτή τη τυχή της κινητικότητας των μεταφορών και των γειτονικών χωρών. Πώς από γεωπολιτική άψη μπορούμε να το πλασάρουμε καλύτερα. Γιατί όλοι ξέρουμε τι κάνουν οι φίλοι μας ε, στη Ρωσία με τρένα που πηγαίνουν στα σύνορα. Ίσως θα μπορούσε η κυρία Πέση να, τα, να το αναλύσει περαιτέρω. Τέλος προς τον κύριο Παβέλ. Υπάρχουν μεταφορείς που δεν πληρώνουν το τούνελ Γκοτάρ και με το σχετικό τίμημα των 323 ευρώ και έτσι ε, περνάνε μέσα από την Ελβετία. Πώς θα το λύσετε σε αυτό. Ήσασταν και εσείς τότε σε αυτή την ε, συνεδρίαση με τους Ελβετούς Πρέπει να προσέξουμε. Γιατί απλά δεν παίρνουν το τούνελ Γκοτάρ και το Μπρένερ. Μάλλον παίρνει πολύ χρόνο το να μπει ένα φορτηγό στο σιδηρόδρομο. Ιδίω αν οι οδοί πρόσβαση προς το τούνελ δεν είναι έτοιμες. Τώρα προς τους κυρίους Μπόντεβιχ και Σέκη. Στην παρουσίασή σας είπατε ότι η γαλλική κυβέρνηση δεν θεωρεί ποια προτεραιότητα τα διασανοριακά έργα. Θέλει να τα υποβαθμίσει δηλαδή. Αυτό ίσχυε μόνο υπό τον Ολάντ ή και τώρα με τον Μακρόν. Γιατί είναι μάλλον ε, δυσάρεστη και αρνητική εξέλιξη. Κάτι που θα θέλω να επισημάνω, κύριε Πρόεδρε. η νοοτροπία ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό που μας προσφέρει αυτή τη στιγμή το ΣΕΦ είναι πολύ παθητική. Ο Έτιγκερ λέει ε, πολυαιρεσιμότητα και προσθέμενη αξία. Το ΣΕΦ αυτό ακριβώς καταδεικνύει. Είναι παράδειγμα προς από αυτή την άποψη. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν όχι να διπλασιάσουν τα χρήματα, τουλάχιστον να τα αυξήσουν του ΣΕΦ. Κάτι ακόμα προς τον κύριο Παβέλ για την, ε, για την σύραγγα Φέιμανα γιατί πρόκειται για ε, συγκεκριμένες περιοχές της Βόρειας Γερμανίας που μπλοκάρονται τον μπλοκάρουν. Και ο κύριος Κράμερ, ή μάλλον οι πράσινοι, συγγνώμη, ε, στη Γερμανία είναι αυτοί που μπλοκάρουν αυτό το ζήτημα και θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Κράμερ που έχει καλή σχέση με τους ε, εκεί να το προχωρήσει. Γιατί θα έρθουν και οι δικαστικέ ε, υποθέσεις και εκεί οι πράσινοι έχουν ε, τριπλάσιο, τριπλάσια ατζέντα και θα πρέπει ο κύριος Κράμερ να αναλάβει δράση. Ευχαριστώ τον Βιμ Βάντεν. Κάποια ερωτήσει, παρότι βεβαίω δεν σεβαστήκατε, σεβαστήκατε το χρόνο ομιλία σα. Ζητώ συγγνώμη. Εντάξει, για μια φορά δεν πειράζει. Ο κύριος Ερτούγκ έχει το λόγο. Ναι, καταρχήν ευχαριστώ για όλες τις παρουσιάσεις. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Μπράιαν πρώτα. Πριν από δύο εβδομάδες ήμασταν στη Σικελία, στην Κατάνια, με την Επιτροπή Μεταφορών και μιλήσαμε με τους, με τους τοπικούς εκπροσώπους και ήταν κάπως ε, έτσι στενοχωρημένοι με την οικονομική κατάσταση στο τεφορετικό του τους ε, λιμάνι ιδιαιτέρως και παραπονέθηκαν κάπως για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εγώ προσπάθησα να τους εξηγήσω πώς ε, θα λειτουργήσουν τα πράγματα και τις προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από πάνω προς τα κάτω. Υπάρχει κάποιο καλό νέο για το λιμάνι της Κατάνια. Είναι μια απόφαση που έχει παρθεί, που μάλλον θα πρέπει να παρθεί από την κυβέρνηση. Και κάτι άλλο τώρα για τον ε, κύριο Μπόντεβιτς. Χαίρομαι που είσαι μαζί μας ε, Κούρτ εδώ και σας ξαναβλέπω. Ε, δύο ερωτήματα θα ήθελα να θέσω. Βασικά μία παρατήρηση και ένα ερώτημα. Καταρχήν σε ό,τι αφορά αυτό που, μόλις, που είπε μόλις τώρα ο συνάδελφος Βίμ Κάμπο, ότι η γαλλική δηλαδή κυβέρνηση προσπάθησε να υποβαθμίσει την προτεραιότητα αυτής της πτυχής. Ότι, δηλαδή σε κάθε περίπτωση δεν θέλει να εστιάσει ε, στις διασυνοριακές ε, περιοχές. Πράγματι ισχύει αυτό. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δοθεί μια απάντηση από την πλευρά της. Και αν πράγματι ισχύει, τότε, και πρόκειται για ένα στρατηγικό ζήτημα, ε, τότε και ακόμα και μετά από πέντε χρόνια θα πρέπει να πούμε ότι ήδη τα όσα επέτυχε εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, σε αυτά, σε τα αντιευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Οπότε μέσα στην επόμενη 7 ετή περίοδο μήπως θα έπρεπε να μεταβιβάσουμε λίγο τις αρμοδιότητες σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Γιατί από τότε που συμμετέχω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, αυτό που ακούω ξανά και ξανά είναι ότι όταν αλλάζει μια εθνική κυβέρνηση, οι προτεραιότητες της αλλάζουν και έτσι κάποιες επενδύσεις οι οποίες έτρεχαν καλά μέχρι τότε ξαφνικά θεωρούνται από τη νέα κυβέρνηση ως ε, όχι ιδιαίτερα χρήσιμες. Τώρα, εγώ δεν είμαι βέβαια νομικός, οπότε δεν γνωρίζω κατά πόσο ε, θα ήταν απαραίτητη μια τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων. Πάντως, αν είναι κάτι τέτοιο δυνατό, σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να απευθύνω μια τέτοια ε, έκκληση, ούτω ώστε δηλαδή τα όσα αποφασίζουν οι κυβερνήσεις να είναι πάκτα sunt σερβάντα. Δηλαδή, οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει πράγματι να ε, πληρούνται από την πλευρά του ασχέτως ποια κυβέρνηση αναλαμβάνει. Τώρα, το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να θίξω. Όταν είχαμε ξεκινήσει ξεκινήσει την ε, διαδικασία αυτή πριν 6-7 χρόνια, οι προποθέσει ήταν τελείω διαφορετικέ, το πλαίσιο ήταν τελείω διαφορετικό. Ε, για παράδειγμα, μέχρι, ε, στο ενδιάμεσο διάστημα υπήρξαν δύο νομοθεσίε σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Έχουμε την Κίνα ω ένα πολύ μεγάλο παίκτη σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ηλεκτροκίνητη ε, κινητικότητα. Έχουμε το ζήτημα των υποδομών σε ό,τι αφορά τη μείωση των υπομπών άνθρακα στι ε, ε, μεταφορέ. Και κατά συνέπεια, κατά τη δική μου άποψη, τα core networks, αυτή, τα βασικά δίκτυα θα πρέπει να συνοδευτούν από υποχρεωτική δημιουργία των σχετικών υποδομών έτσι ώστε να μπορέσουμε πράγματι να επιτύχουμε αυτή την τη μετάβαση αν θέλετε στην ε, ηλεκτροδότηση στην ηλεκτροκίνηση. Ε, εντάξει τώρα δεν ξέρω κατά πόσο Κούρτε είσαι ο αρμόδιος ε, για να θέσω αυτό το ερώτημα αν δεν είσαι ας το απαντήσει όποιος είναι είναι αρμόδιος. Ευχαριστώ τον κύριο Χέρτογκ. Σεβαστήκατε και το χρονικό όριο. Κυρία Μέσνερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο ε, ε, πειθαρχημένη, όπως ο Ερτογ. Θα ξεκινήσω αμέσως, συγγνώμη, Βιμ, εσύ δεν σε βάσκες το χρόνο. Τώρα μου παίρνεις και το δικό μου, λοιπόν, προς τον Μπράιαν το πρώτο ερώτημα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Αναφέρθηκε στο, ε, στην ενιαία θηρίδα. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι αλήθεια ότι τα λιμάνια που χρησιμοποιούν την ενιαία θηρίδα τελικά δουλεύουν διπλά και αυτό τελικά είναι μειονέκτημα, κάτι που θα ήταν αρνητικό βεβαίως. Υπάρχουν χρήματα ε, που να έχουν διατεθεί για τις ε, υποδομές υποδοχή στα λιμάνια. Προς την κυρία Πέις τώρα. Η συντήρηση είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν πολύ καλά οι υπεύθυνοι για, τους, για τις θαλάσσιες οδούς. Γίνεται κάτι προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης για το πολυτροπικό, τις πολυτροπικές μεταφορές ε, υπάρχουν επενδύσεις. Είναι το έτος της πολυτροπικότητας ε, υποτίθεται φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Βοτσικόφσκι, αναφερθήκατε, εδώ είστε ναι, αναφερθήκατε στον πιο πολυτροπικό ε, το πιο, στο πιο πολυτροπικό διάδρομο. Θα ήθελα να μου πείτε κάτι περισσότερο από αυτό. Αναφερθήκατε στο πέρασμα στους σειρόδρομους. Ε, γιατί να μην έχουμε και πέρασμα προς τις ε, θαλάσσιες, θαλάσσιες, ε, εσωτερικές εφόσον υπάρχει δυνατότητα. Κύριε Σέκη, για τη Βόρεια Ισπανία και τη Γαλλία είναι δύσκολο αυτό το σημείο διέλευση. Έχουμε πάει και σχετική αποστολή, προβλέπεται κάποια βελτίωση εκεί επίσης ε, καινοτόμος χρηματοδότηση. Πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό αυτό. Πιλωτικά προγράμματα ή κάποια ε, ομόλογα για project δεν έχουν καταφέρει, καταφέρει να τα χρησιμοποιήσουμε στα πλαίσια του ΣΕΦ. Ξέρετε κάτι από αυτού. Κύριε Μπούντεβιγκ, δύο ερωτήματα. Ε, διασυνοριακή διάσταση. Μας είπατε πως θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερα την περιφερειακή επιτυχή. Τι σημαίνει αυτό. Ότι δηλαδή θα πρέπει να στοχεύσουμε στην κοινή χρηματοδότηση των δύο περιοχών που βρίσκονται σε αυτή τη διασυνοριακή ε, σύνδεση ή κάτι άλλο. Και βέβαια εδώ υπάρχουν μια σειρά από διαφορετικές ε, πλατφόρμες. Ε, τώρα σε ό,τι αφορά τον μεσογειακό σκανδιναβικό άξονα, εδώ αναφέρομαι στην επίσκεψη που είχαμε στην Σιθιλία και εδώ το ανέφερε και ο Ισμαήλ ότι ε, σε ορισμένε περιπτώσει δεν ε, αξιώνονται τα απαραίτητα έργα στην Σικηλία. Ε, δηλαδή ενδεχομένω η εστιάζει υπερβολικά στα επιρωτικά και όχι στην, στην Και μετά σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη γέφυρα με τη Μεσίνα. Πράγματι θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Όλοι πάντω οι κάτοικοι τη Σικυλία το επιθυμούν. Ευχαριστώ την κυρία Μάισνερ. Σεβαστήκατε και το χρόνο ομιλία σα, βλέπω κι εσεί, αντίθετα με κάποιου άλλου. Ο κύριος Κράμερ. Και για αυτές τις παρεμβάσεις θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για μία ακόμα φορά. Καταρχήν σε ό,τι αφορά την αυσιπλοεία. Δεν χρειαζόμαστε κανένα είδου τεχνολογικέ κοινοτομίε. Το βαρύ πετρέλαιο, το αργό πετρέλαιο. Αυτά στο 0,1% παρόλα αυτά παραμένει 500 φορές πιο ε, βλαβερό ε, και πιο μολυσματικό από ότι το δίζελ. Οπότε, αν πούμε ότι εστιάσουμε περισσότερο στον δίζελ, δεν χρειαζόμαστε κανένα είδου τεχνολογική καινοτομία. Γιατί δεν το κάνουμε λοιπόν. Ουσιαστικά δηλαδή το ντίζελ αποτελεί ένα προϊόν της, ε, της ε, ε, του πετρελαίου, οπότε γιατί δεν το επιτυχάνουμε. Όταν κανείς δεν αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο, πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορούμε να επιλύσουμε το ζήτημα. Θα παραμείνει πάντοτε εξαιρετικά ρηπαρή η ναυσιπλοεία και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αντιφάσκουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί λοιπόν δεν γίνεται κάτι σε ό,τι αφορά το ντίζελ. Τώρα αναφέρομαι στα μεγάλα έργα ειδικότερα των διάνοιξης των τούνελ. Για παράδειγμα, έχω ξαναπεί επανειλημμένα, για 100 εκατομμύρια θα είχαμε τη σύνδεση μεταξύ Μπρέσλαου και ε, ε αλλά ε, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Ε, Ποιε είναι οι εμπειρίες που, είχαμε. Ε, για παράδειγμα, η σύμβαση για το τούνελ που ολοκληρώθηκε πριν από 21 χρόνια τρέχει. Ενώ στην Ιταλία δεν συμβαίνει τίποτα ή για παράδειγμα στο το τούνελ ε, ε, ε, Μπρένα Βασιλεία. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει. Βελονίνο Μόναχο 20 χρόνια χρειάστηκαν δύο ώρες συντομεύθηκε η σχετική απόσταση και σε ό,τι αφορά το νέο τούνελ Γκόταρτ ουσιαστικά πάρα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Οπότε Α ε, ας με ρωτήσει κανείς το τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά τις σχετικέ συνδέσεις από αυτά με τη Γερμανία. Ε, κανείς δεν ενδιαφέρεται, δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι θέλουν απλά να φτιαχτεί ένα τούνελ και από εκεί και μετά δεν τους νοιάζει τι άλλο θα γίνει. Δεν θα πρέπει εδώ να είχαμε μια πολυτροπική ε, μεταφορά. Δηλαδή ένα μικρό κομμάτι για παράδειγμα να γίνεται ε, ε, με ε, πλωτά και από εκεί και μετά όλο το υπόλοιπο οδικά. Απλά κανένα δεν ενδιαφέρει το κάτι τέτοιο. Ε, για παράδειγμα την ε, Ιταλία, ναι, τη γέφυρα με τη Μεσένα και ούτω καθεξής, ναι. Αλλά επαναλαμβάνω σε ό,τι αφορά το τούνελ Γκόταρ, μέχρι την δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα είδου σύνδεση γιατί δεν δίνω τα κατάλληλα κονδύλια. Μα δεν είναι τρελό κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν τα μεγάλα project είναι εκείνα τα οποία πραγματικά μα ενδιαφέρουν. Ναι, όλοι λένε χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια. Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια, δεν πρόκειται να τα λάβουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει ε, ε, να αποφασίσουμε ενδεχομένω να μην φτιάξουμε ένα από αυτά τα τούνελ που θέλουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε τι συνδέσει που λείπουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν και εδώ απευθύνομαι και στην Επιτροπή. Μήπω θα πρέπει να ασκήσει πιέσει στα κράτη-μέλη ε, Βερολίνο Μόναχο για παράδειγμα. 500 εκατομμύρια ευρώ έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά η σύνδεση στο σύνολό τη δεν έχει επιτευχθεί. Άρα λοιπόν πολλέ φορέ αυτό που τελικά που συμβαίνει είναι τα κράτη-μέλη εστιάζουν μειοπικά, αν θέλετε, στα δικά του εθνικά συμφέροντα και σε τίποτα άλλο. Άρα, ποιο θα πρέπει να έχει τη γενική συνοπτική εικόνα, η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει αυτό το ρόλο αναφέρθηκε αυτό και από τον συνάδελφο το Μενέξη ό,τι αφορά τα 800 μέτρα και ούτω καθεξής. Ναι, εντάξει, θα μπορούσαμε να συντομεύσουμε την απόσταση κατά μία ώρα. Αλλά όλα αυτά δεν τα επιτυχάνουμε εδώ και 25 χρόνια ακριβώ δεν επιτυχάνεται ε, κάτι τέτοιο. Και για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το τούνελ Γκοτάρ, σα ξαναλέω, ε, το τούνελ ολοκληρώθηκε, αλλά οι συνδέσει προ το τούνελ ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Άρα τι, τι κάνουμε τελικά, δεν κάνουμε τίποτα. Ίσως ε, λοιπόν ε, θα έπρεπε να επιμείνει, συνάδελφε Κούρτο, ότι οι συνδέσει, για παράδειγμα, με αυτά τα μεγάλα έργα, με αυτά τα τούνελ θα πρέπει να διασφαλιστούν. Ε, γιατί αποτελεί ντροπή αυτό για τη Γερμανία, αποτελεί ντροπή για την Ιταλία, αλλά κανένα δεν λέει τίποτα και ε, προσποιούμαστε όλοι ότι όλα λειτουργούν καλά. Και θα ήθελα να ακούσω και μια αντίδραση από του συναδέλφου. Ποια είναι η στάση των κρατών μελών, ποιε απαντήσει δίνουν απέναντι σε κάτι τέτοιο. Και δεν αναφέρθηκα καν, καν για παράδειγμα στο Σούνερ Ζέμερ και ούτω Monsieur Kramer. Ευχαριστώ κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ μάλλον κύριε Κράμερ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στα υπόλοιπα μέλη που δεν είναι συντονιστέ. Δύο λεπτά όμω ο καθένα. Η κυρία Γιάλα Σέντερ πρώτα. Ε, να ευχαριστήσω του συντονιστέ για τι νέε πληροφορίε. Πρώτα απ' όλα τον κύριο Σίμψον ε, και εγώ όπως και ο κύριο Βαντενκάμπ ε, ήθελα σε σχέση με τα αποτελέσματα να πω αν μπορούμε να μιλάμε για νέους, ε, νέες ε, θαλάσσιες αρτηρίες, ε, αν υπάρχουν νέες συνδέσεις μεταξύ λιμανιών που θέλουν να ενισχύσουν την κυκλοφορία τους. Κύριε Βοητσεχόσκη, σε ό,τι αφορά το τούνελ του Ράτστατ, είναι ένα θέμα που εν των μελλοντικών διαδρόμων θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν είναι αναγκαίο, όπως είπε ο κ. Βαντενκάμπ, να αναφέρεται η συντήρηση, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, ποιες είναι οι ε, κατά την ε, κατασκευή και να γνωρίζουμε ποιο θα λάβει τη συντήρηση στο μέλλον. Κύριε Σέκη, ήθελα να αναφέρω όχι μόνο το θέμα ε, του διαδρόμου του Ατλαντικού ε, και το γεγονός ότι η Γαλλία δεν, δεν θεωρεί την προτεραιότητα πλέον στο τεφόρτιο συνοριακό κομμάτι. Ε, για τον κύριο Μπάλλα πάλι εκτό προτεραιοτήτων και η Μεσόγειος Πρέπει να βρούμε όμω μια φόρμουλα. Ε, εγώ στην έκθεσή μου, παραδείγματο χάρη για την λογιστική υποστήριξη, είπα ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εξάμεινο. Αν αυτό που ενοχλεί τους, υπουργούς, τους πρωθυπουργούς και τους πρόεδρους είναι το εξάμεινο, το ευρωπαϊκό εξάμεινο, τότε εκεί, εκεί να τους χτυπήσουμε. Αυτοί που δεν κάνουν τίποτα και επιπλέον ε, κοροϊδεύουν τα project αυτά όταν φτάνουν στο Παρίσι, διότι ο κ. Μακρόν ε, έχει σχέση με την απόφαση που πάρθηκε. δεν είναι κάτι καινούριο, το ήξερε. Ε, πρέπει λοιπόν να τους υποχρεώσουμε ή να πούμε ότι δεν έχουμε τελικά ευρωπαϊκά project, να το πούμε. Να το πει ο κ. Μακρόν στου Γάλλου και στου υπόλοιπου Ευρωπαίου. Διότι όταν είναι κάποιο Ευρωπα... Ευρωπαίο και Ευρωπαϊστή, σημαίνει ότι θα πρέπει να σέβεται ε, ε, τις υποχρεώσεις ε, και όχι επειδή υπέγραψε κάποιο άλλο να μην τις σέβεται ο οποίο ο άλλο ήταν ε, προεδρό του έτσι λοιπόν εδώ μα κοροϊδεύουν εγώ έχω βαρεθεί ε, και είναι και ο κ. Σέρτουγκ εδώ ο κ. Βαντενκάπ να μου λένε ότι οι φορτηγατζίδες οι Ισπανοί κάνουν κοινωνικό ντάμπινγκ στη Γαλλία αλλά δεν έχει ανοίξει ούτε ένας δρόμος από τη Γαλλία. Οπότε κοινωνικό ντάμπινγκ από την πλευρά μου και μάλιστα ε, έχω και λόγο. Ή θα ανοίξει ε, μια οδό ε, σιωδρομική η Γαλλία ή θα περνάμε με τα φορτηγά. Ε, τέλος, ε, κυρία Πρόεδρε, να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είμαι πολύ απογοητευμένη και ε, θυμωμένη. Γιατί ότι ο κ. Γκος και άλλοι είχαν άλλα πράγματα να κάνουν, αλλά στην περίληψη μου λέτε ότι το μόνο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και στον διάδρομο της Μεσογείου είναι τα 707 μέτρα. δεν είμαστε σοβαροί νομίζω έχουμε και τη συζήτηση στο μέλλον για τι δημοσιονομικέ προοπτικέ. Καλό θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει λίγο πιο σοβαρά ε, αυτά, αυτά τα ζητήματα και αυτέ τι εκθέσει. Εμεί το παίρνουμε σοβαρά. Παρακαλώ να το κάνετε κι εσεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γιάλα Σέντερ. Η κυρία Σαλίνη είχε το λόγο για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ. Δεν ε, μπόρεσα να συμμετάσχω στο πρώτο τμήμα της συζήτησης γιατί πρέπει να ασχοληθώ με τις ενέργειες μεταφορές. Θα ήθελα να επισέλθω σε μεγαλύτερο βάθος ό,τι αφορά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και τους τρόπους με τους οποίους ε, σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα διατροπικότητας, διαλειτουργικότητας και το ERTMS. Συνήθως εξετάζουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση για το ERTMS. Σε αυτήν την περίπτωση όμως νομίζω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε και εναλλακτικέ μορφές χρηματοδότησης όπως το σχέδιο Juncker, το EFSI. Δεν μπορούσαν να είναι σημαντικά αυτά τα εργαλεία. Πριν από τρία χρόνια παρουσίασα ένα πιλωτικό σχέδιο από αυτή την άποψη για τη χρηματοδότηση ενός από τα πιο στρατηγικά ε, κέντρα σιδηροδρομικών μεταφορών για το μέλλον, κατά τη γνώμη μου. Το ερώτημα λοιπόν είναι για το ERTMS. Ξέρω ότι ξεφεύγω λίγο από ε, το θέμα συζήτηση αυτή τη στιγμή, αλλά δεν συμμετείχα στην πρώτη συζήτηση. Κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την γενεδορία και συγγνώμη, αλλά θα ήθελα να ήμουν εδώ νωρίτερα, αλλά καθυστέρησε μια άλλη συγκίτρια στην Επιτροπή Αλίας ε, και εγώ ήμουν υπεύθυνη εκεί και δεν μπόρεσα να έρθω νωρίτερα. Ε, ακούω εδώ με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που έχουν υποθεί. Θα είμαι όμω σύντομη και θα απευθυνθώ στον κύριο Σέκη. Εγώ νομίζω ότι εν μέρη η συνάδελφος η Νέσα Γιάλα τα είπε τα βασικά. Ε, ο τίτλος λέει εδώ «Προώθηση για χρηματοδότηση καινοτόμο, για καινοτόμο χρηματοδότηση». Υπάρχει τίποτα πιο καινοτόμο το να σεβόμαστε ε, τις ε, δεσμεύσει μας για τις προτεραιότητες. Είχαμε πει το 2013 ποια είναι τα project προτεραιότητας για την Ευρώπη. Ορίσαμε ποια είναι τα λιμάνια, ποια είναι τα αεροδρόμια που θα πρέπει να συνδεθούν για να υπάρχει αυτή η διαλειτουργικότητα. Και να πετύχουμε και αυτό που έχουμε πει εδώ και καιρό, ότι χρειαζόμαστε και ένα χάρτη ευρωπαϊκό διότι μας έλεγε η Κομισιόν μας σχεδίασε τις προτεραιότητες μας έλεγε ότι πρέπει το 1% του ΑΕΠ του ευρωπαϊκού το χάνουμε αυτή τη στιγμή ε, στα σύνορα, στα, σημεία διέλευση των σύνορων, με τις, ε, τα μποτιγιαρίσματα, στη χώρα των Βάσκων παραδείγματος χάρη, στα σύνορα μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας. Εγώ φοβάμαι να οδηγήσω σε εκείνον τον αυτοκινητόδρομο. Δεν είναι μόνο όλο το δεξίδιο του άνθρακα εκεί, που δεν υπάρχει καμιά άλλη, καμιά άλλο μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει καμία λειτουργικότητα. Υπάρχουν, μπαίνουν και ζητήματα ασφαλεία όμω, όπω ένα και μετά. Το 2013 υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Για άλλη μια φορά ήταν προτεραιότητα αυτό το θέμα είπαμε ότι πρέπει να προωθήσουμε πρόσφυγες τα οποία έχουν η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεταφορών ε, το γνωρίζει αυτό ότι θα χρηματοδοτήσουμε μόνο ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων project Γιατί δεν πετύχαμε τίποτα. Το πιο καινοτόμο λοιπόν θα ήταν να σεβαστούμε τι δεσμεύσει μα, Διότι σε κάποιε περιοχέ έχουν επενδύσει άνθρωποι σε αυτά τα project αλλά δεν πάνε πουθενά αυτέ οι επενδύσει. Είναι καινοτόμο αυτό. Αυτοί που προσπαθούν να σεβαστούν τι δεσμεύσει είναι αυτοί που χάνουν χρήματα αυτή τη στιγμή. Διότι αυτέ οι επενδύσει που δεν χρησιμοποιούνται, που δεν προχωρούν, οδηγούν σε πιστογυρίσματα. Τώρα, εάν θέλουμε να συμμετάσχει ο ιδιωτικό τομέα στον τομέα των μεταφορών, θα πρέπει να του δώσουμε νομική ασφάλεια, να του, δώσουμε, να του παράσχουμε εμπιστοσύνη. Αν τα κράτη-μέλη όμω δεν λογοδοτούν, δεν ανταποκρίνονται στι δεσμεύσει του, τότε δεν υπάρχει καμία ασφάλεια και δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν καινοτόμο χρηματοδότηση εφόσον δεν δεσμευθούν οι ε, εμπλεκόμενοι υπουργοί και τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη. Στον ε, ε, Ατλαντικό η Γαλλία έχει μια στάση η οποία είναι απαράδεκτη όχι τώρα και χθε. Και ελπίζω να μην συμβαίνει αυτό και αύριο. Και η Ισπανία που στο παρελθόν ε, ούτε αυτή τη συμφωνία τη τώρα, τώρα τη σέβεται. Χρησιμοποιήστε λοιπόν αυτή την πίεση ε, από όλου, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τι δεσμεύσει του. Δεν μπορούμε να αναθεωρούμε τα project τα οποία έχουμε ορίσει από το 2000, από το 1994 στο, στο Συμβούλιο του ΕΣΕΝ και άλλη μια φορά να ξαναβλέπουμε το 2018 και το 2019. Πραγματικά είναι κοροϊδία. Είναι κοροϊδία και κακοδιαχείριση. Κακοδιαχείριση των χρημάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτό το θέμα πρέπει να το λύσουμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Αλλά πρέπει κανεί να δείξει πολιτική βούληση για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μπριμπάου. Είχα και εγώ ορισμένε ερωτήσει. Πολύ σύντομα θα τι θέσω. Πρώτον, όλοι οι συντονιστέ συμφωνούν ότι χρειάζονται περισσότερες επιχορηγήσεις για το περιβάλλον στο μέλλον. Από την δική μας Επιτροπή όλοι συμφωνούμε. Γιατί πρόκειται για μοχλούς που θα εξασφαλίσουν την επιβίωση των περιφερειών σε όλη την Ευρώπη. Όμως, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το θέμα του blending. Πράγματι, εντάξει, να περάσουμε και στο blending. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να ε, παλέψουμε για τις επιχορηγήσεις που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το blending. Γι' αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε για να έχουμε τους απαραίτητους πόρους και μετά βλέπουμε πώς θα τα συνδυάσουμε. Το δεύτερο ζήτημα, πολύ σωστά το είπε ο κύριος Σελήνη, είναι σκανδαλώδες ε, ότι από το ΕΦΣΥ βλέπουμε ότι κάτω από το 10% των έργων ε, αφορά τις μεταφορές. Είναι προβληματικό αυτό έχει έρθει ο καιρός, θεωρώ ότι πρέπει και εμείς να σταθούμε αυτοκριτικά. Παρότι ε, ο μηχανισμός ε, των interconnectors έχει αποτελέσει και μία αγορά. Υπάρχει και πρόοδος και προβλήματα όμως, κριτική πρέπει να γίνει. Και στα έργα των υποδομών ε, δεν τα πηγαίνουμε καλά και για τον αντίκτυπο στον περιβάλλον και στη διαφάνεια στο οικονομικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε προδραστικά και σε αυτόν τον τομέα. Εσείς συμμερίζεστε αυτή τη στάση. Δεύτερον, ξέρετε ότι δεν είμαι υπέρμαχος ε, ε, της σύνδεσης αυτής της σύνδεσης Λιών-Τωρίνου, όμως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί κύριε Παβέλη είπατε καθυστερήσαμε τις εργασίες, γιατί υπήρξαν ε, αντιδράσεις των κατοίκων που τους ενοχλούσε ο θόρυβος. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να στηρίξουμε έργα που αντιβαίνουν στις προσδοκίες των κατοίκων. Να, να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν προς αυτό. Πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά από απόψη σαφώ. Δεύτερον, συμφωνώ απολύτω με του συναδέλφου ότι σήμερα έχουμε ε, έργα που είναι, έχουν λάβει προβολικέ διαστάσει και αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε εναλλακτικέ. για κάποιες περιπτώσεις ε, πρέπει να υπάρξει ανακαίνιση. Υπάρχει όμως εναλλακτική. Στο Λιόν, το Ρήνο, ε, υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα θα υπάρξουν στο μέλλον. Τι θα κάνουμε στα 20 χρόνια. Τι θα κάνουμε συγκεκριμένα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει ε, να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία χωρίς να περιμένουμε μέχρι το 2038 ιδίως επειδή σε αυτή την κοιλάδα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα ρήπανσης που τα βλέπουμε καθημερινά ε, στα πρωτοσέλιδα. Τώρα, για τα ποτάμια και τα θαλάσσια λιμάνια, συμφωνώ με τον κύριο Σίμψον ότι πρόκειται για πραγματικό διακύβευμα. Γιατί οι ωκεανοί και οι θάλασσες είναι το μέλλον. Συχνά τα αμελούμε. Αλλά Πώ θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ένα σωστό μέλλον για αυτού τους ε, κλάδους. Ε, καλησπέρα κύριε Μαρινέσκου, αργήσατε βέβαια λίγο. Θα σας δώσω χρόνο τώρα να απαντήσετε. Ο κύριος Σέκη, γιατί πρέπει να πάρει και το τρένο μετά, παρακαλώ. Uh, thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ορισμένες παρατηρήσεις, εν συντομία. Πρώτα απ' όλα, Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στη Γαλλία σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις ε, της γαλλικής κυβέρνησης που βέβαια δεν τις έχει υιοθετήσει ακόμα, δεν έχει κλείσει τίποτα, δεν θέλουμε κι εμείς να παρέμβουμε, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθούν οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις. και για την υποστήριξη της ενιαίας αγοράς και για τον κανονισμό TNT. Θεωρούμε και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα τηρηθούν ε, μέχρι κεραίας. Αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε να μην ισχύσει αυτός ο όρος που αναφέρατε, η υπονόμευση, η υποβάθμιση της προτεραιότητας. Θα το προσέξουμε λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε και θα ήταν και ενδιαφέρον να γίνει μια ανταλλαγή αποφασίων και στο μέλλον για αυτό το θέμα στο νότο χώρο, το Βάσουν και Τα, τα πράγματα ναι, βαίνουν καλώς, ε, παρότι υπάρχουν προβλήματα. Με τον νέο κανονισμό ΣΕΦ και ο ορισμός των έργων στο διάδρομο είναι κάτι το οποίο αναλαμβάνει Move και έτσι υπάρχει βελτίωση για αυτή την άποψη. Εκτιμούμε λοιπόν όλες ε, τις εξελίξεις ε, στη Γαλλία και παρακολουθούμε τι συμβαίνει και από την άλλη πλευρά. Σίγουρα όλα αυτά θα πάρουν χρόνο, αλλά εμείς είμαστε υπέρ των μεταβατικών μέτρων που μας οδηγούν σε καλύτερα προγράμματα, καλύτερα αποτελέσματα. και νομίζω ότι και εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις. Τα ομόλογα των έργων και καινοτόμους χρηματοδότηση, τα ομόλογα αυτά ήταν ε, πρόγονοι και πρόδρομοι των, ε, του σχεδίου Juncker. Κάποια από αυτά λοιπόν χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή και το αναφέρουμε ε, αναλυτικά και στην έκθεσή μας. Είμαστε λοιπόν στη διάθεσή σας, αν θέλετε περαιτέρω διευκρινήσεις. Υπήρχαν καθυστερήσεις ε, σε όλα τα αεροπλάνα από την Ιταλία. Τώρα ελπίζω να είναι στην ώρα του. Ευχαριστούμε πολύ που απαντήσατε κύριε Σέκη. Θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας, εάν υπάρχουν ακόμα ερωτήσεις και είστε πάντα ευπρόσδεκτο στην Επιτροπή μα. Συνεχίζουμε με τον κύριο Μποντεβίκ. Ισμαήλ, <laughs> ε, ε, <clears throat> και εγώ να πω ότι πράγματα ε, με χαρά μου συμμετέχω κάθε φορά στι εργασίε του Κοινοβουλίου, γιατί κατά τη δική μου άποψη αποτελούν οι ευρωβουλευτέ υπέρμαχου ενό ε, κατάλληλου προπολογισμού για το ΣΕΦ και χρειαζόμαστε αυτή την υποστήριξη από, τα, από τους ευρωβουλευτές γιατί εκείνοι που θα πρέπει να πείσουμε είναι τα κράτη-μέλη. Ε, και αυτό με φέρνει στο επόμενο ζήτημα, το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, δεν θα είναι αποφασιστική σημασία ω προ την περαιτέρω εξέλιξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα είναι και αποφασιστικό και για το δικό μα τομέα αρμοδιότητα. Δηλαδή, κατά πόσο τα όσα έχουμε κάνει κατά τα τελευταία 7 ή 4 χρόνια στην δική μου περίπτωση ε, είχαν τελικά νόημα ή όχι. Αν θα λάβουν δηλαδή συνέχεια ή όχι. Και το ερώτημα που εμεί θέτουμε ξανά και ξανά είναι η Ευρωπαϊκή ε, προστιθέμενη αξία. Δηλαδή όταν δημιουργώ κάτι, όταν κάνω μεγάλα έργα αλλά δεν καταφέρνω να ολοκληρώνω το σχετικό δίκτυο τότε αυτό που κάνω είναι λανθασμένο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ο ε, συνάδελφος Κάλλο αναφέρθηκε σε αυτό, βέβαια χρειάστηκε να φύγει τώρα, αλλά ήδη στη δική μα έκθεση αναφέρουμε μία σειρά από προτάσεις στο τι μπορούμε να κάνουμε συμπληρωματικά έτσι ακριβώ να διασφαλιστεί αυτή η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε σχέση με αυτά τα προγράμματα. Και αυτό είναι η δική μα τοποθέτηση στην κοινή δήλωση από την πλευρά όλων των συντονιστών ότι πράγματι χρειαζόμαστε αυτή την ευρωπαϊκή προστέμενη αξία. Πρόκειται δηλαδή για μια επιτυχία την οποία έχουμε σημειώσει, κατά τη συνέπεια σε καμία περίπτωση θα έπρεπε να διακοπεί αν θέλετε αυτή η επιτυχία. Θα ήταν τρελό κάτι τέτοιο. Ενώ πολύ συχνά ένα μεγάλο τμήμα των δαπανών ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνονται ε, προ ε, έργα τα οποία ακριβώ δεν έχουν αυτή την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, αυτή την ευρωπαϊκή διάσταση. Από εκεί και μετά. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι αυτό τη. Ε, περισσότερης ε, ε, της μεταστροφής στην ηλεκτρική ενέργεια. Αναφερθήκαμε σε αυτό το ζήτημα στις, στις αδειοδοτήσεις και όπως ανέφερε ο Μάρκος ότι ήδη σε ένα βαθμό έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Άρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να οργανώσουμε λίγο τα σχέδια εργασιών και να διασφαλίσουμε τις ανάληψη δεσμεύσεων από τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να, να, να, τα πιέσουμε να κάνουν κάτι άλλο. Ε, τώρα σε ό,τι αφορά τις οδούς σύνδεσης, για παράδειγμα, το καταφέραμε αυτό στο παρελθόν. Βγαίνει η Μπρατισλάβα για παράδειγμα. Ε, σίγουρα θέλουμε σε κάθε περίπτωση ε, και το Ζέβερν και άλλες, ε, άλλα μεγάλα έργα, τούνελ κτλ. να στεφτούν με επιτυχία, αλλά και πάλι εδώ εξαρτάται βέβαια από την τρόπο υλοποίηση του κάθε επιμέλου έργο του, αν τελικά επιτυχάνονται αυτέ οι περαιτέρω συνδέσει. Και εδώ έρχομαι και πάλι στο ζήτημα που τέθηκε σε ό,τι αφορά την απλουστευμένη διαδικασία διοδότηση, χωρί δηλαδή να υποβαθμίζουμε την ποιότητα. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενίσχυση, απλώ να κάνω μια διευκρίνηση ώστε να μην ε, να κατανοήσετε με, με λανθασμένο τρόπο. Δεν είπα να κατευθούμε εντελώ τώρα στην περιφερειακή εντοδιάσταση, αλλά λέω πως έχει νόημα η ενοποίηση σε περιφερειακό επίπεδο κονδυλίων. Γιατί δηλαδή να παίρνω κονδύλια τα οποία ε, ε, κατευθύνονται στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασία, γιατί να μην πάρουμε κονδύλια από αυτά και να μην τα ενοποιήσουμε με τα έργα που κάνουμε εδώ, με τι επενδύσει στι υποδομέ. Γιατί βέβαια, εάν δεν έχουμε την την αποσπασματική προσέγγιση δεν θα λειτουργήσουν καλά τα πράγματα. Αν ενοποιήσουμε τις προσπάθειες θα έχουμε αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν το διευκρινίζω για να μην γίνω με λαθασμένο τρόπο κατανοητός. Ε, αυτό δηλαδή που θέλω να πω ότι σίγουρα θέλουμε επικοδομητική συνεργασία. Τέλος, σε ό,τι αφορά το συντονισμό, ε, το blending calls ε, πήγαν καλά. Θα μπορούσαμε βέβαια να δούμε τι θα μπορούσε να βελτιωθεί, πώς μπορεί να καταστεί ακόμα πιο αποτελεσματική αυτή η συνεργασία και από εκεί και μετά βέβαια όλοι όσοι είμαστε υπέρ αυτών των ε, έργων αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να ταχθούμε υπέρ της αύξησης των κοντιλιών του ε, ΣΕΒ. Δεν μπορούμε απλώς και μόνο να ε, βελτιώσουμε τις διαδικασίες. Από κοινού θα έχουμε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Δηλαδή και αύξηση των κοντιλιών και καλύτερες διαδικασίες. Και μετά κάτι τελευταίο. Όλοι ναι θα πρέπει να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ευχαριστώ. Intervention. Ευχαριστώ για την παρέμβαση σας. Ο κύριος Σίμψον έχει το λόγο, παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν για αυτό που είπατε προηγουμένως για μένα. Θα το βάλω μαζί με τα υπόλοιπα παράσημά μου. Πρέπει να ξέρετε ότι οι εξελίξεις στον τομέα των θαλάσσιων ουσιαστικά συνδέονται με τις εξελίξεις στην ψηφιακή εποχή. Γνωρίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό στο θαλάσσιο τομέα σε ό,τι αφορά την ενιαία θηρίδα τώρα τέτοιο σχετικό ερώτημα κατά πόσο είναι μειονέκτημα εγώ θέλω να υπάρχει τέτοια θηρίδα. Έχει νόημα. Πρέπει να το διευρύνουμε και να υπάρχει μόνο ένα στο τέλος. Δεν έχει νόημα να μου το λέτε εμένα αυτό όμως. Πηγαίνετε να δείτε τα κράτη-μέλη, διότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία δεν δίνουν όθηση σε αυτό το project και που είναι ικανοποιημένοι να βλέπουν ένα φορτικό από την Πορτογαλία ως τη Δανία ε, να έχει ένα ε, πακέτο εγγράφων και να περνάει από ε, για ένα, ένα πακέτο γράφων να έχει 7-8 διαφορετικά έγγραφα. Εγώ είμαι υπέρ λοιπόν τη ενιαία θηρίδα. Τώρα μεταξύ Ισπανία και Ιταλία υπάρχει μια κάποια συνεργασία για την επίλυση του ζητήματο. Εμεί ε, συμμετέχουμε σε αυτό ενεργά. Τώρα η Σικελία. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε χρήματα σε ένα λιμάνι το οποίο δεν αποτελεί μέρος του πυρήνα ή μπορεί να είναι ένα συμπεριληπτικό λιμάνι αλλά πρέπει να συνδέεται και με ένα άλλο κράτος μέλος αυτός είναι, αυτός είναι ο κανόνας, αυτοί είναι οι κανόνες πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη Βεβαίω θα μου πείτε αυτά είναι βλακίες αλλά τι να σας πω, αυτοί είναι οι κανόνες προσπαθούμε στις εργασίες μας να το αλλάξουμε αυτό. Να δούμε αν υπάρχει περιθώριο να συνεργαστούμε και με αυτά τα λιμάνια. Γιατί είναι και άλλα πολλά λιμάνια στη Φιλανδία, στη Σουηδία, κάποια στην Ισπανία, όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Να τους βοηθήσουμε δηλαδή. Και για την Ινές κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον στην διασύνδεση των Μαξιτών λιμανιών. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, βεβαίω. Μα πήρε τέσσερα χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ενδιαφέρον. Τα λιμάνια μιλούν ε, για διασύνδεση. Δηλαδή δεν λένε πια να δω πρώτα τι θα κάνει ο άλλο πριν κάνω εγώ το οτιδήποτε. Ε, αυτή είναι η φύση του κλάδου αυτού. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι τα λιμάνια είναι ιδιώτε ιδιώτες κυρίως και είναι πολύ επιφυλακτικοί μεν απέναντι στους δε. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά υπάρχει σίγουρα ενδιαφέρον. Μάικλ, αυτό το bonky feel είναι πολύ προβληματικό. Και εγώ θα ήθελα να υπάρχει μία ε, άλλη εναλλακτική πέρα από αυτά τα καύσιμα. και τα καύσιμα. Αυτό το στο καύσιμο, το bunker fuel, είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Κάτι περισσότερο. Τα καύσιμα κίνησης. Επίσης, εδώ έχουμε πάλι το κανόνα με τα δύο κράτη-μέλη. Πρέπει να υπάρχει διασύνδεση με τα δύο κρατών μελών για, αυτό που είπατε προηγουμένω για τι ε, υποδομέ υποδοχή των λιμανιών. Προηγουμένως, κυρία Μπιλμπαϊρ, εγώ συμφωνώ με αυτά που είπατε, αλλά δεν λέτε σωστό, δεν απευθύνει στους ανθρώπους. Πρέπει να το πείτε στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά που κάθε τέσσερα χρόνια αλλάζουν γνώμη και πάνε προς άλλο project. Και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό για μας ως συντονιστές να, να χαράξουμε μια μακροπρόθεσμη πολιτική ενώ τα κράτη-μέλη αλλάζουν κυβερνήσεις ε, κάθε λίγο και λιγάκι. Τέλος, Πρόεδρε, ε, είστε πραγματικά η ηρωίδα της εβδομάδας, του, του χρόνου. Λέτε την πραγματική πρόκληση είναι ότι το, το μέλλον είναι η θάλασσα. Επι, επιτέλους, αλληλούια, κάποιος το είπε και αυτό. Ε, δεν θέλει και πολύ για να είναι κάποιος ευχαριστημένος από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Η κυρία Πέιζ έχει το λόγο τώρα για να απαντήσει και αυτή σε κάποια ερωτήματα. Ik begin, ik begin, eh, I start with, eh, eh, with Wim van ehm, Θα αρχίσω με τον κύριο Βαντεν Κάμπ. Βιμ, οι μεταφορές ως υπηρεσία. Αυτή είναι η αρχή και η αφετηρία. Στις 6 Μαρτίου υπάρχει ένα μεγάλο συνέδριο ε, για αυτό το ζήτημα, αν σας ενδιαφέρει. Το μόνο σίγουρο λοιπόν είναι ότι μπορεί να υπάρξει έτσι η προσπάθεια του Υπουργείου και μπορεί κανείς να ακολουθήσει κάθε ε, μεταφορικό μέσο που θέλει. Όμως και τα εμπορεύματα τώρα θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτή την οδό. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Θα ίσως να μάθω στο συνέδριο και θα σας ενημερώσω. Η συντήρηση δεν είναι στο TNT και ούτε πρέπει να είναι. Το μοναδικό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αν οι υποδομές γίνονται με τα κράτη-μέλη ιδίω κράτη-μέλη που δεν ε, έχουν μεγάλο περιθώριο χρηματοδότησης, ε, είναι και δική μας ευθύνη να εξετάσουμε κατά πόσο έχουν τα χρήματα για τη συντήρηση. Ιδάλλως ε, είναι μεγάλο το ρίσκο. Αν κάνουμε μια καινούρια αρτηρία ή σιδηροδρομική γραμμή, το σημαντικό είναι να υπάρχει μία μακρόπνοη γραμμή προπολογισμού για πολλά χρόνια για τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Αυτό είναι σημαντικό. Βέβαια είναι ε, πολύ πιο ελκυστικό το να φτιάχνει κανείς νέους δρόμους και νέες σιδηροδρομικές γραμμές παρά να τη συντηρεί. Αλλά είναι σημαντικό για την ασφάλεια. Τώρα για τον Δούναβη που είπατε, δεν συμφωνώ ότι είναι επένδυση, είναι ε, συντήρηση. Όμως σε όλους τους κανονισμούς και σε ΕΦ και σε άλλους ε, η συντήρηση αυτή μπορεί να γίνει ε, με ένα dredger. Αυτό κάναμε λοιπόν και σήμερα το πρωί μάθαμε ότι έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, είναι εκεί το σκάφος και θα ξεκινήσει η βυθοκόρηση στην κοινή ζώνη Βουλγαρίας-Ρωμανίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γίνει αυτό και να ξεκινήσει αυτή η εξκαφή. Δεν είναι λοιπόν η ίδια εξκαφή, είναι ο εξοπλισμός που χρειαζόμαστε. Και οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν με χρήματα του ΣΕΦ. Τώρα, γειτονικέ χώρε ή τρίτε χώρε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σκέλο γιατί αν έχουμε έναν διάδρομο, πάρουμε το παράδειγμα τη Σερβία. Γιατί είναι ακριβώ στη μέση. Η Σερβία λοιπόν έχει αυτή την σιδερά πύλη που για 40 χρόνια διατηρούσαν αυτό το εμπόδιο, αλλά σίγουρα τώρα χρειάζεται ανακαίνιση. Εάν δεν υπάρχουν τα χρήματα όμως δεν μπορεί να γίνει αυτό και έτσι δεν λειτουργεί ο διάδρομος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να το συμπεριλάβουμε αυτό στο επερχόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Να δούμε τι είδους βοήθεια μπορούμε να, δούμε, να δώσουμε σε τέτοια συνοριακά έργα. <laughs> Oh. <laughs> so, um, Κυρία Μάισνερ. Α, δεν έχω άλλο χρόνο. Okay, Εντάξει. Αν υπάρχει διατροπικότητα, υπάρχει. Θέλουμε εμείς να συνδέεται το λιμάνι με το σιδηροδρομικό δίκτυο οπωσδήποτε με το δικό δίκτυο, αλλά όπου αυτό είναι δυνατόν και με, το σιδηροδρομικό δίκτυο. Σε πολλές περιπτώσεις το καταφέρνουμε. Heavy oil. I tell you about heavy oil. Θα σας πω εγώ για, τα, για το πετρελοκίνηση στη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπαλάς δεν, δεν είναι εδώ. Παβέλ. Μου επιτρέπετε να σας ε, απευθύνω το λόγο με το μικρό σας όνομα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Πρώτον, το ζήτημα για το ποιο μπλοκάρει ποιον. Έχουμε ε, αρνητικές επιπτώσεις ε, στην τοπική κοινότητα. Είναι ένα κλασικό πρόβλημα που έχουμε. Κύριε Βαντερκάμπ, είπατε ότι οι πράσινοι εμποδίζουν τη διαδικασία της ε, ζώνη Φέρμεντ. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με τι νομικέ διαδικασίε. Κάποιες χώρες έχουν, ε, ε, δίνουν μεγαλύτερο ρόλο και μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης στις τοπικές κοινότητε. Μπορεί αυτό να γίνει και στη Βουλγαρία με τις πρωτοβουλίες πολιτών και με αρνητικές εξωτερικές επιπτώσει και σε άλλα έργα. Αυτό πρέπει κάπως ε, να συγκεράζεται με τη σωστή προσέγγιση και οι λύσει να προκύπτουν από τα πάνω προς τα κάτω. Γιατί χωρίς αυτά τα μέσα, το μετριασμό για παράδειγμα του θορύβου ε, στο σιδηρόδρομο, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τους διαδρόμους. Ε, τα επίπεδα θορύβου στο σιδηρόδρομο ήταν ένα κλασικό πρόβλημα. Ποιο να το χρηματοδοτήσει όμω η Deutsche Bahn ή ε, ίσως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να στη χρηματοδοτήσει μέσω του ΣΕΦ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση μέσω του ΣΕΦ. Γιατί δεν, ε, είναι δεν ευθύνεται η Deutsche Bahn για το γεγονός ότι ο κόσμος θέλει να μένει κοντά ε, στο σιδηρόδρομο και έτσι πέφτουν οι τιμές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της συνεργασίας μας ε, με ε, τον διάδρομο αυτό για την ε, αναδρομική μείωση των αρνητικών επιπτώσεων για να μετριάσουμε ακριβώς αυτό το ρήπο και τα επίπεδα θορύβου. Μετά. Πώς Μπορούμε να προλάβουμε τις ε, διόδους πρόσβασης. Για παράδειγμα, στο τούνελ Γκόταρτ. Οι Ελβετοί την περσμένη εβδομάδα ήταν εδώ και μας είπαν ότι θα ολοκληρωθεί αυτό μέχρι το 2020. Ίσως άλλοι όμως να ολοκληρώσουν αυτή την ε, προσπάθεια σε 20 χρόνια. Όμως, ε, η, σύνδεση μεταξύ των Άλπαιων ε, ωφελεί τη διέλευση. Το 80% θα αφορά λοιπόν διέλευση εμπορευμάτων μεταξύ των δύο πλευρών των Άλπαιων. Ποιος λοιπόν ε, ωφελείται και πάλι οι χώρες που θέλουν να συνεχίσουν αυτή τη διαμετακόμιση μάλλον. Τέλος για τη διατροπικότητα που έδειξε η κυρία Μάισνερ, βεβαίως ε, και εννοούσα την πολυτροπικότητα με την ε, γενική έννοια και για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Όμως ε, δεν ισχύει καθολικά. Στο Ρήνο έχουμε πολλές τριτροπικές πλατφόρμες που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικέ. Στην εσωτερική ναυσιπλοεία, στο Ρήνο βλέπετε ότι είναι το 20% της ικανότητα. Όταν είχαμε το συμβάν στο Ράνστατ, κάποια από την κίνηση πήγε ε, σε άλλους λιμένες. Οι περισσότεροι βέβαια στράφηκαν προς το δικό δίκτυο. Και έτσι υπήρχε μια αντίστροφη μεταστροφή προς το δικό δίκτυο. Κύριε Κράμερ, μίλησατε για τη συντήρηση. Όπως είπε και η Κάρλα, νομίζω ότι αυτό δεν εντάσσεται στο ΣΕΦ. Πρέπει όμως και εμείς να αποστέλουμε συνεχώς αυτό το μήνυμα προς τους αρμόδιους, να εξετάζουν το συνολικό κόστος που είναι ο πλήρης κύκλος ζωής του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης. Τέλος. Κάποιε από τι άλλε παρατηρήσει που αφορούν τον άξονα Σκανδιναβία τη Μεσογείου, καλό είναι να αποσταλούν γραπτό στον αρμόδιο για να απαντήσει. Ευχαριστούμε πολύ για όλε τι απαντήσει. Πραγματικά μπορούμε να συγχαρούμε του συντονιστέ μα. Περάσαμε πολύ ωραία. Αλλά είναι σημαντικό γιατί πάντα μας ακούτε και πάντα όταν σας καλούμε έρχεστε με μεγάλη χαρά στην Επιτροπή μας. Και αυτό πραγματικά είναι μια, μια συνεργασία σημαντική και θετική. Συγχαρητήρια, λοιπόν. Euh, Για την επόμενη φορά ε, θα βοηθήσουμε το ΣΕΦ να λάβει το του διάσταση. Δεν έχουμε, ολοκληρωθεί, δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει την συνεδρίαση. Όλοι αναφερθήκατε ε, στα προσκόμματα που θέτουν τα ίδια τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το φαινόμενο το οποίο οδηγεί σε καθυστερήσεις ε, γιατί υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Ορισμένα κράτη-μέλη παρεμποδίζουν και παρακολουθούν τη διαδικασία. Ελπίζουμε στο μέλλον να καταφέρουμε να προσδώσουμε αυτή την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που θα μας δώσει πραγματική διασυνδεσιμότητα που όλοι χρειαζόμαστε. Και το λέω έτσι τόσο έντονα, γιατί πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά έργα δεν μπορούν να ελοπιθούν χωρίς ε, σωστές μεταφορές και διασυνδέσεις που θα μας επιτρέψουν να ανταλλάσσουμε εμπειρίες, εμπορεύματα. σα ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. και οι συνάδελφοι θα σας στείλουν ε, ενδεχομένως και γραπτός ε, ερωτήσεις, αν θέλουν προσθέρες λεπτομέρειες. Ε, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα τον Απρίλιο στη Λουβλιάνα. Ευχαριστώ λοιπόν. Τα λέμε σύντομα. Κύριε Βαντερκάμπ, έχετε ερώτηση? Α, τόσο το καλύτερο. Τα λέμε αύριο στις 9 το πρωί. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς.